Αξιότιμοι συνάδελφοι, δυστυχώς πριν δύο ώρες μάθαμε ότι ο Πάβελ Αντάμοβιτς, ο δήμαρχος της δεν, του Ντάνσκ, δεν επιβίωσε από τη χθεσινή επίθεση. Όσοι τον γνωρίζουν θα ξέρουν πόσο αφαισιωμένος ήταν στην υπηρεσία των πολιτών, το ανοιχτό του πνεύμα και την ικανότητά του για να ακούει τους ανθρώπους. Θα ήθελα να εκφράσω εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα συλληπιτηριά μας ε, στους συγγενείς τους και σε ολόκληρη την πόλη του Τάνσκα. Πριν ένα μήνα η ε, δειλή επίθεση που χτύπησε την καρδιά του Στρασβούργου σκότωσε τη ζωή στο Σκαλβερτέν, ε, στον Καμάλα Σαμπάντ, στο Νοπόγκ Σοπιστάν, στον Αντώνιο Μεγκαλίτσι και στον Μπάρτ Πρέντο ε, Όριεν Νετζέλσκι. Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά θρηνούμε θύματα του μίσους, του εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικοποίησης στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γεννήθηκε καταρχήν για να εγγυθεί την ειρήνη και για να καταπολεμήσει κάθε μορφή βίας. Και όμως ε, λίγους μήνες πριν από τις εκλογές του ΜΕΙΟΥ βλέπουμε να αυξάνεται η ένταση σε διάφορα κράτη-μέλη. Τις τελευταίες εβδομάδες είδαμε επιθέσεις σε πολιτικούς στην Ουγγαρία, στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο και είχαμε διάφορα επεισόδια αντισημιτισμού ακόμη ε, και σε κάποιες, ε, κάποιους αγώνες ποδοσφαίρου και θα ήθελα να πω ότι η ευθύνη ανήκει σε όλους ε, και θα πρέπει η συζήτηση να γίνεται με το σεβασμό του αντιπάλου που δεν θα πρέπει να μετατρέπεται σε εχθρό. Πολλές φορές έχουμε βιώσει και φεραστική βία και μπορούμε να δούμε πώς μπορεί να καταλήξει σε σωματική βία. Πρέπει να έχουμε διαφορετική γλώσσα και να εξαλείφουμε κάθε δήλωση μίσος που δεν συνάδει με την ειρηνική συμβίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν απευθύνω έκκληση όλοι να χαμηλώσουν τους τόνους και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η επίθεση του Στρασβούργου μας δείχνει ότι δεν μπορούμε να εφησυχαζόμαστε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει αμελητή να μάχεται κατά της τρομοκρατίας κάθε τύπου. Και δεν θα ξεχάσουμε κανένα από τα θύματα. Αυτή την εβδομάδα, όπως ζητήσατε, θα συζητήσω με το Δήμαρχο του Στρασβούργου για να δούμε πώς μπορούμε να ποτίσουμε φόρο τιμή στα θύματα του Δεκεμβρίου και ήδη απόψε θα προτείνω στο Προεδρείο ε, να ε, κατονομάσουμε τον Αντώνη Μεγκαλίτση και τον Πάρτο Σπέτρο Όρεν σε σε ραδιοφωνική εκπομπή. Είναι δύο δημοσιογράφοι που δολοφονήθηκαν και θα ήθελα να τηρήσουμε ένα λεπτό σιωπή στη μνήμη όλων των θυμάτων της βίας και του μίσους. Επανάληψη τη Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που είχε διακοπεί στι 23 Δεκεμβρίου 2018. Παρακαλώ, κύριος και έχει το λόγο. Ευχαριστώ, πρόεδρα για το μήνυμα που στείλατε στο Twitter και πλέον που δεν υπάρχει πλέον ελπίδα. Πρέπει να πούμε ότι αυτά που συνέβησαν στον Τάνσκ αποτελούν μια προσωπική τραγωδία για έναν πολύ δημοφιλή και νέο νεοεκλεκτήσα, πρόεδρο στο Ντάνσκ, δήμαρχο στο Ντάνσκ. Καλός φίλος λοιπόν ε, και καλός φίλος των ευρωπαϊκών αξιών. Μεγάλο δράμα για την οικογένειά του και μεγάλο σοκ για την κοινότητα του Γκτάνσκ. Που χθε ε, μαζεύτηκε για μια αρκετά ευχάριστη ευκαιρία, για έναν φιλανθρωπικό, για μια φιλανθρωπική εκδήλωση. Αλλά εδώ μιλάμε και για την μνήμη της τρομοκρατικής επίθεσης στο Στρασβούργο, μια μνήμη φρέσκια. Είναι υπερβολικά συχνές λοιπόν στην σημερινή Ευρώπη οι εκδηλώσεις βίας που αντικαθιστούν το διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη πέρα από τις διαφορές μας. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει τροφή για σκέψη. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, συνάδελφος Ροντρίγκης. Uh, Όντω, εξ ονόματο του Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και επειδή τον ήξερα και προσωπικά, θα πρέπει να σα πω και δύο λόγια για το τι σημαίνει αυτός ο φρικτός ε, φόνος του ε, Δημάρχου του Γκτάνσκ, του κυρίου Παβέλ Αντάμοβιτς. Τον ε, ήξερα ως εξέχοντα τοπικό αμ, πολιτικό δήμαρχο που έχει εκλεχθεί πολλές φορές και κάποιον ο οποίος πραγματικά ήταν ένα σύμβολο μιας ανοιχτής κοινωνίας που ήταν σε θέση να λειτουργήσει με τον υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποστηρίζοντας ε, τα δικαιώματα των μειονοτήτων όπου αυτές ε, υπήρχαν. Και θυμάμαι να λέει ότι στα δύσκολα, ναι, το Γκτάνσκ θα ήταν ανοιχτό να υποδεχτεί πρόσφυγες ε, που θα χρειάζονταν ασύλο στην Ευρώπη. Αυτό αποτελεί απλά ένα παράδειγμα των όσων ήταν σε θέση να πετύχει. Άρα ναι, είναι πραγματικά σοκαριστικό το γεγονός ότι έξαφνα όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιούμε για τους δημοκρατικούς θεσμούς αντικαθιστώνται από μαχαίρια και από δολοφονίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν μπορούμε να δεχτούμε. Και να είμαστε και ξεκάθαροι. Θα υποστηρίξουμε όσους υποστηρίζουν αυτή την ανοιχτή κοινωνία και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάση θυσία, όποιο και αν το τίμημα. Ο κύριος Καστάλντο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπω και εσεί υπενθυμίσατε πριν, σήμερα είναι μια θλιβερή μέρα, μια μέρα πένθουση για πολλού λόγου. Ακριβώ πριν από ένα μήνα ε, χάσαμε τον Αντώνη Μεγκαλίτσι, Μαζόν και μαζί και με τον κύριο Νετζιέλσκι από έναν αιματηρό φανατισμό. Ο δικό του ενθουσιασμό και η δέσμευσή του δεν πρέπει να ξεχαστούν. Πολλοί συνάδελφοι και αντιπροσωπείε τι ημέρε αυτέ εκφράστηκαν δηλώνοντα τη βούληση να του αποτίσουμε φόρο τομή. Και εγώ και ο συνάδελφο Κρασνοντέσκι, πέρα από την δική σα πρόταση, ε, που θέλετε να τους αφιερώσετε μία ραδιοφωνική αίθουσα, εμείς προτείνουμε να υπάρχει και ε, στο όνομά τους μία υποτροφία για τους νέους δημοσιογράφους που θα χρηματοδοτείτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί τα θύματα της δημοσιογραφίας είχαν αφιερώσει τη ζωή τους ε, χάρη στο project Eurofonica. Και με αυτή την πρωτοβουλία θέλουμε να αποτίσουμε φόρο τιμής ε, σε αυτά τα παιδιά και να συνεχίσουμε να ενισχύουμε την πορεία άλλων νέων δημοσιογράφων. Ε, και θέλω να δηλώσω την υποστήριξη των βουλευτών. Με αυτή τη μικρή χειρονομία θέλουμε να επαναλάβουμε το κράτος δικαίου και η λογική στην Ευρώπη ποτέ δεν θα ιτηθούν από τη βία και τον εξτρεμισμό. Ευχαριστώ. Πολλοί βουλευτές ζητούν το λόγο. Όμως, ξέρετε ποιο είναι πάντοτε το επιχείρημα. Εγώ θα έδινα το λόγο σε έναν από κάθε ομάδα, γιατί διαφορετικά κινδυνεύουμε να διαρκέσει μια ώρα η συζήτηση. Ο κ. Παπαδημούλης, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ εκ μέρου τη πολιτική μας ομάδα θα ήθελα να ενώσω τη φωνή μου με όσου συναδέλφου μίλησαν για τον θάνατο του δημάρχου του Γκτάνσκ όπως και για την δολοφονία του Ιταλού δημοσιογράφου πριν λίγες εβδομάδες στο Στρασβούργο. Νομίζω ότι ανεξάρτητα από τις πολιτικές μας διαφορές, όλες οι πτέρυγες του Ευρωκοινοβουλίου οφείλουν να είναι ενωμένες στην υπεράσπιση της δημοκρατίας, της ανεκτικότητας, του κράτους δικαίου, του πλουραλισμού, κόντρα στο μίσος, τη βία και το ρατσισμό. Σας ευχαριστώ. Έχουν ζητήσει το λόγο για Βαλέσα και Μοντέρο, τα Παρντέλ. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Δεν θα κάνουμε συζήτηση τώρα. Έχουμε καταδικάσει όλα αυτά τα θέματα και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη οι θέση. Παρακαλώ, κύριος Βαλέσα. Szanowni Państwo, Paweł Adamowicz Κυρίες και κύριοι, ο Πάβελ Αντεμόβιτς δολοφονήθηκε και έγινε θύμα του μίσους, ε, θύμα της ρητορικής του μίσους. Θα πρέπει να σκεφτούμε για το πώς ε, θα καταπολεμήσουμε τέτοιες συμπεριφορές και τέτοιες ρητορικέ ε, από τη δημόσια συζήτηση. Αυτή η τραγωδία ε, έγινε κατά τη διάρκεια μιας φιλανθρωπικής εκδήλωσης. Ο Πάβελ Ανταμοβίτς μιλούσε για αλληλεγγύη και για αδελφοσύνη που πρέπει να επιδεικνύουμε ένα τον άλλο και λίγο μετά τον μαχαίρωσαν. Λόγω αυτής της ε, ρητορική ε, του μίσους ε, συνέβη αυτό. Θα ήθελα να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι το Γκτάνσκ έχει χάσει τώρα έναν εξαιρετικό πατριώτη αλλά και φιλοευρωπαίο γιατί ο Πάβελ Αντάμοβιτς έχει καταλάβει ότι μπορούμε να είμαστε και πατριώτες αλλά και να οικοδημήσουμε μια καλύτερη Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν να τον θυμόμαστε. Σας ευχαριστώ. παρακαλώ. Κύριε Πιτσότα, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τα όσα ο Πρόεδρο και όλοι εσεί και να εκφράσω τα συλληπιτηριά μου για το χαμό του Δημάρχου του Ντάνσκ και να, υπενθυμίσω και τα θύματα εδώ στο Στρασβούργο. Όμως σήμερα θα ήθελα να στραφώ σε όλους εσάς, γιατί ίσως να μην ε, το ξέρετε, ότι ε, ο Τσέζαρ Μπατίστη με επιτέλους παραδόθηκε στην Ιταλική δικαιοσύνη, ένας τρομοκράτης που για πολλά χρόνια έχερε της καλυψή τόσων κυβερνήσεων και ευρωπαϊκών. Εγώ εύχομαι όλοι οι τρομοκράτες να παραδίδονται στη δικαιοσύνη και η γαλλική κυβέρνηση να ξαναδώσει, να ξαναπαραδώσει στην Ιταλία ε, τους τρομοκράτες τους οποίους προστατεύει. Συνάδελφος Βυσνιέσκα. Βυσνιέσκα. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, η δολοφονία του Παβέλα Αντάμοβιτ αποτελεί ένα παράδειγμα εξαιρετική βαρβαρότητα. Πρόκειται για μια μεγάλη τραγωδία για όλου μα. Πρόκειται για μεγάλο κακό και αυτό οδηγεί φυσικά σε καταδίκη της πράξης αυτής. Μεγάλη αδικία και μεγάλη λύπη λοιπόν αισθανόμαστε. Θα πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε πώς αυτό το κακό θα το ξεριζώσουμε από την δημόσια κοινή αυτή ζωή. Πώς μπορούμε να ξεριζώσουμε το μίσος αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι περνάει από το χέρι μας για να γίνουν αυτές οι ευαίσθητες συζητήσεις πιο α, ανώδυνες και να είναι πιο ασφαλές το κράτος στην Ευρώπη. Κυρία Τόγια. Ευχαριστώ. Θέλω να θυμίσω το έγγραφο που ψηφίσαμε σε αυτή τη συνεδρίαση. Ε, ε, είχαμε μάθει όλα αυτά τα τρομερά που συνέβησαν ε, στην πόλη όταν ο Αντώνιο και άλλα θύματα ε, επλήγησαν. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η πρόταση που έγινε την επόμενη μέρα του θανάτου του Αντώνιο, κυρίως από τη Σίλβια Κώστα, γιατί τον είχε γνωρίσει και είχε συνεργαστεί μαζί του και με το δίκτυο ε, του ραδιοφώνου του. Έτσι λοιπόν ε, θα έλεγα σήμερα ότι η ιδέα που ακούστηκε είναι εξαιρετική, να έχουμε αυτή την υποτροφία, αλλά και να τους αφιερωθεί ε, και μία αίθουσα τύπου, γιατί οι άνθρωποι αυτοί προήγαγαν τις αξίες. Όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι συνάδελφοι και να θυμόμαστε ότι ο καλύτερο τρόπο για να υπενθυμίζουμε τη θυσία του Αντωνίου και του συναδέλφου του είναι και εμεί να είμαστε καθημερινά φιλοευρωπαίοι και όχι μόνο στο δημοσιολόγο. Παρακαλώ, κύριο Δεγκράφ, και μετά κλείνουμε. Δεγκράφ. Και από τη δική μου πολιτική ομάδα και εγώ θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για τη φρικτή δολοφονία του κυρίου Αμπραμόβιτς. Πρόκειται για περιστατικά που κλειδονίζουν όχι μόνο την Πολωνία, αλλά θεωρώ όλες ε, τι βουλές της Ευρωπαϊκή Ένωση. και δυστυχώ. Δεν πρόκειται για την πρώτη τέτοια περίπτωση και πολύ φοβάμαι ότι δεν πρόκειται και για την τελευταία τέτοια υπόθεση. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια πολιτική ατμόσφαιρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι όλο και πιο βεβαρημένη τα τελευταία χρόνια. Η συζήτηση πλέον δεν διεξάγεται στις ολομέλειες, ε, αλλά στο δρόμο και αποτελεί σκηνικό. Το είδαμε και με τα κεντρινά γυλαίκα. Και βλέπουμε ότι το μήνυμα προς την πολιτική είναι ότι αντί να μιλάμε και να κοφεύουμε, θα πρέπει να ακούσουμε και τι ακούμε. Και αυτό θεωρώ ότι θα βοηθήσει το αίσθημα μίσους που επικρατεί στις περιπτώσεις αυτές. Τελευταία παρέμβαση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα θέμα πάρα πολύ επικαιρό και σχετικό γι' αυτό θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να καταδικάσει και ένα ακόμα κεφάλαιο της ιστορία της Βενεζουέλας. Έχουμε μια δραματική κρίση που βιώνει η χώρα όμως χωρίς ε, την ε, ε, αντίδραση της διεθνούς κοινότητας, ο Νικολάς Μαντούρο λαμβάνει τη δεύτερη θητεία του. Νομίζω ότι θα πρέπει εμείς να θετήσουμε ένα ψήφισμα που να προτείνουμε νέες προεδρικές εκλογές και να θεωρήσουμε ότι δεν είναι νόμιμη η δεύτερη θητεία του. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι στη Βενεζουέλα έχουν τρομερές, αντιμετωπίζουν τρομερές ελλείψεις στα φάρμακα και εγκαταλείπουν τη χώρα. Εγκαταλείπουν τη χώρα τους λόγω του φόβου και λόγω της βίας. Μιλάμε για ένα αποτυχημένο κράτος, για ένα κράτος ε, που τελικά ε, στέλνει πίσω τους Βενεζολάνους στη Μαδέιρα, ε, στην, στο δικό μου νησί. Εμείς θα πρέπει να υποστηρίξουμε τον λαό της Βενεζουέλα και να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς εδώ στην Ευρώπη. Κύριε Σταπαρτέλ. Κυρία Ταπαρντέλ, αγαπητοί συνάδελφοι. Πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να φέρω ένα ε, πρόβλημα που θίγει πολλά παιδιά τη Ρουμανία, αλλά και στην Κεντρική και στην Ανατολική Ευρώπη και πιστεύω ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αντιδράσουν άμεσα για την επίλυση αυτού του προβλήματο. Από την 1η Ιανουαρίου 2019 στην Αυστρία τέθηκε σε ισχύ ένας νόμος ε, βάσει του οποίου ε, τα παιδιά που προέρχονται από τη Ρουμανία και από την Ανατολική και Ανατολική Ευρώπη αλλά και οι γονεί του που εργάζονται στην Αυστρία είδαν τρομέρέ. Ε, περικοπές τα επιδόματα που λάμβαναν. Ένα τέτοιο μέτρο δεν μπορεί να επιτρέπεται σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης όπου τα ε, δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών καθιερώνονται από τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες και μάλιστα στην περίπτωση αυτή μιλάμε για ένα μέτρο που αφορά το μέλλον και την εκπαίδευση των παιδιών μας. Μου φαίνεται λοιπόν τρομερό το γεγονό ότι αυτοί οι εργαζόμενοι που έρχονται από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη συνεισφέρουν μεν στο κοινωνικό σύστημα της Αυστρίας, πληρώνουν τους φόρους τους στην Αυστρία ε, και δεν λαμβάνουν ε, τα ίδια επιδόματα και τα ίδια ωφέλη όπως οι Αυστριακοί πολίτες. Ζητώ λοιπόν και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο να αντιδράσουν ανάλογα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το καθήκον να επιβάλλει κυρώσει κατά αυτού του αυθαίρετου νόμου που υποσκάπτει το μέλλον δεκάδων χιλιάδων παιδιών. Δεν μπορούμε να δεκτούμε τέτοιες καταστάσεις. Σας ευχαριστώ. Στις 13 ε, Δεκεμβρίου έχουν εγκριθεί τα πρακτικά, έχουν διανεμηθεί, υπάρχουν παρατηρήσεις. Κατόπιν τη παρέτηση τη κυρία Στίνελ, το Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τον κανονισμό, διαπιστώνει τη, με θέση τη Μένη από την 1η Φεβρουαρίου 2019 και ενημερώνει την αρμοδιαρχή. Ο κύριο Τζέβι Χάρβερ έχει εγκαταλείψει του μη και προσχωρεί στο FTD από τι 10 Ιανουαρίου 2019. Αρμόδιε αρχέ Γερμανία μου έστειλαν ένα αίτημα άρση ε, τη ε, ασυλία τη κυρία Χολμάιερ προκειμένου η εισαγγελία του και να ξεκινήσει έρευνα σύμφωνα με τον κανονισμό, το αίτημα αυτό στέλνεται στην αρμόδια Επιτροπή Νομικών Θεμάτων από το FTD. Έχω λάβει αιτήματα τροποποίηση στη σύνθεση των Επιτροπών. Αυτέ οι τροποποιήσει θα τι δείτε στα πρακτικά τη συνεδρίαση αυτή. Αν δεν παρουσιαστούν παρατηρήσει μέχρι την υιοθέτηση των πρακτικών, οι τροποποίησει αυτέ θεωρείται ότι εγκρίνονται διάφορες επιτροπές αποφάσισαν να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσει ε, σύμφωνα με το άρθρο 69 C, παράγραφο 1 του ιστορικού κανονισμού. Οι έκθεσει που ε, αποτελούν τι εντολέ για τι διαπραγματεύσει είναι διαθέσιμε στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου και οι τίτλοι του θα δημοσιευτούν στα πρακτικά τη συνεδρίαση. Σύμφωνα με το άρθρο 69C, παράγραφος 2, ε, τα μέλη ή ε, πολιτικές ομάδες που φτάνουν τουλάχιστον ε, στο μέσο κατόφλι μπορούν να ζητήσουν μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα, 15 Ιανουαρίου, η απόφαση να μπουν σε διαπραγματεύσεις να τεθεί σε ψηφοφορία. Αν δεν υπάρξει τέτοια αίτηση, τότε μπορούν οι επιτροπές να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 46.2 ε, του ιστορικού κανονισμού έκανε αποδεκτή μία πρόταση για μία πράξη της Ένωσης για την πρόθεση της συλλογή πλάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υποβλήθηκε από τον κύριο Καπούτο και άλλα μέλη. Αυτή η πρόταση παραπέμπεται στην Επιτροπή Περιβάλλοντος που είναι αρμόδια. Μαζί με τον πρόεδρο του Κιβουλίου, την Τετάρτη υπογράψω έξι πράξεις που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την τακτική νομοθετική διαδικασία βάσει του άρθρου 58 ε, του εσωτερικού κανονισμού του Κοινοβουλίου και οι τίτλοι των πράξεων αυτών θα δημοσιευτούν στα πρακτικά της συνεδρίασης. Τώρα περνάμε στην ημερησία διάταξη. Έχει εγκρίνει σύμφωνα με το άρθρο 140. Έχει διανεμηθεί το σχετικό έγγραφο και σε ό,τι αφορά τη Δευτέρα η ομάδα των Πρασίνων ζήτησε να προσθεθεί ως τέταρτο σημείο πριν από τις παρουσιάσεις μια κοινή συζήτηση για δύο εκθέσεις, ε, έκθεση ΣΑΚΕ για την ε, Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Μαρόκου. Θα έχουμε παρέμβαση και από τις πολιτικές ομάδες. Ε, θα δώσω τώρα το λόγο για να παρουσιάσετε το θέμα. Ναι, Εάν ε, ε, χωρίς συζήτηση στην Ολομέλεια περάσει συμφωνία με το Μαρόκο, θα υπάρξει βεβαίως μια ε, νομολογία η οποία είναι κατά του διεθνούς δικαίου και είναι σημαντικό για τα κράτη-μέλη να ενημερωθούν, να ψηφίσουν. Επίσης βασίζεται στην έκθεση της κυρίας Βαλός που, που, για την οποία ίσως υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Επίσης δεν ξέρουμε αν η συμφωνία συμφωνεί ε, με την Ευρωπαϊκή Νομολογία και το Διεθνές Δίκαιο. Θα ήθελα λοιπόν να έχουμε αυτή τη συζήτηση και ζητώ από τον κύριο Σιμεσκόσκα ε, να ε, αναθεωρήσει την αντίρρησή του σε αυτήν την συζήτηση διότι δεν θέλει ανοιχτή διαφανή συζήτηση για το θέμα αυτό. Ποιο θέλει να μιλήσει κατά, παρακαλώ κυρία Ροντρίγκε, θέλετε να μιλήσετε κατά της πρότασης τη κυρίας Χαουτάλα. Against. Ε, because κατά διότι η ομάδα ε, των σοσιαλιστών είναι ανοιχτή για αυτήν την συζήτηση αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε τη συζήτηση αύριο το βράδυ και όχι σήμερα. Αυτό θα μας βοηθήσει να έχουμε μια ενδελεχέστερη θέση σχετικά με τη συζήτηση. Θέλουμε τη συζήτηση αλλά θέλαμε να την έχουμε αύριο το βράδυ διότι αν εάν ε, ε, ε, φτάσετε μέχρι τα μεσάνυχτα, ίσως να είναι αυτό εφικτό. Κυρία Χαουτάλα, θέλετε να διατηρήσετε τη θέση που εκφράσατε ή είστε διατηρημένοι να αλλάξετε, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή πρόταση από τους σοσιαλιστές και ο κύριος Βερχόφσαντ επίσης είναι υπέρ. Παρακαλώ, Να διευκρινίσουμε ε, η πρόταση που έκανα ήταν έτοιμα τεσσάρων συντονιστών, τεσσάρων ομάδων. Αν θέλετε λοιπόν μια συζήτηση, δεν έχω τίποτα εναντίον της συζήτησης, αλλά αυτοί οι τέσσερις συντενιστές της ΙΝΤΑ όταν ζητήσαμε να έχουμε αυτόν τον τρόπο εργασίας στη συζήτηση εγώ απλώς μετέφερα τη γνώμη τους και δεν έχει τίποτα να κάνει με την πολιτική και ελπίζω η κυρία Άουταλα να δει τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Εγώ συμφωνώ. Λοιπόν, να θέσουμε σε ψηφορία την πρόταση της κυρίας Χατάλα, έτσι όπως διορθώθηκε από την πρόταση της κυρία Ροντρίγκε. Ονομαστική ψηφοφορία, προκειμένου την Τρίτη το βράδυ να έχουμε ένα σημείο στη διάταξη πριν από τις σύντομες παρουσιάσεις. Δηλαδή ως τελευταίο σημείο θα μπει. Για το θέμα της συμφωνίας με το Μαρόκο. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η πρόταση. Λοιπόν, να περάσουμε στην τρίτη. Οι σοσιαλιστέ έχουν ζητήσει να αποσυρθεί από την επίσημη διάταξη δήλωση του Συμβουλίου και τη Επιτροπή για τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τη 13η και 14η Δεκεμβρίου. Επομένω, η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στι 9. Εξ ονόματο των Σοσιαλιστών, Ποιο θα παρουσιάσει την πρόταση. Παρακαλώ, κυρία Ροντρίγκε. Κανένα δεν θέλει να παρουσιάσει την πρόταση. Κάποιο θέλει να τοποθετηθεί κατά. Να περάσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία για το αίτημα. Καθώς ε, αποσιάζουν οι πρόεδροι Τούσκ και Γιούνκερ και αν κατάλαβα καλά αυτή ήταν η αιτιολογία για να αφαιρέσουμε από την ίδια διάταξη στο σημείο αυτό. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Επομένως εγκρίνεται η πρόταση, επομένως η δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα συμπεράσματα που από την ημερήσια διάταξη και θα ξεκινήσουμε αύριο τη συνεδρίασή μας στις 9. Έτσι λοιπόν, ορίστηκε και η μερίσια διάταξη. Περνάμε τώρα στις συζητήσεις που έχουμε για σήμερα το απόγευμα. Παρακαλώ, όσοι δεν θέλουν να παραμείνουν στο ημικύκλιο, ησύχως να αποχωρήσουν, παρακαλώ. Και όσοι παραμείνουν, επίσης να σιωπάσουν. Λοιπόν, να περάσουμε στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης ε, σε σχέση με την έκθεση των κυρίων Λίνς και Στάς ε, σε σχέση με την ε, διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έγκριση των φυτοφαρμάκων. Ο κύριος Λίνς, ο εισηγητής, έχει το λόγο. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα καλούμαστε να συζητήσουμε μέτρα τα οποία αφορούν την υγεία των 500 εκατομμυρίων πολιτών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ειδική λοιπόν επιτροπή του Κοινοβουλίου συζήτησε τη διαδικασία έγκρισης των φυτοπροστατικών ε, μέσων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βασικό στοιχείο στις εργασίες μας ήταν η ασφάλεια της δημόσιας υγείας. Εγώ ε, μεγάλωσα σε αγορόκτημα και όλη μου την παιδική ηλικία την πέρασα κοντά σε τέτοια μέσα και ξέρω πόσο σημαντική είναι η σωστή εφαρμογή και τι σημασία έχουν τα προστατευτικά μέτρα για την γεωργία. Εκ παραλίλου θα ήθελα να τονίσω ότι και τα δικά μου παιδιά και τα δικά σας παιδιά θέλουν να συνεχίσουν να μπορούν να τρώνε χωρίς να ανησυχούν λαχανικά και φρούτα από την Ευρώπη. Δύο πράγματα με απασχόλησαν. Καταρχά, λοιπόν, πώ θα συνεχίσουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα τρόφιμα τα οποία έρχονται στο τραπέζι μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ασφαλή. Και κατά δεύτερον, πώ θα εξασφαλίσουμε ότι και οι Ευρωπαίοι αγρότε θα μπορέσουν να συνεχίσουν σε μακροπρόθεσμο επίπεδο να παράγουν αυτά τα προϊόντα. Τι διαπιστώσαμε λοιπόν μετά από εννέα μήνε προσεκτική ανάλυση ε, ότι η διαδικασία έγκριση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πιο αυστηρή στον κόσμο καλό νέο. Αλλά φυσικά ο, και ο καλύτερος μπορεί να βελτιωθεί ακόμα παραπάνω. Και γι' αυτό λοιπόν ακολουθούμε μια εξέλιξη. Δεν θέλουμε επανάσταση, θέλουμε μια μεταξέλιξη του συστήματος, όχι να καταρρύψουμε το σύστημα. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να επικεντρωθούμε σε τρία σημεία. Καταρχάς, επιστήμη. Δεύτερον, διαφάνεια και ανεξαρτησία. Και τρίτον, καινοτομία. Επιστήμη λοιπόν, καταρχάς. Ήταν καθοριστικό παράγοντα το γεγονό ότι θα πρέπει η διαδικασία έγκριση να ακολουθεί επιστημονικά κριτήρια, γιατί σε πολλέ ε, σημαντικέ ε, αποφάσει το πιο σημαντικό είναι ε, το επιστημονικό σκέλο. Η απόφαση αυτή δεν μπορεί να αποφασιστεί από συναισθηματισμού και από πολιτικές σκοπιμότητες. Κατά δεύτερον, ανεξαρτησία και διαφάνεια είναι βασικό. Η αυτή παρα... η διαδικασία αυτή να παραμείνει διαφανής. Στο μέλλον, λοιπόν, θα πρέπει να αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι η βιομηχανία, ποια, ποιες ουσίες ε, επιτρέπονται και σε τι βαθμό και πώς ε, θα εγκρίνονται. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη δημόσια πρόσβαση στις μελέτες, αλλά θα πρέπει παράλληλα να μην ε, πληχθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Κατά τρίτον, καινοτομία. Θέλουμε να προωθήσουμε τις καινοτομίες. Νέα πιο αποτελεσματικά προϊόντα. Αυτά είναι το κλειδί για μια βιώσιμη καλλιέργεια. Και αυτό θα πρέπει να υποστηριχθεί από τη διαδικασία χορήγηση έγκριση. Επιτρέψτε μου λοιπόν μία μικρή πρόβλεψη στο μέλλον να κάνω. Η ψηφιοποίηση θα αλλάξει δραστικά το τοπίο της αγροτικής εκμετάλλευσης και εδώ θα πρέπει να μπούμε στο προσκήνιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ασχοληθεί επισταμένως με την διαδικασία έγκρισης των φυτοπροθεστικών μέτρων μέσων. Είμαι πεπισμένος ότι οι συστάσεις μας θα δημορφώσουν πιο αποτελεσματικό, διαφανή και στεναρό τρόπο τη διαδικασία αδειοδότηση τέτοιων ουσιών. Γιατί, γιατί δίνουμε υψηλή προστασία για τους καταναλωτέ και τους καλλιεργητέ, αλλά επιτρέπουμε και εγγυόμαστε και την γεωργική καλλιεργία και προωθούμε και τι καινοτομίε. Αυτέ τι συστάσει λοιπόν θα ήθελα την Τετάρτη να τι ψηφίσουμε με μεγάλη πλειοψηφία. σα. ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον Παρτιστά τον συγητή μου για την καλή συνεργασία, αλλά ευχαριστώ και όλους τους υπόλοιπου σκιώδεις εισηγητές και προσβλέπω στην ε, συζήτησή μα σήμερα και στην ψηφοφορία την Τετάρτη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σαστάς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι, κύριε Επιτροπέ. Ένα εκατομμύριο 786.000 πολίτες έχουν εκκινήσει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για να μας ζητήσουν μεταξύ άλλων να, να εξετάσουμε τη διαδικασία αντιοδότηση φυτοπροστατικών μέτρων και να την μεταρρυθμίσουμε. Αυτή λοιπόν η έκθεση αποτελεί απόδειξη ότι αυτό το αίτημα το παίρνουμε στα σοβαρά και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα γιατί καταρχάς το θέμα είναι να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στη διαδικασία λήψη αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι πολίτες λοιπόν θα πρέπει τυφλά να εμφυστεύονται ότι όταν λαμβάνουμε μία απόφαση, αυτή η απόφαση βασίζεται στο κοινό συμφέρον και όχι στα ιδιωτικά συμφέροντα λίγων και κάποιων οργανώσεων τις βιομηχανίες. Εδώ λοιπόν προβαίνουμε σε συστάσεις. Αυτό που είπε ο κ. Λίντς στέκει ο συνεισηγητής μου. Αναγνωρίζουμε ότι η διαδικασία, μάλλον διαπιστώσαμε ότι ο τρέχοντα μηχανισμό είναι από του πιο αυστηρού, ο πιο αυστηρό στον κόσμο, αλλά παράλληλα αυτά επιτέχεται βελτίωση. Εδώ κοιτάμε λοιπόν στην ε, εφαρμογή. Τι γίνεται. Καταρχά, θέλουμε να εφαρμοστεί η αρχή τη πρόληψη και κατά δεύτερον, θα πρέπει να φροντίσουμε η διαδικασία λήψη αποφάσεων για τα φύτα προστατευτικά να γίνεται με ανεξάρτητο, αντικειμενικό και διαφανή τρόπο. Μόνο τότε θα κερδίσουμε εκ νέου την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών. Για το γλυφωσάτι, λοιπόν στην Επιτροπή ΠΕΣΤ διαπιστώσαμε ότι δεν έχει ακόμα επιληθεί α, το επίμαχο αυτό θέμα. Δεν το επιλύσαμε αυτό το θέμα στην Επιτροπή μας. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε ο μηχανισμός, ο επιστημονικός μηχανισμός συμβουλευτικής ο οποίος προσφέρθηκε να ξεκινήσει μια συστηματική ανάλυση όλων των εφιστάμενων μελετών για ενδεχόμενες καρκινογόνες επιπτώσεις της γλυφοσάτης προκειμένου να αναλύσουμε κατά πόσο χρειάζεται μεταρρύθμιση της διαδικασίας έγκρισης που έχουμε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε διαφάνεια και ανεξαρτησία. Διαφάνεια. Θέλουμε ο ετών να υποχρεούται να καταχωρεί τα αιτήματά του σε ένα δημόσιο μητρό και θέλουμε πρόσβαση σε αυτό το μητρό να έχουν όλοι οι πολίτες προκειμένου όλα τα υποστηρικτικά στοιχεία, τα τεκμήρια, οι μελέτες να είναι ελεύθερες, να μπορεί να τις ε, συμβουλεύεται ο πολίτης και να ελέγχει κατά πόσον έχουν ακολουθηθεί ίσως τις διαδικασίες. Ζητούμε επίσης από τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της μόνιμης ε, επιτροπής που οφείλεται, στην οποία μάλλον ε, επαφίεται η λήψη αποφάσεων για τα κράτη-μέλη. Θέλουμε πλήρη δημοσιοποίηση του πώς ψηφίζει ο καθένας. Θέλουμε επίσης τα αιτήματα να μην ε, ορίζεται ποιο θα εξετάσει τα αιτήματα από τα κράτη-μέλη, να, να το ορίζει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θέλουμε σωστέ ε, επιστημονικά τεκμήρια, να υπάρχουν σωστέ διαδικασίε εσωτερικά για να αποτρέπονται συγκρούσει συμφερόντων. Θέλουμε επίσης να υπάρχουν και να προβλέπονται επαρκή πόροι και για την ΕΦΣΑ και για την ε, Ευρωπαϊκή Οργανισμό Χημικών Προϊόντων. Θέλουμε επίσης και από τον Horizon να χρηματοδοτήσει προγράμματα ανεξάρτητης έρευνας και για τον αντίκτυπο στην υγεία του κόσμου και των ζώων, αλλά και για το περιβάλλον. Τέλος, έχουμε το θέμα ενδεχόμενης ε, κλοπής πνευματικών δικαιωμάτων. Μπορεί κάποιος να κάνει copy-paste, δηλαδή, τα αιτήματα των ετώντων και να τα χρησιμοποιήσει ο ίδιος σε του σκοπούς. Θέλουμε τέτοια αντιγραφή δεδομένων να γίνεται όσο πιο λίγο γίνεται, όσο πιο σε περιορισμένο βαθμό γίνεται. Και αν γίνεται να δηλώνεται τουλάχιστον. Στην έκθεσή μας δίνουμε μεγάλη σημασία στο μακροπρόθεσμο επίπεδο τοξικολογική ανάλυση των ε, φυτοπροστατευτικών ε, σε ό,τι αφορά όλες τις επιπτώσεις των ε, φυτοφαρμάκων σε ό,τι αφορά το σωρευτικό χαρακτήρα που μπορεί να υπάρχει. Θέλουμε επίσης ε, τα κριτήρια του άρθρου 5 να συνεχίζονται να εφαρμόζονται χωρίς ε, καμία εξαίρεση, γιατί έχουμε διαπιστώσει ότι αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Θέλουμε επίσης ε, να μην χρησιμοποιείται η γλυφοσάτη σε πάρκα, σε σχολεία, σε παιδικές χαρές, σε αθλητικά γήπεδα κτλ και κοντά σε νοσοκομεία. Και τέλο, ε, το άρθρο 53 είναι το άρθρο που προβλέπει τι εξαιρέσει. Αυτό το άρθρο πλέον ε, χρησιμοποιείται υπερβολικά συχνά ω μία μόνιμη εξαίρεση. Δεν μπορεί να είναι μόνιμη με τέτοια εξαίρεση. Και τέλο, προ την κυρία Χάζενκαμ από την Ολλανδία, θα πρέπει να κοιτάξουμε να αποφεύγουμε, να μειώσουμε και να υποκαταστήσουμε τελικά τις δοκιμές στα ζώα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ανδρουκαίτης έχει το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τα αξιότιμα μέλη. Βεβαίως οι Ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν να έχουν ασφαλή τρόφιμα και ενώ βεβαίως η ασφάλεια των τροφίμων είναι επίγουσα ανάγκη, αλλά δεν αρκεί από μόνη της όλο και περισσότερο οι πολίτες ενδιαφέρονται για το πώς τα τρόφιμα παράγονται και για την βιωσιμότητα της παραγωγής και για την προστασία του περιβάλλοντος. Μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προσδοκίες αν μαζί διδαχθούμε από τις πρόσφατες προκλήσεις και δράσουμε προς όφελος όλων των πολιτών. Μέσα στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο διότι ε, έχετε ε, θεσπίσει αυτή την ειδική επιτροπή σχετικά με τα φυτοφάρμακα της αγοράς πέρυσι ε, και έχουμε την έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας για την βιώσιμη αηφόρο εφαρμογή των φυτοφαρμάκων και για το θέμα της γλυφοσάτης. Η εργασία της Επιτροπής είναι πάρα πολύ σημαντική διότι θέλουμε να εξασφαλίσουμε όλη η διαφάνεια ε, και συστήματα ασφάλειας τροφιμένων που να βασίζονται σε αποδείξεις, να μην υπάρχουν αμφιβολίες μεταξύ των πολιτών ως προς την ουδετερότητα της επιστήμης. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η επιστήμη είναι ε, τέλεια και ότι δεν μεροληπτεί και ότι είναι ουδέτερη. Αυτή η ειδική επιτροπή ε, ιδρύθηκε ε, το Δεκέμβριο 2017 για την, την έγκριση της γλυφοζάτης για ακόμα πέντε χρόνια για να αναλυθεί το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έγκριση ουσιών και ε, την έγκριση φυτοπροστατευτικών ουσιών και για να εντοπιστούν τομείς που μπορούν να βελτιωθούν. Ε, τα, τα συμπεράσματα της Επίτροπης ΠΕΣΤ είναι η ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο σύστημα το ενωσιακό ε, στην αξιολόγηση των ουσιών εμπιστοσύνη ε, στην, στην διαχείριση των κινδύνων. Βεβαίως χρειάζεται πολύ μεγάλη διαφάνεια και όλες οι μελέτες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως βάση για την αξιολόγηση κινδύνων και να είναι διαθέσιμες. Επίσης, οι συζητήσεις, οι θέσεις της Ρυθμιστικής Επιτροπής που αποφασίζει ποιες ουσίες πρέπει να εγκριθούν, πρέπει οι εργασίες να είναι διαφανείς μπορούμε ε, με βεβαιότητα να πούμε ότι από πέρσι διανύσαμε μεγάλο δρόμο. Η πρόταση του Απριλίου 18 από την Επιτροπή για την διαφάνεια και βιωσιμότητα στην τροφική αλυσίδα αποβλέπει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο σύστημα. Ακολουθεί πολλές συστάσεις Επιτροπής ΠΕΣΤ. Διαφάνεια κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης κινδύνων επίσης ποιότητα των μελετών και αύξηση της επικοινωνίας. Όπως είπα το Δεκέμβριο στη συζήτηση για την πρόταση αναθεώρησης του Γενικού Νόμου για τα τρόφιμα, ε, πολλοί εξέφρασαν έτοιμα για περισσότερες διαφάνεια, για περισσότερη διαφάνεια στην αξιολόγηση κινδύνων. Ε, και ακούμε τους πολίτες ε, και ε, βρούμε για το θέμα αυτό από την αρχή της θητείας μας. Έχουμε επίσης το ψήφισμα που ψηφίσατε πριν από ένα χρόνο, όπου τονίζεται ότι η, διαδικασία έγκρισης Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αξιολόγηση επιστημονική των ουσιών θα πρέπει να βασίζεται μόνο σε δημοσιευμένες μελέτες. Νομίζω ότι με μεγαλύτερη διαφάνεια μπορούμε να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο σύστημα αξιολόγησης κινδύνων. Αυτή η διαφάνεια θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε την μεροληψία και να έχουμε ένα σύστημα ασφαλείας που να χέρι εμπιστοσύνη, όπως και η επιστήμη. Αυτή η πρόταση μα βοηθάει πολύ από την άποψη αυτή. Σα. ευχαριστώ άλλη μια φορά για την ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον περισμένο μήνα και τον επικοδομητικό τριμερή ε, διάλογο. Λόγω της σημασίας του θέματος αυτού για τους Ευρωπαίους πολίτες, ξέρω ότι θα προοδεύστε στις συζητήσεις με το Συμβούλιο για να μπορέσει να βρεθεί μια συμφωνία σε αυτήν την θητεία. Βεβαίως μπορείτε να βασιστείτε σε μένα και στις υπηρεσίες μου, ώστε να συνεργαστώ μαζί σας για να επιτύχουμε αυτήν, αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ ως ενδιάμεσος έχουμε πολύ καλή συνεργασία. σχετικά με το θέμα της έκθεσης αυτής. Ε, ο νέος κανονισμός θα μπορούσε να εμφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό για τον τομέα των φυτοφαρμάκων, αλλά στον τομέα των φυτοφαρμάκων έχω λάβει ορισμένα μέτρα για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των ε, πολιτών απέναντι στις αποφάσεις και αξιολόγηση κινδύνων, όπως για τη γλυφοσάτη, τα νοικοτινοειδή ε, και για τους διαταράκτες της ενδοκρινικής λειτουργίας. Έχουμε έναν ιστότοπο ο οποίος αναφέρει όλες, όλα τα στοιχεία ε, του σχεδίου ε, πρότασης και των συζητήσεων των κρατών μελών. Επίσης, η Επιτροπή έλαβε πολλά αιτήματα για πρόσβαση στα έγγραφα σχετικά με τα φυτοφάρμακα. Από τον Απρίλιο όλα ε, τα έγγραφα είναι προσβάσιμα δημόσια. Επιπλέον, με την πρόταση που αναθεωρεί την επιτροπολογία θέλουμε να αυξήσουμε την διαφάνεια στο επίπεδο αυτό, ούτως ώστε ε, να έχουμε τη θέση των κρατών ε, που να κοινοποιούνται δημόσια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει από τα πιο αυστηρά συστήματα στον κόσμο για τη ρύθμιση των φυτοφαρμάκων. Αλλά υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωση. Συμφωνώ. Δεν υπάρχει ποτέ τέλειο σύστημα. Είναι πάντοτε δυνατόν να βελτιωθούν οι διαδικασίες ε, για την έγκριση των φυτοφαρμακευτικών ουσιών Υπάρχει ένα πρόγραμμα απόδοσης ε, για να βελτιωθεί η νομοθεσία που περιλαμβάνει ε, ε, τα προϊόντα φυτοπροστασίας, τα προϊόντα, τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων. Οι εργασίες αυτές θα ολοκληρωθούν σύντομα και θα δούμε πού χρειάζονται βελτιώσεις και θα ήθελα να το Κοινοβούλιο να εστιαστεί πάνω στο σύστημα αυτό με την Επιτροπή ΠΕΣΤΑ και την έκθεση αυτή. Επίσης εξετάζεται ο κανονισμός για την φυτοπροστασία και θα υπάρξει μια μελέτη για το θέμα αυτό. Έχουμε επίσης τα μηχανήματα, τα, τις μηχανισμούς του συμβουλευτικούς και του ε, τους ελέγχους των υπηρεσιών της Επιτροπής στα κράτη-μέλη. Όλα Όλα αυτά τα στοιχεία ε, θα περιληφθούν στις αναλύσεις της Επιτροπής ενώ θα προχωρούμε. Ε, και η Επιτροπή ΠΕΣΤ επίση παρέχει πολλά στοιχεία για αυτή την άσκηση. Έχουμε λοιπόν ανάγκη από βελτιώσεις και θα έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο είναι απαραίτητο και θα πρέπει η επόμενη βεβαίως Επιτροπή να δει αν θα προτείνει αλλαγές στην νομοθεσία που ε, θα πρέπει τελικά να υιοθετηθούν από το Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Αξιότιμα μέλη για να κλείσω. Θα ήθελα να τονίσω ότι έχουμε όλοι έναν ίδιο στόχο, να διατηρήσουμε την ασφάλεια των τροφίμων, να προστατεύσουμε τους πολίτες, τα ζώα, τα φυτά. Σας ευχαριστώ για την δέσμευση της Επιτροπής ΠΕΣΤΑ και για την δική σας δέσμευση και συγχαίρω ε, τον ε, πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τους συνεισηγητές, ε, Λίντς και Στάς και τους κοιόδης εισηγητές. Περιμένω την τελική έγκριση την Τετάρτη και σας διαβεβαιώνω ότι τα συμπεράσματά σας θα ληφθούν υπόψη, θα εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε αδιάκοπα για την διαφάνεια, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και για την διατηρησιμότητα και βιωσιμότητα. θα υποβληθούν τα συμπεράσματά σας, τόσο ώστε να βελτιώσουμε την νομοθεσία σχετικά με τα φυτοφάρμακα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πίτροπε. Κυρία Γιούσο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, καταρχήν ε, θα ήθελα να συγχαρώ τους δύο εισηγητές ε, για το πολύ καλό έργο τους και εσάς ε, κύριε Πέτροπε, για τη συμμετοχή σας σε αυτά τα ευαίσθητα ζητήματα. Στην Επιτροπή εδώ και μήνες εργαζόμαστε και ακούσαμε τους εμπειρογνώμονες, αναλύσαμε τις διαδικασίες ε, τόσο ενωσιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών σε σχέση με την έγκριση των φυτοφαρμάκων. Εγώ συμμερίζομαι τους στόχους διαφάνειας προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών ή να το σχετικό και να προστατευτεί η ανθρώπινη υγεία. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να αποφύγουμε να αμφισβητούνται τα αποτελέσματα των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ε, λόγω ιδεολογικών παραγόντων και να αμφισβητείται η ικανότητα καινοτομία και ανταγωνιστικότητα. Αν ε, λάβουμε υπόψη την διαδικασία έγκριση των φυτοπαρμακών, θα πρέπει η συζήτηση να γίνει σε τεχνικό και επιστημονικό επίπεδο. Οι αποφάσει για τα φυτοφάρμακα θα πρέπει να λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει επιστημονικών κριτηρίων, χωρί ε, πολιτική ανάμειξη. Εγώ ε, ως ε, αρμόδια επικοινωνίας με την ΕΦΣΑ ε, θέλω να πω ότι είναι αμερόληπτος αυτός ο οργανισμός και βασίζεται το έργο του στον ισχύοντα κανονισμό. Όμως να μην ξεχνάμε ότι η διαδικασία που χρησιμοποιήσει η Ένωση για την έγκριση των φυτοπροσταυτικών προϊόντων είναι μία από τις πιο αυστηρές παγκοσμίω. Βέβαια δεν υπάρχει μηδενικός κίνδυνος και η χρήση των προϊόντων αυτών επίσης ενέχει κινδύνους που πάντα μπορεί να ελαχιστοποιηθούν και αναφέρομαι, παραδείγματο χάρη, στι ε, δόσεις εφαρμογή και στη διαδικασία εφαρμογή. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον για να κλείσω η Επιτροπή να παρουσιάσει μία ανακοίνωση προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της αναθεώρησης της νομοθεσίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με στόχο να ενοποιηθούν κριτήρια και να ομολογοποιηθούν οι διαδικασίες ανάλυσης κινδύνου. Εγώ νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γιούσο, η κυρία Μποναφέ. Ευχαριστώ πρόεδρε με τις εργασίες της ΠΕΣΤΟ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήθελε να παρουσιάσει τα κύρια προβλήματα και να απαντήσει στις κύριες επικρίσεις που αφορούσαν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκρισης ε, Φυτοφαρμάκων. Με μεγάλη πλειοψηφία ψηφίστηκε η έκθεση και η Επιτροπή ήθελε να απαντήσει ξεκάθαρα στους εκατομμύρια πολίτες που τα προηγούμενα χρόνια ε, μίλησαν για την έλλειψη δαφάνεια του συστήματο μέσω τη πρωτοβουλία Stop Glyphosat. Ε, προκειμένου να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στο σύστημα και να διασφαλίσουμε ότι οι στόχοι τη ανθρώπινη υγεία και του περιβάλλοντο είναι κυρίω στόχοι τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτά είναι απαραίτητα σημεία επί των οποίων σταθήκαμε. Καταρχήν η διαφάνεια, η ανεξαρτησία και η έλλειψη σύγκρουση συμφερόντων στα επιστημονικά πάνελ τη ΕΦΣΑ. Προβλέψαμε κάθε μέλο, θα πρέπει να παρουσιάσει μία δήλωση συμφερόντων. Η κατανομή Ω δεύτερο σημείο των οικονομικών πόρων, μάλλον επαρκών πόρων στι αρμόδιες αρχέ για την αξιολόγηση των κινδύνων και κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη για τη διαδικασία τη έκθεση. Η τελική έκθεση καλύπτει και πολλέ άλλε πτυχέ που αναφέρθηκαν σε προηγούμενες παρεμβάσεις και που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διαδικασία αναθεώρησης του κανονισμού, Όπω το αίτημα τη δημιουργία ενό μηχανισμού εποπτείας μετά τη θέση εμπορία εμπορίας, που να μπορεί να παρακολουθεί τα αποτελέσματα στην πραγματική ζωή τη χρήση των φυτοπαραγματών. Ε, ε, την ομάδα των σοσιαλιστών πρέπει να δώσουμε προσοχή στην αξιολόγηση των κινδύνων για τι πιο ευπαθεί ομάδε και αναφέρομαι συγκεκριμένα στη χρήση των φυτοφαρμάκων κοντά στα σχολεία, στα νοσοκομεία ή σε δημόσια πάρκα. Επίση, είναι απαραίτητο να επενδύσουμε στην καινοτοπία για να αναπτύξουμε εναλλακτικά ε, τέτοια αυτοπροστατευτικά προϊόντα. Αυτό είναι απαραίτητο, όπως ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο, να υπάρχει και συγκεκριμένος κανονισμός για φυτοφάρμακα με χαμηλό κίνδυνο. Εύχομαι να υπερψηφιστεί την Τετάρτη η έκθεση, καθώς αποτελεί ε, ουσιαστικά ένα πολύ καλό αποτέλεσμα της εργασίας των δύο εισηγητών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μποναφέ. Η κυρία Μακεντάιρ. E Η διαδικασία έγκριση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα φυτοπροστατικά προϊόντα αποτελεί μία από τι πιο αυστηρέ σε όλο τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, αν διαβάζοντα την έκθεση τη Επιτροπή ΠΕΣΤ, δεν θα το θεωρούσε κανεί αυτό Παρά το γεγονός ότι μια σειρά επιστομών και εμπειρογνωμόνων μας αναφέρουν κάτι τέτοιο, η έκθεση επικεντρώνεται σε πολύ περιορισμένο τρόπο και πολλές από τις μαρτυρίες αυτών των εμπειρογνωμόνων αγνοούνται. Το περιεχόμενο δεν αποτυπώνει αυτά που ακούσαμε, αλλά επαναλαμβάνει τις ίδιες πεπιθήσεις και τους ίδιους μύθους που είχαμε στην αρχή της διαδικασία. Ακόμα και αν το γεγονός είναι ότι αυτό ομόφωνα το απέρριψαν οι εμπειρογνώμονες. Ε, για την αδυναμία των, ε, του συστήματος ε, του κράτους μέλους του ΝΤΑ σε ό,τι αφορά την αποτυχία του συστήματος κτλ. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι παραμένει στην έκθεση παρά το γεγονός ότι έχει απορριφθεί από τους, επιστήμονες από επιστήμονες και τους εμπειρογνώμονες για να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα για, τις για την προεκλογική διαδικασία το Μάιο. Αυτό λοιπόν δίνει φτωχά αποτελέσματα και παρουσιάζει με άσχημο τρόπο την κοινοβουλευτική μας εργασία και γι' αυτό υποβάλαμε τροποποιητικές ε, προτάσεις, τροπολογίες για να ακούσουν οι συνάδελφοι και την άποψη αυτή και όχι μόνο τις επιλεγμένες αυτές απόψεις κάποιων ευρωβουλευτών. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε λοιπόν ποια είναι η άποψη των εμπειρογνωμόνων για τα θέματα αυτής της πολιτικής και πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα διαπιστώσει την αξία τη διαδικασία και θα υποστηρίξει τις τροπολογίε του ECR. Το σύστημά μας σύμφωνη δεν είναι τέλειο. Μπορεί να βελτιωθεί. Μπορούμε να βελτιώσουμε τη διαφάνεια, το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη το έχει πράξει στην πρόταση για τη μεταρρύθμιση του Γενικού Νόμου για τα τρόφιμα. Μπορούμε να ενθαρρύνουμε την καινοτομία, να υποστηρίξουμε νέε μεθόδου καλλιέργεια για τη μείωση των φυτοπροστατευτικών και να χρησιμοποιούμε ουσίες που θα υποκαταστήσουν πιο παλιές και παροχημένες ουσίες. Ε, ο εμπειρογνώμονας της Greenpeace στην τελική ακροασή είπε ότι δεν πρόκειται για αδυναμία της νομοθεσίας. Το θέμα είναι η βελτίωση της εφαρμογής. Αυτό χρειάζεται. Άρα η έκθεση αυτή θα πρέπει να βρει την ισορροπία και σε ό,τι αφορά τις μαρτυρίες των επιστημόνων ακόμα και αν αυτό δεν βολεύει κάποιες πολιτικές ομάδες για την προεκλογική τους εκστρατεία. Ευχαριστώ. κυρία Ρίς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, πολλές εργασίες, τρεις αποστολές στο εξωτερικό, οκτώ συνεδριάσεις, μια εντολή σαφής δεν ξέρω. Το σύστημα έγκρισης ε, νομίζω δίνει ιδέες για το μέλλον. Αυτό το είπαμε με την ανανέωση το τέλος του 2017 για την έγκριση της Γλυφοσάτς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εισήγητες για την πολύ καλή συνεργασία και τον Ερικόντριο, ένας πρόεδρος απαιτητικός, ένας πρόεδρος που έχει ενσυναίσθηση οι συστάσεις τις οποίες κάνουμε είναι επίγουσες και δύνατες. Νομίζω ότι η έκθεση ΠΕΣΤ λαμβάνει υπόψη την υγεία ε, των πολιτών. Είδαμε ποια είναι τα κενά στην διαδικασία έγκρισης και προτείνουμε έναν κατάλογο συστάσεων που θα πρέπει να εφαρμοστούν αμέσως από τα κράτη-μέλη. Πρώτη απέτηση, και αυτό το λέμε για την ΕΦΣΑ, οι εμπειρογνώμενες οι οποίοι εργάζονται με την βιομηχανία θα πρέπει να αποκλείονται από την διαδικασία έγκρισης των φυτοφαρμάκων. Σημαντικό για τη διαφάνεια να υπάρξει ένα δημόσιο μητρό που θα αναφέρονται αναφέρονται τα στοιχεία και οι μελέτες που χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία. Ζητούμε επίσης η Ευρώπη να αυξήσει τον προπολογισμό της ΕΦΣΑ για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του οργανισμού και είναι ο προπολογισμό τέσσερις φορές μικρότερος από τον οργανισμό για τα φάρμακα. Η ασφάλεια των τροφίμων αξίζει πολύ ε, περισσότερα. Ε, για ε, τους μολυσματικούς ε, παράγοντες, τους τρόφιμογενείς. Έχουμε, πρέπει να μελετηθούν οι επιπτώσεις πάνω στον καρκίνο. Η ερώτησή μου, κύριε Επίτροπε, πότε εσείς θα εφαρμόσετε τον νόμο και θα δημοσιεύσετε τον πρώτο αρνητικό κατάλογο, δηλαδή απαγόρευσης των βοηθητικών ουσιών που είναι στο επίκεντρο της τοξικότητας των προϊόντων. Πρέπει η Ευρώπη να προωθήσει μια πολιτική για τους δημόσιους χώρους, τους βρεφικούς σταθμούς, τα ε, σχολεία, τους χώρους άθλησης ε, παιχνιδιού ε, και να απαγορευθούν πολύ περισσότερα προϊόντα. Νομίζω τελικά και κλείνω κύριε Πρόεδρε, η Ευρώπη δεν έχει επιλογή, θα πρέπει να ακολουθήσει τη συμπεράσματα της Επιτροπής ΠΕΣΤΑ που θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο των αποφάσεών μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βάιτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συχνά 10-15% των ε, απόψεων μιλούν για επικίνδυνα φυτοπροστατευτικά. Αλλά ποια είναι η τιμή των ε, φυτοπροστατευτικών αν τελικά ε, χαθεί η βιοπικιλότητα, αν ε, δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα στο σύστημα υγείας. Όλα αυτά λοιπόν οδηγούν σε απόλυση, έχουν κόστος. Αυτό θα κληθούμε εμείς να το πληρώσουμε. Προφανώς κάποια φυτοφάρμακα δεν είναι ασφαλή. Προκαλούν ζημιά στους πολίτες, αλλά σας παρακαλώ να διευκρινίσουμε το εξής. Με τη διαφάνεια και με τον έλεγχο των ομίλων και με την πιο αυστηρή τήρηση των κριτηρίων για το περιβάλλον και για την υγεία σε ό,τι αφορά τα φυτοφάρμακα και στον έλεγχο και στις δοκιμές. Σας ζητώ λοιπόν να υποστηρίξετε την εκθέση αυτή. Κυρία Μάκινταϊρε, υποστηρίζετε μία ομάδα, ιδεολογική άποψη μιας ομάδας. Τι εννοείτε ότι πρέπει να βρούμε μία, ένα συμβιβασμό με την ΟΕΛΚ, με την ΚΟΕ, με τους φιλελεύθερους. Όλοι εδώ στο, στην αίθουσα είναι υπέρ. Μόνο εσείς, ε, κυρία Μακιντάιρ, έχετε υποβάλει τέτοιες τροπολογίες για να διαλύσετε την έκθεση αυτή και να σκύψετε μπροστά στι ε, επιχειρήσει, στη βιομηχανία. Δεν νομίζω ότι αυτό περιμένουν από εμά οι πολίτε μα. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάζενκαμπ. Η έγκριση από πλευρά της Ευρώπης ε, τη. Ε, γλυφοσάτη τη Μοσάντο αποτελεί ένα μεγάλο σκάνδαλο. Έχει περάσει πάνω από ένα χρόνο που η Μοσάντο η ΕΦΣΑ τη Γερμανική Επιτροπή, το Βοηνικό Ίδρυμα Υγείας ε, ε, υπέβαλαν τέτοιε απόψει σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτέ οι αποφάσεις έλαβαν χώρα βάσει αμφίβολων μελετών που είχε υποβάλει η βιομηχανία. Η Ευρώπη λοιπόν θεωρώ ότι αναλαμβάνει ε, απαράδεκτο ρίσκο για την υγεία των 500 εκατομμυρίων πολιτών και των ζώων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν Επιτροπή ε, επιτρέπει όλο και πιο πολύ ε, δηλητήριο στα, στο περιβάλλον, στο σώμα μας, ε, στα νερά μας. Και γι' αυτό λοιπόν δημιουργήθηκε αυτή η ειδική επιτροπή για να εξετάσει τη διαδικασία χορήγησης έγκρισης στα φυτοφάρμακα και κατά από την σύσταση της Επιτροπής αυτής για την έγκριση των φυτοφαρμάκων, τα πράγματα είναι πλέον αισιόδοξα. Η Ευρώπη θα πρέπει να εφαρμόζει πιο αυστηρά κριτήρια. Θα πρέπει να χρησιμοποιεί λιγότερο δηλητήριο, λοιπόν, συνολικά. Και στου δημόσιου χώρου θα πρέπει να απογορεύεται η χρήση δηλητηρίου. Τα ζώα δεν μπορούν να συνεχίζονται να τη χάνουν κακομεταχείριση υπό το, τη δικαιολογία της ασφάλειας και πρόκειται για πολύ καλές συστάσεις τις οποίες το κόμμα για τα ζώα τις προσυπογράφει και χαίρομαι που τα αγκαλιάζει αυτά τα στοιχεία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μένουν, ε, στην, μένουν και στην νομοθεσία για τα τρόφιμα. Θα πρέπει λοιπόν αυτά να αποτελέσουν στοιχεία του παρελθόντος. Η γλυφοσάτη θα πρέπει να βγει από την αγορά. Και αυτό ζήτησαν άλλωστε και ένα εκατομμύριο πολίτες. Και επίσης πρέπει να, ότι θα πρέπει να καταργηθούν οι αγροτικές επιδοτήσει. Ευχαριστώ πολύ, η κυρία Ντορνανό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε κύριοι συνσηγητές, κυρία Επίτροπη, το Μάρτιο του 2017 η Ομοσπονδιακή Δικαιοσύνη των ΙΠΑ αποκάλυψε πάνω από 200 ε, σελίδες εσωτερικών ε, εγγράφων. Το περιεχόμενά τους ε, αποδεικνύει ότι οι αγροχημικές εταιρείε ανησυχούσαν εδώ και 20 χρόνια για μεταλλαξιογόνες συνέπειες του γλυφοσάτ, τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται περισσότερο τον κόσμο όμως την προηγούμενη των αποκαλύψεων δημοσιεύτηκε μία έκθεση από τη βιομηχανία αυτή που θεωρούσε την κλειφωσάτη ούτε καρκινογόνο ούτε μεταλλαξιογόνα. Όμως ε, ξέσπασε το σκάνδαλο και είχε παγκόσμια συνέπεια. Στα τέλη του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε παραδεκτή την ε, πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών ε, για την απαγόρευση του γλυφοσάτ και την προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτών από τα τοξικά φυτοφάρμακα. Υπεγράφει έτσι αυτή από πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες και λίγο μετά δημιουργήθηκε μια ειδική επιτροπή για τα φυτοφάρμακα φάρμακα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ ε, παρακολούθησα το σύνολο των ακροάσεων που ε, οργανώθηκε με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων για τη διαδικασία της έγκρισης. Μπορώ να πω ότι εξεπλάγει ε, από την αμφισημία και από τα κατάφορα ψέματα που ακούστηκαν από κάποιους ψεύδο ε, ε, επιστήμονες που υπεράσπιζαν τα φυτοφαρμακά. Είχαμε 1.141 τροπολογίες που κατατέθηκαν στην Επιτροπή ε, λόγω ε, αυτού του σχεδίου έκθεσης που λάμβανε εντελώ ανταγωνιστικές θέσεις. Σήμερα στην Ολομέλεια έχουν κατατεθεί 152 τροπολογίες, οι περισσότερες από τις οποίες είναι υπέρ των φυτοφαρμάκων. Αυτές οι τροπολογίες προτείνουν να ε, διαγραφεί ένα μέρος του κειμένου και να ξαναγραφεί. Εγώ κατέθεσα μία μόνη τροπολογία που νομίζω ότι είναι ε, ιδιαίτερα επίγουσα και ε, είναι και κάτι πολύ σοβαρό. Πρόκειται για την τροποποίηση του κανονισμού για να διασφαλίσουμε την προστασία των ευπαθών ομάδων. Ο στόχος είναι, χωρίς χρονοτριβή, να ε, απαγορεύσουμε τη χρήση των φυτοφαρμάκων κοντά σε σχολεία, ε, σε παιδικές χαρές, σε νοσοκομεία ή σε μονάδες υγείας. Έχω λάβει την υποστήριξη των περισσότερων πολιτικών ομάδων, συνυπέγραψαν ε, την τροπολογία αυτή και επομένω βλέπουμε ότι είναι ισορροπημένη. Αν αυτή η σε μοναδες υγειας εχω λαβει την υποστηριξη των περισσοτερων πολιτικων ομαδων συνυπεγραψαν την τροπολογια αυτη και επομενως βλεπουμε οτι ειναι ισορροπημενη αν αυτη η τροπολογια το τροποποιούσε το κείμενο που ήδη είναι πάρα πάρα πολύ ε, μετριοπαθές, νομίζω ε, ότι θα είχαμε μία νίκη το λόμπι. Όμω, αν υιοθετηθούν οι τροπολογίε ε, που αφορούν την προστασία των ευπαθών ομάδων ε, και τη δημόσια υγεία, τότε οι βουλευτέ θα σημειώσουν μία νίκη. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λουαζό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η Επιτροπή ΠΕΣΤΑ δημιουργήθηκε μετά τα Monsanto Papers. Ο σκοπός δεν ήταν να γίνει δίκη, ούτε να απαλλάξει τα φυτοφάρμακα, αλλά να δει ποια ήταν τα κενά και οι στην διαδικασία την ευρωπαϊκή. Όπως βλέπουμε, βγήκε ένα ποντίκι από το βουνό και ε, η στεναρότητα, η πολιτική και οι λαοί αντικαταστάθηκαν και έχει σχετικά με το, έγινε, μιλάμε για το consensus και όχι για την ουσία. Εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε τους πάντες και κυρίως τους αδελφούς μας. Παρα, ε, εκτός εάν ανήκει στην Ευρώπη ε, των εθνών και των ελευθεριών. Και ε, έτσι επιδεινώνεται η κατάσταση και οι προτάσεις μας για την ε, επιθυμία των λαών που θέλουν περισσότερη εθνική ε, κυριαρχία, οι προσδοκίες αυτές γίνονται ε, θύματα ενός φανατισμού. Βεβαίως έχουμε οι φιλοευρωπαίοι είναι αφελείς όπως έλεγε, ε, ίσως να λυπούμαστε τους ανθρώπους που αγαπούν τα αποτελέσματα των οποίων αγνοούν τις αιτίε. Αυτό ισχύει για αυτήν την Επιτροπή. Οι περισσότεροι συνάδελφοι λένε ότι έχουμε μια διακυβέρνηση ε, ζωφερή, διαφανή ε, και έχουμε προσέγγιση με την μεγάλη βιομηχανία πολλοί θέλουν να ενισχύσουν τα μέσα της και την επιρροή της. Με άλλα λόγια, όταν στην Ευρώπη έχουμε προβλήματα, θα έπρεπε ε, να είμαστε όλοι ενωμένοι για να λύσουμε τα προβλήματα. Οι ευρωσκεπτικοί παντού, στην Γαλλία, στην Ιταλία, ε, στην Πολωνία, το Brexit, τα κίτρινα γυλαίκα στην Γαλλία, όλα αυτά τα σημάδια είναι ε, μιλούν από μόνα τους. Δεν θέλουν μια Ευρώπη που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Και αυτό ισχύει και για την έγκριση των ουσιών. Θα πρέπει τα κράτη να λαμβάνουν υπόψη τις εμπειρίες των ε, διαφόρων αγροτών για ένα σύστημα επαγρύπνησης που να είναι διαφανές και να συνάδει βεβαίως με την εμπορική πολιτική της Ευρώπης. Αν απαγορεύεται μια ουσία ε, στην Ευρώπη θα πρέπει να απαγορεύονται και προϊόντα που περιλαμβάνουν, περιέχουν αυτήν την ουσία. Νομίζω ότι το αστείο δίρκες αρκετά θα πρέπει ο οργανισμός να αναδιαμορφώσει πλήρως το σύστημα έγκρισης, πράγμα που εμείς προτείναμε με τροπολογίες τελείως αντίθετες με τα έγγραφα που βγαίνουν από αυτό, το θεσμό. Ευχαριστώ, κύριος Πέτερλε. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι συνεισηγητές ε, έκαναν ε, πολύ καλή δουλειά και θα πρέπει να τους ευχαριστήσουμε. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο. Στόχος ε, της ε, τελικής έκθεσης της Επιτροπής ΕΠΕΣΤ είναι να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στο να αυξηθεί η ποιότητα των τροφίμων. Θα πρέπει να σταματήσουν τα φυτοφάρμακα να δηλητηριάζουν και την πολιτική μας συζήτηση πριν, η περίοδος πριν τις εκλογές ε, σημαίνει ότι μπορεί να τίνουμε για κάποιες πρόσκαιρες ε, λύσεις ε, και φέτος δεν αποτελεί εξαίρεση η κατάσταση. Έτσι λοιπόν η έκθεση της ΠΕΣΤ που καλεί συστηματική αναθεώρηση όλων των μελετών σε σχέση με τον αντίκτυπο της γλυφοσάτης στο περιβάλλον και στην υγεία αποτελεί βάση για μελλοντική δράση. Όμως πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Διάφοροι οργανισμοί έχουν παρουσιάσει διάφορα αποτελέσματα σχετικά με ε, τους καρκινογόνες συνέπειες του γλυφοσάτ και άλλων φυτοφαρμάκων. Όμω, ε, ο χρόνο τρέχει. Η χρήση των ε, φυτοφαρμάκων στην παραγωγή των τροφίμων ε, είναι κάτι επιλογέ για τη βιοπικιλότητα, το έδαφο και το νερό. Δεν μιλάμε μόνο για την αποκατάσταση τη εμπιστοσύνη του κοινού, αλλά πρέπει να σε σεβαστούμε και τα πορίσματα της επιστήμης και να διασφαλίσουμε ότι ως πολιτικοί δεν δεχόμαστε πλέον συμβιβασμούς εις βάρος της υγείας. Ως ε, πρόεδρος της ομάδας για την καταπολέμηση του καρκίνου μπορώ να πω ότι ως ε, κοινωνία επικεντρωνόμαστε στο να βρούμε θεραπείες και συχνά ξεχνάμε την καταπολέμηση των αιτιών. Δεν είναι με ιδιωτική υπόθεση ο καρκίνο μεταξύ ασθενού και γιατρού, αλλά είναι και ένα κοινωνικό ζήτημα. Αν θέλουμε να πετύχουμε τις αλλαγέ, θα πρέπει να αλλάξουμε και το ευρωπαϊκό παράδειγμα και στην γεωργική πολιτική. Υπάρχουν εναλλακτικέ ε, των χημικών φυτοφαρμάκων, όμω λείπει η πολιτική βούληση για την τροποποίηση τη νομοθεσία. Νομίζω ότι η έκθεση τη Επιτροπή ΠΕΣΤ αποτελεί βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πότ. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τους εισηγητές και με όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί τους ε, για ένα χρόνο σε ό,τι αφορά την έκθεση μου αυτή. Άκουσα τι είπε ο Επιτροπός και την τελευταία χρόνο τα πορίσματα κατέδειξαν ότι τα συστήματά μας λειτουργούν, λειτουργούν καλά και διαπιστώνουμε παρόλα αυτά ότι δεν επαρκούν τα συστήματα αυτά για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του κόσμου. Και σήμερα λοιπόν έχουμε μπροστά μας ένα καλό, πολύ καλό κείμενο με καλές συστάσεις για τη βελτίωση του συστήματος χορήγησης έγκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενισχύσουμε και την εμπιστοσύνη των πολιτών στην διαδικασία λήψη αποφάσεων. Γι' αυτό λοιπόν προκαλεί μεγάλη έκπληξη και σοκ το γεγονό ότι προσπαθούν οι συνάδελφοι του ECR να καταστρέψουν αυτό το έργο. Θέλουν να διαγράψουν ολόκληρα αποσπάσματα για την καλύτερη προστασία των ε, παιδιών, τη υγεία των παιδιών. Θέλουν να μπλοκάρουν, να ληφθεί υπόψη ε, το κριτήριο της νευροτοξικότητας στην αξιολόγηση και άλλα στοιχεία τα οποία αποσκοπούν στην προστασία της υγείας. Μα αυτός είναι ο πότερος στόχος μας, ασφάλεια των τροφίμων και υγεία. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί οι συνάδελφοι του ECR θέλουν να το στερήσουν αυτό από τους Ευρωπαίους πολίτες και να πω ότι οποιαδήποτε νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τηρεί την αρχή της πρόληψης. Η αρχή λοιπόν αυτή τι επιτάσσει, ότι πάντα θα λειτουργούμε με τον πιο μετροεπαθή τρόπο όταν υπάρχει επιστημονική αμφιβολία για την υγεία του κόσμου. Αυτή λοιπόν η αρχή της πρόληψης είναι πάρα πολύ σημαντική. Για να δοθεί διαφάνεια στο σύστημα αντιδότησης και να βοηθήσουμε και τους γεωργούς μας στην τελική ανάλυση. Ελπίζω λοιπόν ο κόσμος να λάβει υπόψη αυτή την έκθεση και αυτό να καθορίσει και τις εκλογές. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκέρικ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ένα χρόνο περίπου έχει περάσει ε, από την έγκριση της γλυφοσάτης. Τότε κοιτάξαμε όχι μόνο τα τρόφιμα, αλλά και τη δυνατότητα επιβίωσης των καλλιεργητών και την έκθεση αυτή της Επιτροπής πέστε περιορισμένα μόνο μπορώ να την προσυπογράψω. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουμε επιστημονικά πορίσματα, αλλά επιρροή των λόμπιν σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την πρόταση για την ΕΦΣΑ. Καλή ιδέα, αλλά μόνο αν τελικά ο οργανισμός αυτή η αρχή έχει επαρκή σπόρους στη διάθεσή της. Και να κοιτάξουμε και την ευθύνη των κρατών μελών και των γεωργών, γιατί ο τοπικός παράγοντας ξέρει πώς παράγονται τα προϊόντα. Ας ε, δούμε πώς μπορούμε να δημορφώσουμε ένα οικολογικό μέλλον. Θέλω λοιπόν ε, να είναι υγιής ο κλάδος αυτός στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ, κύριος Χαουτέμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. ότι με επιτροπέ. Είναι η πολλωστή συζήτηση που κάνουμε για τα φυτοπροστατευτικά και ξέρω ότι πριν από τι εκλογέ θα έχουμε κι άλλε ακόμα. Αυτό που με ανησυχεί είναι το εξή. Κάθε φορά ξανά και ξανά αμφισβητούμε τα επιστημονικά δεδομένα και θα πρέπει να έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τις πιο αυστηρές διαδικασίες και τις πιο ασφαλείς διαδικασίες σε όλο τον κόσμο σε ό,τι αφορά το αλκοόλ, την καφεΐνη, τη βιταμίνη D. Δεν ε, επιτρέπονται σε πολλά μέσα. Και καταλαβαίνω πόσο έντονα συναισθήματα προκαλεί το θέμα αυτό της ασφάλεια των τροφίμων και φυσικά για την ασφάλειά μας πάντα θα πρέπει να φροντίζουμε. Αλλά αυτό που φοβάμαι είναι ότι πέρα, πέρα από τα επιστημονικά δεδομένα που αμφισβητούμε, καταπιάζουμε και τους γεωργούς. Ό,τι συστήματα και να χρησιμοποιούμε για την καλλιέργεια, κατα... παραμένουμε στη φύση. Υπάρχει αντίκτυπος περιβαλλοντικός. Να μην ξεχνάμε όμως ότι την τελευταία δεκαετία οι γεωργοί έχουν προσπαθήσει να μειώσουν τον αντίκτυπο αυτό και θέλουν να συνεχίσουν να επενδύουν προς την κατεύθυνση αυτή. Αν λοιπόν παράγουν, αν θέλουμε να παράγουν τρόφιμα, πρέπει να επιτρέπεται να χρησιμοποιούν κάποια προϊόντα, γιατί αυτά τα παίρνουμε από την φύση. Αν δεν χρησιμοποιούμε κανένα μέσο, θα χάσουμε τις οδιές μας και... Εδώ αυτό λοιπόν που θέλω να υποστηρίξω είναι να έχει τελικά ο Γεωργός επαρκή μέσα προκειμένου να ε, προστατεύει τις καλλιεργίες τους με τεχνολογικά μέσα αλλά και με οικολογικές ε, λύσεις, ε, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα φυσικά μέτρα για πιο, πιο πολύ σεβασμό προς το έδαφος. Gracias. Σας ευχαριστώ, κυρία Ριβαζή. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, κύριοι εισηγητές, βεβαίως αυτό το σκάνδαλο της Γλυσοβάτης έδειξε την ε, χειραγώγηση της οποίας όλοι είμαστε θύματα. Πόσοι οι μεγάλες επιχειρήσεις ε, ε, χρησιμοποίησαν την πιστήμη για το δικό τους όφελος. Το είδαμε στα Monsanto Papers και με την πράσινο και τους Σοσιαλιστές κατορθώσαμε να επιτύχουμε μια ειδική επιτροπή για τη διαδικασία έγκρισης των φυτοφαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χάρη σε αυτήν την επιτροπή μπορέσαμε να ανακαλύψουμε τα κενά και τις ελλείψεις του συστήματος. Ένα σύστημα πολύ περίπλοκο και που κατορθώνει πάντοτε να εγκρίνει τα φυτοφάρμακα στην αγορά. Είναι απίστευτο το ότι ξέρουμε ότι ο βιομήχανος διαλέγει ποιον θα μελετήσει την αίτηση, ε, πώς θα παρακάμψει τις μελέτες που δεν τον βολεύουν πώς αποφασίζει. Δεν είχαμε βεβαίως την έγκριση για να έχουμε τις μελέτες που οι βιομήχανοι είχαν ε, λόγω ε, της μυστικότητας, του απορρίτου των επιχειρήσεων. Και έχουμε αντίγραφα των αξιολογήσεων των μελετών που ε, τους ενδιαφέρουν. Βεβαίως, ορισμένες ουσίες εγκρίθηκαν, ενώ δεν έχουμε τις κανονιστικές ε, μελέτες και έχουν παρεκκλήσεις ε, οι εγκρίσεις προσωρινές που ανανεώνονται. Απίστευτο που τα φυτοφάρμακα στις χώρες δεν αξιολογούνται όπως οι ουσίες που είναι εγκεκριμένες σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Στις τα κράτη δεν γίνεται το ίδιο θα είναι σημαντικό οι συνάδελφοι να ψηφίσουν αυτήν την έκθεση. Θα έχουμε τις ευρωεκλογέ τον Μάιο. Θα πρέπει όλοι να υποστηρίξουμε, να υπερασπιστούμε την υγεία των πολιτών. Οι πολιτικοί πρέπει να αποφασίζουν τις εγκρίσεις και όχι οι πολυεθνικές. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό για το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Η κυρία Κόνετσνα. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ ήμουνα στην αρχή του εισθητίας ε, όταν ορίσαμε την ειδική αυτή επιτροπή και με πάρα πολύ καλά επιχειρήματα που, το, που είχαν προταχθεί τότε από τις ε, δεξιές πολιτικές ομάδες. Και συχνά εκνευρίστηκα γιατί αν ε, η Επιτροπή ακολουθούσε τις συστάσεις θα υπήρχε κανένα λόγος να λειτουργήσει αυτή η Επιτροπή. Το αποτέλεσμα θεωρώ ότι ανταποκρίνεται στις εργασίες μας. Έχουμε πολλές θετικέ ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια των ε, μελετών, ε, τη σύγκρουση συμφερόντων που την επιλύσαμε και κάποια άλλα θέματα πήγαν λίγο πιο πίσω, όπως η γλυφοσάτη και η βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων. Γενικά όμως οι εργασίες κινήθηκαν σε καλό κλίμα. Το γεγονός ότι τίθεται το θέμα των εμπειρογνωμόνων, θεωρώ ότι αποτελεί λιγότερο σημαντικό πλέγμα. Και θα ήθελα λοιπόν να σα ζητήσω να μην συνεχίσετε να αποδυναμώνετε εκθέσει στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ, ο κύριος Πιεντιτσίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτέλους, ε, αυτή η παγκόσμια μάχη κατά των φυτοφαρμάκων και των πραστοκτόνων ε, κατά μιας γεωργίας που να βασίζεται στη χημεία δίνει τα πρώτα αποτελέσματα και σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Αυτό είναι σημαντικό κατόπιν. Είναι ε, σημαντικό το αποτέλεσμα που πέτυχαν οι πολίτες γιατί υπήρξε αυξημένη συνειδητοποίηση απέναντι στους κινδύνους που θέτουν για την υγεία αυτές οι ουσίε Η έκθεση που ψηφίστηκε στην Επιτροπή ΠΕΣΤ είναι καλή. Εμεί όμως θεωρούμε ότι μπορεί και να βελτιωθεί. Δεν ανταποκρίνεται ακόμη στο αίτημα διαφάνειας ε, και διασφάλισης της υγεία που έρχεται από του πολίτε. Γι' αυτό παρουσιάσαμε τροπολογίε για να υπάρχει ε, άμεση ε, πάυση της ε, χρήσης τέτοιων ουσιών. Αυτές οι πρακτικές δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι θα εξελίψουν την χημεία. Οι τροπολογίες για την εξάλληψη των ουσιών που έχουν να κάνουν με ενδοκρινικούς διακταράκτες. Αυτές οι τροπολογίες λοιπόν που θεωρούνται νευροτοξικές και δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επέτρεψε εκ νέου την ε, έγκρισή τους. Όπως ξέρετε, είχαμε μία περίπτωση με τις μπανάνες. Ε, η πρώτη κίνηση ήταν ε, να απαγορευτεί η εισαγωγή. Δηλαδή ε, δεν έχει νόημα να κάνουμε όλη αυτή τη συζήτηση εδώ στην Ευρώπη όταν ε, κατόπιν επιτρέπουμε από το εξωτερικό να εισάγονται αγαθά που έχουν, όπου έχει χρησιμοποιηθεί γλυφοσάτ. Θα μπορούν να χρησιμοποιούνται αυτές ε, οι ουσίες ε, μόνο αν τα γνωρίζουν οι πολίτες. Ε, γι' αυτό πρέπει να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών εδώ. Ευχαριστώ όλους όσους έδωσαν αυτόν τον αγώνα, όλους τους συναδέλφους που έδρασαν προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπόγκοβιτς. Ευχαριστώ για το λόγο. Καταρχήν, θα ήθελα να συγχαρώ και τους δύο εισηγητές που προετοίμασαν μια πολύ ισορροπημένη έκθεση. Και πρόκειται για έναν ιδιαίτερα προβληματικό τομέα. Και το γλυφοσάτ ήταν ένα σημαντικό στοιχείο της συζήτησης. Η υγεία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και το επιβεβαίωσαν και οι πολίτες με την αίτησή τους. Και όταν ε, μιλάμε για την υγεία, χρησιμοποιούμε φάρμακα, αλλά όσο λιγότερα φάρμακα χρησιμοποιούμε, τόσο το καλύτερο. Το ίδιο ισχύει και για τη γεωργία. Πρέπει να προστατεύσουμε την υγεία των φυτών και μερικές φορές χρησιμοποιούμε φυτοφάρμακα. Όμως, ε, και για τη συμβατική και για τη βιολογική γεωργία είναι αληθές ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτά τα φυτοφάρμακα όσο το δυνατόν ε, λιγότερο. Εδώ μιλάμε για εξέλιξη και εγώ είμαι γεωργός, αλλάζει ο τομέας, ξέρω τι πρέπει να κάνουν ε, οι αγρότες και ξέρω ποιες αλλαγές έλαβαν χώρα τα τελευταία 30 χρόνια. Ε, χρησιμοποιούσαμε λιγότερα φυτοφάρμακα και τώρα είμαστε πιο διαφανεί σχετικά με τη χρήση τους. Αυτοί οι κανόνες θα πρέπει να ενδυναμωθούν Επίσης πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε επαρκείς ε, αρμοδιότητες σε επίπεδο ΕΦΣΑ προκειμένου να μπορεί να εφαρμόζει και να υλοποιεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους. Πρέπει να έχουμε και ένα περιθώριο για την καινοτομία, να χρησιμοποιήσουμε τη ρομποτική για να έχουμε μια πιο πράσινη ευρωπαϊκή γεωργία. Νομίζω ότι αυτός, αυτή πρέπει να είναι η οδός ε, που θα ακολουθήσει η νέα ΚΑΠ και θα υπερψηφίσω την έκθεση. Ο κύριος ε, Αντρία, παρακαλώ, για δύο λεπτά. να προστατεύσει κανείς την υγεία 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων, να προστατεύσουμε τα πλούτη μας. Αυτή είναι η ευθύνη μας και για τον λόγο αυτό η έκθεση την οποία έχουμε συντάξει ζητάει περισσότερη διαφάνεια, ανεξαρτησία από τους οργανισμούς μας ε, και αυστηρή εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης. Αυτή είναι η δομή της έκθεσης ως πρόεδρος αυτής της Επιτροπής. Θα ήθελα να συγχαρώ και ε, τους δύο συνεισηγητές που έκαναν εξαίρετη εργασία, αλλά πέραν αυτού θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο των μελών που εργάστηκαν κατά τη διάρκεια των εννέα μηνών της Επιτροπής. Όλοι δεν εργάστηκαν με την ίδια αποτελεσματικότητα και μερικοί έμειναν με την βεβαιότητα που είχαν στην αρχή, όπως είπε η κυρία Μακιντάερ και δεν θα άλλαζε τίποτα στην βεβαιότητά τη αν η Επιτροπή αυτή διαρκούσε κατά τη διάρκεια όλη τη θητεία και δεν θα διευρυνόταν η δημοκρατία. Έχουμε λοιπόν απαιτήσει από του συμπολίτε μας για την διαφάνεια και την ανθρώπινη υγεία. Μερικοί βιομήχανοι ε, προσπαθούν και παρεκτρέπουν ορισμένους βουλευτές. Ε, λένε ότι δεν είναι υπεράνω των νόμων. Ο Μονσάντο έχει βασίσει όλες ε, τις μελέτες σε αυτό και έχει κρύψει τις μελέτες στη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την διαδικασία από την ΕΦΣΑ και Νομίζω ότι οι προτάσεις που ψηφίσαμε πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει γίνει πολύ καλή εργασία. Θέλουμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Η Κομισιόν θα πρέπει να προτείνει μια ανακοίνωση και μια αναμόρφωση της νομοθεσίας για τα φυτοφαρμακευτικά προϊόντα, διότι από αυτό εξαρτάται η χρησιμότητα των εργασιών μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και των εργασιών σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Δημεσμάκρη. Για ένα λεπτό έχει το λόγο. Επίτροπε, συνάδελφοι, όταν ξεκίνησε η συζήτηση για τη γλυφοσάτη πριν από τρία χρόνια, επανάλαβα πολλές φορές το, τη σημασία της μεγαλύτερης διαφάνειας και της ανεξάρτητης έρευνα. έρευνας. Και αυτό είναι και το βασικό συμπέρασμα άλλωστε της ειδικής αυτής επιτροπής σε ό,τι αφορά τα αυτοφάρμακα. Και η πολιτική μου ομάδα υποστηρίζει, η αντιπροσωπεία μου υποστηρίζει αυτά τα συμπεράσματα. Η έγκριση τέτοιων μέσων θα πρέπει να γίνεται βάσει επιστημονικών στοιχείων και μάλιστα με αντικειμενικούς τρόπους, με διαφανή α, αντικειμενική διαδικασία. Όντω, έχουμε ένα από τα πιο αυστηρά συστήματα σε όλο τον κόσμο. Αλλά πάντα υπάρχει περιθώριο για βελτίωση και ακριβώ αυτή η βελτίωση χρειάζεται για να πετύχουμε πάλι την ε, εμπιστοσύνη του πολίτη και για να έχουμε και μεγαλύτερη προστασία της δημόσιας υγείας. Δύο κριτικά, επικριτικά στοιχεία ε, επιτρέψτε μου. Το θέμα της γλυφωσάτης, κατά πόσον είναι καρκινογόνα ή όχι. Αυτό μπορεί να απαντηθεί μόνο με συμπληρωματική έρευνα, όχι με πολιτικές επιτροπές. Και τέλος, ελπίζω αυτή η συζήτηση να ξεκινήσει μια... Αυτή η έκθεση να ξεκινήσει μια πιο ευρεία συζήτηση για την πιο βιώσιμη γεωργία. Ευχαριστώ κύριε Ντεμέσμακερ. Ο κύριος Ταραμπέλα θέλει να σας κάνει μια ερώτηση στα πλαίσια μιας μπλε κάρτας. Τη δέχεται ο κύριος Ταραμπέλα προφανώς και δέχομαι την ερώτηση του. Ο κύριος Ταραμπέλα. Σας άκουσα να λέτε ότι υποστηρίζετε τη σύσταση της Επιτροπής. Παρ' όλα αυτά είσαστε μέρος της πολιτικής ομάδας με την κυρία Μακιντάιρ. Για εξηγήστε μου λίγο πώς ε, εξηγείται το γεγονός ότι εσείς υποστηρίζετε τα συμπεράσματα της Επιτροπής ε, ενώ η κυρία Μακιντάιρ είναι αντίθετη. Για διευκρινίστε μου λίγο τι γίνεται. Ο κύριος Ντεμέμς Μάκερ για να απαντήσει. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Εγώ εδώ μιλώ και ψηφίζω εξ ονόματος της ε, αντιπροσωπείας και ακολουθώ το πρόγραμμα της δικής μου πολιτικής, του δικού μου πολιτικού κόμματος. Κύριε Χόισλινγκ, έχετε ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να πετύχουμε λοιπόν να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του πολίτη, γιατί χάσαμε πολύ από αυτή την εμπιστοσύνη σε ό,τι αφορά τη διαδικασία άδειας για αντιδότηση της γλυφωσάτης. Και φαίνεται λες και τα συμφέροντα της χημικής βιομηχανίας μας υπερισχύουν σε σχέση με το συμφέρον της δημόσιας υγείας. Αυτό θα πρέπει να το βελτιώσουμε λοιπόν. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε πιο ανεξάρτητες ε, γνωμοδοτήσεις. Χρειαζόμαστε επίσης ε, απόλυτη διαφάνεια. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό το βλέπουμε και στη νέα νομοθεσία για το τρόφιμα. Μπορεί να εφαρμοστεί η αρχή αυτή. Ρωτώ λοιπόν τους συντηρητικού και αυτό θα έχει ενδιαφέρον κατά πόσο και αυτοί υποστηρίζουν ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι το βασικό λοιπόν ζήτημα, απόλυτη διαφάνεια. Αλλά θα πρέπει να να προωθήσουμε και εναλλακτικέ για τη γεωργία. Πραγματικά δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται χημικά προϊόντα τα οποία θα πρέπει να παραμένουν πραγματικά ω εξαίρεση. Ευχαριστώ πολύ, πολύ ο κύριο Ομαζέ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, η έκθεση αυτή είναι τόσο σημαντική και κανείς πια δεν θα μπορεί να πει, δεν το ήξερα και όλοι γνωρίζουν σήμερα ότι εσείς φέρετε την ευθύνη για ένα από τα μεγαλύτερα υγειονομικά σκάνδαλα στην Ευρώπη, δηλαδή το σκανδάλου του γλυφοσάτα, γιατί ε, με πάση γνώση αποφασίστηκε να συνεχιστεί η δηλητηρίαση του κόσμου. Ναι, η Κομισιόν απέτυχε στην προστασία της υγείας των πολιτών και προτίμησε να προστατεύσει τα λόμπι και τις πολυεθνικές όπως η Μοσάντο και το λέω πολύ σοβαρά αυτό η σημερινή διαδικασία της ε, θέσης εμπορία ε, παρασιτοκτόνων ε, δεν είναι η Ευρώπη που προστατεύει, η Ευρώπη που ρηπαίνει και που σκοτώνει τη ζωή. Έτσι λοιπόν απευθύνω εκ νέου έκκληση σε εσά για να ακυρώσετε τώρα την έγκριση της θέσης σε αγορά αμφισβητούμενων φυτοφαρμάκων ξεκινώντας από το γλυφοσάτ και των φυτοφαρμάκων που σκοτώνουν τις μέλισσες. Η κυρία Εράνς Καρτσία για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Συζητάμε μέτρα για να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών και προστατεύεται η υγεία με την προστασία του περιβάλλοντος και των τροφίμων. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα χρησιμοποιούνται σωστά και έχουμε και το επιθυμητό αποτέλεσμα την υγεία και το περιβάλλον. Επίσης πρέπει να συνεισφέρουμε στο να μπορούν να συνεχίσουν να παράγονται οπορκυπευτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι εδώ νομίζω ότι όλοι μπορούμε Μπορούμε να συμφωνήσουμε όμω η επαγόρευση η χάρη τη απαγόρευση δεν είναι κάτι Πρέπει να λάβουμε τι αποφάσει μα βάσει επιστημονικών κριτηρίων τα θεσμικά μας όργανα με επικεφαλή στην ΕΦΣΑ μπορούν να προσφέρουν πληροφορίε και διαφάνεια και ασφάλεια ε, και βεβαιότητα στους Ευρωπαίου πολίτε. Έτσι λοιπόν α αφήσουμε του επιστήμονε να εργαστούν και εμεί ω πολιτικοί να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν τα μέσα για να συνεχιστούν οι εργασίε χωρί να πολιτικοποιούμε την επιστήμη γιατί δεν θα εξυπηρετήσουμε του πολίτε αν αντί για επιστημονικέ βεβαιότητε, του στέλνουμε ιδεολογικά ε, μηνύματα και αμφίσιμε απόψει όπω την περίπτωση του γλυφοσάτ. Αυτό θέλω να σας πω σήμερα. Σας ευχαριστώ για την εργασία σας και ευχαριστώ και τον κύριο Λίν. Θεωρώ ότι ήταν εξαντλητική δουλειά του και έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια για τη σύνταξη του γράφου αυτού. Σα ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, μετά τι διάφορε ακροάσει που είχαμε με την Επιτροπή ΠΕΣΤΑ, η διαδικασία έγκριση φυτοφαρμάκων πρέπει να βελτιωθεί στην Ένωση ε, πρέπει να δούμε ποιες είναι οι ελλείψεις και χαιρόμαθε που το κείμενο των δύο συνεισηγητών που συγχαίρω ε, μπορεί να βελτιωθεί ε, σε διάφορα σημεία έξι. Πρώτον, μια καλύτερη εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης, ανεξαρτησία στη διάρκεια όλης της διαδικασίας, ανάγκη να υπάρχουν πόροι αρκετοί για να ενισχύσουν την ανεξαρτησία. τέσσερων ανάγκη να βρεθούν εναλλακτικά προϊόντα ευνοώντας την καινοτομία. Πέντε, μια εποπτική ε, διαδικασία και έξι να προσθεθούν κριτήρια ανεξαρτησίας, ε, διαφάνειας, ε, κυρίως για το κράτος μέλος εισηγητής. Χαίρομαι που αυτή η ειδική επιτροπή έκανε συστάσεις που θα διευκολύνουν την ψηφοφορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Ναι, Βεβαίως, εγώ θα υποστηρίξω την άποψη της κυρίας Μακεντάερ για αυτό ε, το θέμα. Ε, νομίζω η άποψή μου είναι απλή. Η παραγωγή ε, δεν είναι μια αναγκαιότητα, δεν είναι πολυτέλεια και θα βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη εφαρμογή και να μειώνουν βεβαίως τις εκπομπές αερίων. Βεβαίως ε, θέλουμε να έχουμε καλούς κανόνες υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα τρόφιμα, να προστατεύουμε τη δημόσια υγεία. Συμφωνώ, η ασφάλεια και το, των τροφίμων και το περιβάλλον είναι νομίζω κάτι που πρέπει να βασίζεται σε αποδείξεις επιστημονικές. Συμφωνώ με τον Επίτροπο πώς θα διασφαλίσουμε ότι ε, ότι σε κάποιο σημείο πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη σε κάποιον. Θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη ε, σε αυτούς που βασίζονται στην επιστήμη. Δεν νομίζω ότι είναι ασφαλές 100% το σύστημα. Δεν έχουμε 100% ασφάλεια, αλλά πρέπει ε, να έχουμε εμπιστοσύνη σε κάποιον από επιστημονικής απόψεως. Η κυρία Ριμπέρο για έχω ξέρω ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα ε, το να ε, αναδείξουμε την επιστήμη έναντι των ψευδών ε, δεδομένων. Ε, στο ΕΛΚ εμείς δεν μπαίνουμε σε τέτοιες ε, λαϊκιστικές συμπεριφορές. Πάντοτε είμαστε στο πλευρό των πολιτών, υπερασπίζουμε τα δικαιώματά τους και στην αναζήτηση καλύτερων λύσεων και στην παροχή καλύτερων πληροφοριών. Το ίδιο ισχύει και σε σχέση με τη γεωργία. Πολλοί θέλουν να θεωρηθεί ως ένας υπεύθυνο τομέα για την λανθασμένη χρησιμοποίηση αυτών προϊόντων. Αυτό είναι εντελώς ψέμα. Ε, τα ε, φυτοπροστατευτικά προϊόντα χρησιμοποιούνται από πάρα πολλούς τομείς, όμως οι γεωργοί είναι αυτοί που κυρίως τα χρησιμοποιούν. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ ότι στο 27,2% ε, των χρήσεων στην Ευρώπη ήταν εντός της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ αυστηρή νομοθεσία νομοθεσία. Γι' αυτό οι πολίτε μπορούν να εμπιστεύονται τα θεσμικά του όργανα καθώ και τι ελεκτικέ αρχέ. Γι' αυτό ε, στο έγγραφο της Επιτροπής Γεωργίας το έχουμε αναδείξει αυτό. Εγώ χαιρετώ την αύξηση της χρηματοδότηση και για την ΕΦΣΑ και για τι αρχέ των κρατών μελών έτσι ώστε οι αρχέ αυτέ να μπορούν να υλοποιούν καλύτερα τη δουλειά του. Γι' αυτό είμαστε εδώ να εργαστούμε για να ε, μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους πολίτες να επαναφέρουν την εμπιστοσύνη τους στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Η κυρία Αγγιλέρα Γκαρσία για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ όλους τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή ΠΕΣΤ και ιδίως τους εισηγητές γιατί πιστεύω ότι τελικά το ψήφισμα που εγκρίθηκε από την Επιτροπή αποκαλεί μια πολύ καλή πρόταση. Θα ήθελα να δηλώσω την ξεκάθαρη υποστήριξή μου σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία που ενισχύει τη διαφάνεια, την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών, αύξηση της εμπιστοσύνης τους, ε, μείωση του διοικητικού άχθους, όπως και τη διασφάλιση της ε, ποιότητας ε, των επιστημονικών εκθέσεων, των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων. Ε, το να υποστηρίξουμε αυτές τις πρωτοβουλίες ήταν όλη η εργασία που έγινε. Όμως, καθώς η λήψη αποφάσεων σε σχέση με τη χρήση των προϊόντων αυτών έχει προβληθεί πολύ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παραγνωρίζοντας τα επιστημονικά στοιχεία Θεωρώ ότι θα πρέπει ε, να ξαναφέρουμε τη συζήτηση σε επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν, ακόμη και έτσι, εγώ νομίζω ότι είναι καλή συμφωνία και θα πρέπει όλοι να την εγκρίνουν κατά την ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σκούσμιουκ, για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Συζητάμε λοιπόν την έκθεση αυτή κάτω ιδείας πρωτοβουλίας. Μιλάμε για μια διαδικασία για την έγκριση φυτοπροστατευτικών. Και θα ήθελα να υποστηρίξω, να υπογραμμίσω στο σημείο αυτό, ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Δεκεμβρίου του 2017 οδήγησε σε, μια μεγάλη, σε ένα μεγάλο αίσθημα ανησυχίας στο κοινό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν δημιουργήθηκε η Επιτροπή ΠΕΣΤ. Αυτό αφορά και την απόφαση του δικαστηρίου του Αυγούστου 2018 στη ΣΥΠΑ για τις ε, επιζήμιες συνέπειες της χρήσης της γλυφωσάτης. 300 εκατομμύρια δολάρια καταβλήθηκαν ως αποζημίωση. Η ειδική λοιπόν αυτή η Επιτροπή ΠΕΣΤ ζήτησε μεγαλύτερη διαφάνεια. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά την απαγόρευση της αγλυφωσάτης σε κάποια ευαίσθητα σημεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Ντελαέ, έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η ή μη γλυφωσάτη. Αυτό περιμένουν οι πολίτες μας. Είναι απλό. Θέλουν να ασφαλιστεί η ασφάλειά τους, η υγεία τους με τα τρόφιμα και η συμμετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων. Η απάντηση είναι απλή. Επιστήμη. Ακούσαμε εμπειρογνώμονες, επαγγελματίε του τομέα και είμαι πεπισμένη ότι η επιστήμη πρέπει να είναι η βάση των αποφάσεών μας. Αυτό υποστηρίζω εδώ και τρία χρόνια σε αυτό το ημικύκλιο και χαίρομαι ότι η έκθεση καταλήγει στα ίδια συμπεράσματα. Θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη κατανόηση από τους πολίτες των διαδικασιών. Πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη απέναντι στους θεσμούς και στους οργανισμούς. Έχουμε στην Ευρώπη ένα από τα συστήματα τα πιο απαιτητικά, τα πιο αυστηρά στον κόσμο. Θέλουμε υψηλό επίπεδο απαιτήσεων για την ασφάλεια. Αυτό είναι απαραίτητο, αλλά όχι επαρκές η αγρότησα που είμαι, που εδώ και δέκα χρόνια μάχεται ε, για ε, προϊόντα φυτο-υγειονομικά μπορεί να σας το επιβεβαιώσει, να είμαστε απαιτητικοί, αλλά ενώ έχουμε ασφάλεια θα πρέπει να έχουμε τα μέσα, να υποστηρίζουμε την έρευνα, ας μην είμαστε αφελείς, να μην επιτρέπουμε στις επιχειρήσεις να κάνουν έρευνα να υποστηρίξουμε ε, τα, τα, τις επαγγελματίες. Θα πρέπει να έχουμε πρακτικές που να προστατεύουν το περιβάλλον. Όλες οι γεωργίες έχουν τη θέση τους και ανταποκρίνονται σε άλλες προσδοκίες. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους αγρότες απέναντι στην παγκόσμιο ανταγωνισμό. Ας μην εισάγουμε την γεωργία που δεν θέλουμε. Ε, θα είναι σαν να ρίχνουμε σφαίρα στον εαυτό μας. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή που έχουμε εδώ ανταποκρίνεται σε αυτούς τους στόχους και θα ήθελα να χαιρετήσω την εργασία των συνεισηγητών. Όλα δεν είναι τέλεια, ορισμένες από τις προτάσεις μας δεν λήφθηκαν πλήρως υπόψη, αλλά τα ουσιώδη βρίσκονται στην έκθεση. Και ελπίζω ότι θα έχουμε σύντομη απάντηση από την Κομισιόν στο τέλος αυτής της ψηφοφορίας, η οποία θα εγκρίνει με μεγάλη ε, πλειοψηφία. Ε, Σόλτεμος, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε και η συζήτηση γύρω από την γλυφοσάτη έχει λάβει μεγάλη έκταση τα τελευταία χρόνια και δικαίω, γιατί συζητήσαμε κατά πόσο η ουσία αυτή είναι επικίνδυνη, κατά πόσο χρησιμοποιείται σωστά και γι' αυτό λοιπόν όσα έγιναν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν σωστά. Δημιουργήθηκε μια ειδική επιτροπή για να εξετάσει κατά πόσο χρειάζεται μια καλύτερη διαδικασία, ένα καλύτερο σύστημα έγκριση τέτοιων φυτοφαρμάκων. Και μετά από ένα χρόνο σχεδόν εργασιών, η Επιτροπή κατέληξε σε μια σειρά πολύ καλών συστάσεων, απαραίτητων όλων τους. Και να σας πω ότι τρεις από αυτές είναι οι πιο σημαντικές κατά τη γνώμη μου. Καταρχάς, εστιαστήκαμε πιο πολύ στη διαφάνεια. Στην διαδικασία διαδότηση. θα πρέπει να γνωρίσουμε από πού προέρχεται η μελέτη, η εκάστοτε, ποιο την πλήρωσε και ποιο την ανέθεσε. Χρειαζόμαστε και πιο μεγάλη ανεξαρτησία στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΦΣΑ χρειάζεται πιο πολλά χρήματα για να μπορέσει να προωθήσει τέτοιε ανεξάρτητε έρευνε. Και όλα αυτά θα πρέπει να βασίζονται στην αρχή τη πρόληψη. Υποστηρίζω λοιπόν τα πορίσματα και θέλω λοιπόν να εγκριθούν για να γίνουν ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει ο πρόεδρο ο κ. Κέλλη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Και χαίρομαι. Και... Χαίρομαι που παίρνω το λόγο για αυτό το θέμα και που έχουμε μία συζήτηση σήμερα το απόγευμα στο Κοινοβούλιο. Καλωσορίζω το έργο αυτή της Επιτροπής και την ευκαιρία του κοινοβουλίου να εξετάσει το θέμα αυτό. Όπως ε, είπε νωρίτερα και η Κομισιόν, ε, είναι ένα θέμα που έχει ιδιαίτερη προσοχή ε, και λάβαμε όλοι πάρα πολλές ερωτήσεις και ανησυχίες από τους πολίτες για το θέμα αυτό. Εγώ προέρχομαι από την Νότια Πρόκειται για μια ιδιαίτερα αγροτική περιοχή. Καθημερινά συζητώ με αγρότε για το έργο του και τα φυτοφάρμακα, ιδίω το γλυφοσάτ. Ε, ήταν ε, μια κύρια ανησυχία τους. Κατανοούν το πρόβλημα οι γεωργοί, αλλά ταυτόχρονα ε, δεν έχουν εναλλακτικέ και αυτό τους προκαλεί ανησυχία. Είναι σημαντικό ε, να ε, διασφαλίσουμε την αξιοπιστία των επιστημονικών οργανισμών, γιατί χρειαζόμαστε ασφαλή πλαίσια και κανόνες. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στο σύστημα. Διαφορετικά θα μπορούσαμε να μην έχουμε και καμία διαδικασία έγκρισης αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ε, το σύστημα έγκρισης Ευρωπαϊκής Ένωση είναι από τα πιο ασφαλή στον κόσμο και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κρατάμε τα υψηλότερα πρότυπα για τους πολίτες, την υγεία, το περιβάλλον, αλλά και να προστατεύσουμε και την επιβίωση των ε, ε, γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ε, στην Ιρλανδία, παραδείγματος χάρη, οι Ιρλανδοί μπορούν να εφαρμόσουν ένα προϊόν φυτοπροστασίας πριν από τη σοδιά. Δεν έχουμε όμως τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες και μερικές φορές είναι απαραίτητο. Πρέπει να βρεθούν εναλλακτικέ για να θέτουμε καλύτερα προϊόντα στην αγορά και αν δεν υπάρξουν εναλλακτικέ, τότε αυτό θα ζημιώσει ε, πάρα πολύ ε, τις ε, θα σημειώσω πάρα πολύ τι αγροτικέ επιχειρήσει. Ε, ευχαριστώ και ζωή Ο κύριο Καπούτο, για ένα λεπτό. Η Ευρωπαϊκή Αρχή τη Προφύλαξη είναι σημαντική για την διατροφική ασφάλεια. Όμω τα τελευταία χρόνια η αξιοπιστία του συστήματο μα έγκριση για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα υποσκάπτηκε από αδιαφάνεια από την διαδικασία ε, νέα έγκριση ε, του γλυφοσάτ. Και μάλιστα εμφανίστηκαν και μεγαλύτερε ανησυχίε για την επικινδυνότητα του γλυφοσάτ και επιβεβαιώθηκαν και από δικαστικές αποφάσεις ε, που ε, αναγνωρίζουν ε, ότι μπορεί να είναι καρκινογόνος η ουσία. Οι ανησυχίες για τη σύγκρουση συμφερόντων μας δείχνουν το πόσο αναγκαία είναι, αναγκαίο είναι πλαίσιο για την εφαρμογή του. Η έκθεση της ΠΕΣΤ θέλει να θέσει στο επίκεντρο την υγεία των πολιτών, το περιβάλλον και τη διατροφική ασφάλεια, προσφέροντας δίνοντας στην ΕΦΣΑ απαραίτητους πόρους, ανεξαρτησία από τα λόμπι και επαρκείς αρμοδιότητες στη διαδικασία της έγκρισης. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να διορθώσουμε τα λάθη του παρελθόντος ε, και να βοηθήσουμε τη Γεωργία να υιοθετήσει βιώσιμες πρακτικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γκέρλινγκ. έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ναι. Είμαστε υπέρ αυτής της Ειδικής Επιτροπής. Δεν νομίζω ότι χρειαζόταν ένα ε, μέσο ε, για ε, το θέμα της γλυφοσάτης, διότι δεν μιλήσαμε για, για αυτό περισσότερο από οτιδήποτε άλλο θέμα σχετικά, σε σχέση με τα χημικά για την γεωργία. Βεβαίως είναι σημαντικό. Δεν θέλαμε ποτέ να μειώσουμε την σημασία των θεμάτων αυτών. Αλλά βεβαίως το σύστημα το ενωσιακό είναι το καλύτερο που υπάρχει και ε, δεν θέλουμε, ξέρουμε ότι η Κομισιό και ο Επίτροπός μας έχει στην πρόταση γενική για τα τρόφιμα μερικές προτάσεις που αναφέρονται στα θέματα τα οποία ανέφεραν πολλά μέλη αυτού του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι χρειάστηκαν πάρα πολλές προσπάθειες και ενέργεια από και συγχαίρω και ευχαριστώ ε, τους εισηγητές. Αλλά τι κερδίζουμε με αυτό. Διότι παράλληλα έχουμε μια ε, έκθεση ε, νομοθετική που είναι περίπου καλύπτει περίπου όλα τα θέματα που αναφέρθηκαν εδώ. Βεβαίως που είναι και καθήκον αυτού του Κοινοβουλίου βεβαίως. Δεν λέω ότι δεν είχαμε τροπολογίες που ήταν κάπως ιδεαλιστικές, αλλά νομίζω ότι καταλήξαμε σε συμβιβασμούς για τους οποίους είμαστε καλοί. Κυρίες και κύριοι, δεν θα ψηφίσω για αυτήν την έκθεση. Νομίζω ότι θα πρέπει προχωρήσει για ένα μνημείο που δείχνει πώς είμαστε καλοί στο να χάνουμε το χρόνο μας ε, και θα ήθελα να ασχοληθούμε με τον γενικό νόμο για τα τρόφιμα που είναι κάτι που νομοθετικά είναι πολύ πιο σημαντικό. Ο κύριος ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Με ικανοποίηση καταγράφω την αναγκαιότητα ε, στην έκθεση να ενισχυθεί η έρευνα και η καινοτομία για την προστασία των καλλιεργειών. Θα πρέπει να είναι η κύρια οδό μα ε, να βρούμε νέε τεχνικέ λύσει και μεθοδολογίε που να μα επιτρέπουν να μειώσουμε την χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και όταν είναι απαραίτητη η χρήση του ε, θα πρέπει να το κάνουμε με πιο αποτελεσματικό και συγκεκριμένο τρόπο. Έχοντα πάντα ω απόλυτε προτεραιότητε στην αρχή της πρόληψης και την προστασία της ανθρώπινης υγείας, της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος. Επίσης, πρέπει να εγγυθούμε ότι έχουν οι τα απαραίτητα εργαλεία στη διάθεσή τους για να προστατεύουν κατάλληλα την καλλιέργειά τους, προκειμένου να είναι βιώσιμη η αγροτική τους παραγωγή. Έτσι λοιπόν το σύστημα έγκρισης των προϊόντων αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς βασίζεται πάντοτε στα πιο ε, αυστηρά αποτελεσματικά κριτήρια πρέπει να είναι ένα ε, σύστημα ευέλικτο και ικανό να παρουσιάσει λύσεις ε, για να αντιμετωπίσει τις πολύ μεγάλες προκλήσεις που συναντάμε και στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές. Σας ευχαριστώ. Φτάνουμε τώρα στο Έχω τέσσερα αιτήματα και όλοι θα λάβετε το λόγο. Ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε η διασφάλιση υψηλού επίπεδου προστασίας της υγείας των ανθρώπων και των ζώων είναι βασικός στόχος της ευρωπαϊκής ένωσης. αυτό σημαίνει λήψη μέτρων και κυρίως εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης η οποία ως γνωστόν είναι θεμελιώδης αρχή της ευρωπαϊκής ένωσης και προβλέπεται στο άρθρο 191 συνθήκης λειτουργίας της ευρωπαϊκής ένωσης. επιπλέον πρέπει να υπάρξει διαφάνεια στη λήψη των μέτρων να γίνεται η μελέτη από ανεξάρτητη αρχή να μην παίρνονται αποφάσεις οι οποίες επί της ουσίας υπηρετούν την χημική βιομηχανία. άλλωστε είχαμε το σκάνδαλο με την γλυφοσάτη έχουμε απόφαση των πολιτών της ευρωπαϊκής ένωσης οι οποίοι έχουν κινηθεί με ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. όμως κύριε επίτροπε κύριε αντρουκάητης ήθελα να σας θέσω ένα σοβαρό θέμα. γίνονται εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από την τουρκία. αυτά τα προϊόντα καλλιεργούνται δυστυχώς με φυτοφάρμακα τα οποία απαγορεύονται επομένως τι θα γίνει με τις εισαγωγές των προϊόντων των τουρκικών αγροτικών προϊόντων που καλλιεργούνται στην τουρκία με φυτοφάρμακα που απαγορεύονται και παρά τα αυτά εισάγονται στην ευρωπαϊκή ένωση εισάγονται στην ελλάδα και είναι επικίνδυνα για την υγεία των πολιτών. σε αυτό το θέμα θέλω να πάρουμε μέτρα. ευχαριστώ. Ε, ε- Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε ξεκάθαρα ότι η έγκριση της γλυφωσάτης δεν είχε τι απαραίτητε εγγύησει και μεγάλη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου τα αναγνώρισε και αυτό χάρη στου πρασίνου. Η διαδικασία αναγνώριση και έγκριση της χρήση φυτοφαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ συχνά οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων. Πρέπει να αρχίσουμε να αξιολογούμε με ένα ανεξάρτητο και διαφανή τρόπο τις επιπτώσει των φυτοφαρμάκων στην υγεία μα και στο περιβάλλον. Ξεκινώντας βεβαίως με τη γλυφοσάτη. που σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας είναι καρκινογόνος. Να έχουμε αξιολογήσεις επιστημονικές και όχι απλώς τους ισολογισμούς εταιριών όπως η Μονσάντο. Χάρη στον αγώνα μας υπέρ της σωστής γεωργίας θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια Ευρώπη που βάζει πάνω απ' όλα την υγεία και το περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Φερέιρα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, η δημιουργία της ειδική Επιτροπής για την Αδειοδότηση Φυτοφαρμάκων έγινε λόγω της δημόσιας ανησυχίας σχετικά με την διαφάνεια και αυστηρότητα της διαδικασίας. Αυτό δεν έγινε από μόνο του. Είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι διάφοροι οργανισμοί πιέζονται από ε, δραστηριότητες λόμπι των φαρμακευτικών ε, και βιομηχανικών ε, ενώσεων. Και η αρχή της πρόληψης και της προφύλαξης δεν τηρούνται πάντα. Η δημόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος θα έπρεπε να υπερτερούν της βιομηχανίας και του βραχυπρόθεσμου κέρδους. Η ανάλυση κινδύνου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αιτιολόγηση παραβίασης της βασικής αυτής αρχής. Όσον αφορά την παρακολούθηση και τη μέτρηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, θα πρέπει να εξετάσουμε τι γίνεται όταν χρησιμοποιούνται ε, ε, ευρέως νέα προϊόντα. Ε, ναι το. Πιστεύω ότι η υγεία των πολιτών μας είναι ε, ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα που μας έχουν ανατεθεί και γι' αυτό η εκθέση αυτή είναι τόσο σημαντική. Ακριβώς διότι ζητάει μια διαφανή και ανεξάρτητη αξιολόγηση των φυτοφαρμάκων. Αρκεί να θυμηθούμε ολόκληρη την ιστορία της γλυφοσάτης που δημιούργησε τόσες πολλές συζητήσεις για τις ε, ε, επιβλαβείς επιπτώσεις ε, της γλυφοσάτης. Και οι μελέτες ήταν αμφιβόλου ποιότητας. Ήταν μελέτες που είχαν γίνει κατ' εντολή της επιχειρήσης που παρήγε τη γλυφοσάτη. Χρειαζόμαστε ανεξάρτητες και αντικειμενικές αξιολογήσεις και επίσης πρέπει να δίδεται πρόσβαση στο κοινό στις επιστημονικές μελέτες. Και για να μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα είναι ανεξάρτητες οι μελέτες, θα πρέπει να υπάρχει και μία εποπτεία επί των μελετών, για να μπορέσουμε να έχουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ένα λεπτό. Merci. Ε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα ορισμένου συναδέλφους που είπαν ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλειας των Τροφίμων είναι αποτελεσματικό και ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στις αρχές φυτοπροστασίας. Αλλά με βάση την αρχή της προφύλαξης πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα που είχαμε παραδείγματος χάρη στις Γαλλικές Αντίλες γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλα τα προβλήματα του πληθυσμού. Αυξήθηκε πάρα πολύ ο καρκίνος του προστάτη. Βλέπουμε ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου το 80% του πληθυσμού έχει πληγεί. Ναι, να ενισχυθεί η διαφάνεια, αλλά στο όνομα της αρχής της προφύλαξης θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ούτως ώστε όλοι οι πολίτες μας να είναι καλύτερα προστατευμένοι. Και ο κ. Σαντριό και εγώ ζητήσαμε να μειωθούν ε, ε, τα όρια ε, LMR, αλλά μέχρι τώρα δεν μας έχει δοθεί απάντηση και περιμένουμε από εσά ότι θα καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να έχουμε καλύτερη εγγύηση για την υγεία του πληθυσμού μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία Eye. Θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο. Παρακαλώ κύριε Πίτροπε. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητά μέλη, άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά τα οποία είπατε. Σας ευχαριστώ για αυτά. Θα μου επιτρέψετε να αντιδράσω για ορισμένες από τις παρεμβάσεις αυτές. Η κυρία Ρίση. να πω ότι γίνονται προσπάθειες και σε επίπεδο καταλόγου και σε επίπεδο κριτηρίων. Το Δεκέμβριο είχαμε επίσης ε, συζητήσει τα θέματα έλλειψης συμβατότητας τα οποία ε, είχαν τεθεί από πλευρά των κρατών ε, μελών όπως επίσης και τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες. κανονικά θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι όροι και για τα εισαγόμενα και για τα τοπικά παραγόμενα προϊόντα. Όταν υπάρχει ένα προϊόν το οποίο δεν παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να ζητηθεί μια, ένα ποσοστό ανοχής για προϊόντα τα οποία εισάγονται και μπορεί να εγκριθεί εφόσον επιβεβαιωθεί από την ΕΦΣΑ. και για τα υπόλοιπα προϊόντα προσπαθούμε να διασφαλίσουμε το υψηλό επίπεδο παραγωγής στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι προσπαθούμε να ρυθμίσουμε λοιπόν τα εισαγόμενα προϊόντα. Τώρα το να με κατηγορείτε γιατί δηλητηριάζω τους πολίτες είναι λίγο περίεργο. Ε, το, βασικό μήνυμα που μου άφησε ο πατέρας μου είναι να μην λέω ψέματα και το ίδιο κάνω και στις εκλογές. Είναι ένα απλό μήνυμα για τις εκλογές. Πρέπει να λέμε την αλήθεια και θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην επιστήμη και εφόσον έχουμε εμπιστοσύνη στην επιστήμη τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Ήταν μια καλή ευκαιρία λοιπόν να ακούσω τις προτάσεις σας, τα συμπεράσματά σας. Δείξατε ότι λαμβάνετε πολύ σοβαρά υπόψη αυτές τις προτάσεις. Εγώ στο τέλος του εξαμήνου θα σας παρουσιάσω μια αρχική πρόταση έτσι ώστε να προστατεύσουμε τους πολίτες, να προστατεύσουμε την υγεία της, ε, των ε, ζώων όπως επίσης και την υγεία του φυτικού κεφαλαίου. Νομίζω ότι τα πράγματα τα κάνουμε σωστά. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα ακούσουμε τώρα τα συμπεράσματα των δύο εισηγητών. Ε, κύριε Λίνς, έχετε δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είδαμε πόσο φορτισμένη ήταν η συζήτηση, και αυτό δείχνει ότι έχουμε πολύ διαφορετικές απόψεις πάνω στο θέμα αυτό. Ωστόσο, αποτελεί επιτυχία το ότι καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια συνενετική έκθεση, ξεπερνώντας ε, τα όρια των ε, πολιτικών ομάδων και των ιδεολογιών μας. Έτσι λοιπόν ε, έχουμε μία προσέγγιση που βασίζεται στην επιστήμη, κάτι που χρειαζόμαστε διαδικασία αυτή. Τονίζω ότι τα συναισθήματα εδώ δεν έχουν ε, καμιά δουλειά. Ε, θα ήθελα να απαντήσω στους συναδέλφους, αλλά μερικοί από αυτούς έχουν ήδη αποχωρήσει. Στον ε, συνάδελφο Βάιτς θα ήθελα ε, να πω επειδή θεωρεί ότι όλα τα φυτοφάρμακα είναι υπερβολικά επικίνδυνα. Από την άλλη, ε, αποσιωπά ότι ο χαλκός είναι ε, το χειρότερο δηλητήριο για το έδαφος. Ε, ή να απαντήσω στον συνάδελφο Χάζεκαμπ ή την συνάδελφο Ρίβαζη που μιλάει ακόμη για σκάνδαλο ενώ η έκθεση αυτή καταλήγει ακριβώς στο αντίθετο συμπέρασμα. Ε, θα ήθελα να σταματήσουμε ε, να στρέφουμε την, τη γεωργία κατά του περιβάλλοντος. Μαζί πάνε αυτά τα δύο. Θέλουμε αποτελεσματική παραγωγή, βιώσιμα προϊόντα εντός των πολιτικών πλαισίων που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο, μια αξιόπιστη διαδικασία αδειοδότησης και νομίζω ότι με τις συστάσεις μας μπορούμε να βελτιώσουμε τη διαδικασία αυτή και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει τις προτάσεις μας. Σας ευχαριστώ κύριε εισηγητά, ο κύριος Στάς, ο επόμενος εισηγητής. Ένα λεπτό έχει στη διάθεσή του. Eh, ευχαριστώ πρόεδρε. Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνεισηγητή μου όπως επίσης και τον πρόεδρο Αντριού για την πολύ σημαντική προσπάθεια την οποία επιτελέσαμε από κοινό. Η έκθεση αυτή δείχνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακούει τους πολίτες του εναντίον της πόλωσης, εναντίον του λαϊκισμού. Και παρά τις διαφορετικές αντιλήψεις που έχουμε για την παραγωγή οπόρων, όπως επίσης και ε, για την γεωργία μπορούμε να λειτουργήσουμε ζητώντας όλοι υπέρ μια αντικειμενική και ελεύθερη και αξιόπιστη διαδικασία διοδότησης. Αυτό έχει σημασία. Δεν έχει σημασία οι πολιτικοί να κραυγάζουν, θέλουν οι πολίτες οι πολιτικοί να συνεργάζονται διακομματικά και να βρίσκουν τις σωστές λύσεις. Η ασφάλεια των πολιτών και η ασφάλεια των ζώων είναι αυτό το οποίο μετράει. Συνεπώς εξυπηρετούμε το γενικό συμφέρον και όχι το ιδιωτικό και επιμέρους συμφέρον. Ευχαριστούμε κύριε Σίγητα. Κλείνει η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει την Τετάρτη. Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης έκθεση της κυρίας Μοτέρα Ντεαγκιγιάρ για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Κυρία Συγητρία, τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε ε, Μπούλτς, θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ το Συμβούλιο για την ανάληψη της Προεδρίας και ελπίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορέσει να επιληθεί κατά τη Ρουμανική Προεδρία. Η πρόταση την οποία θα ψηφίσουμε αύριο για την χρησιμοποίηση οχημάτων χωρίς οδηγούς, ε, για τη μίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγούς ε, στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Είναι κομμάτι του, της πρώτης δέσμης ε, μέτρων για τις μεταφορές και προσπαθεί να ε, αντικαταστήσει μια οδηγία η οποία ισχύει εδώ και 25 χρόνια. Θέλουμε να προσαρμοστούμε στις ανάγκες των εμπορευομένων και του κλάδου με βάση τις αλλαγές που έχουν γίνει μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια. Αυτό το οποίο προτείνουμε είναι τα κράτη-μέλη να μην περιορίζουν τη χρήση μισθωμένων οχημάτων από εταιρεία η οποία είναι εγκαταστημένη σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον βεβαίως ε, συμμορφούνται προς τις απαιτήσει ασφαλείας. Αυτό μας οδηγεί στην αγορά ε, μίσθωσης και χρηματοδοτική μίσθωσης οχημάτων. Μια αγορά που είναι ιδιαίτερα κοντά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θέλουμε να αποφύγουμε στρεβλώσεις της αγοράς ε, λόγω των διαφορετικών φορολογικών συντελεστών σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Γι' αυτό δίνουμε στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να περιορίσουν τη χρήση μισθωμένων οχημάτων στην επικράτειά τους είτε χρονικά είτε ως ε, αριθμό οχημάτων τα οποία μπορεί να μισθώσει μια εταιρεία. Τέσσερις συνεχείς μήνες χρήσης ενός μισθωμένου οχήματος σε ένα κρατος μέλος ή 25% του συνολικού στόλου οχημάτων ενός ε, ιδιοκτήτη, μιας εταιρείας. Και αν μια εταιρεία έχει μέχρι τέσσερα οχήματα, έχει λιγότερο από τέσσερα οχήματα, ε, θα μπορεί να χρησιμοποιεί τουλάχιστον ένα όχημα μισθωμένο σε άλλη χώρα. Θα πρέπει να υπάρχουν βέβαια ηλεκτρονικά μητρώα καταγραφής οχημάτων και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών μέσω του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών της ε, ενίας αγοράς όπως προτείνεται και για υπόλοιπα τμήματα της δέσμης ε, μέτρων για την κινητικότητα. Έτσι θα φτάσουμε στην ενιαία αγορά στον τομέα αυτό με ένα ήπιο τρόπο, τηρώντας ε, και τους ε, κανόνες της αγοράς και τους κοινωνικούς κανόνες. Ζητώ λοιπόν από όλους τους συναδέλφους, κυρία Πρόεδρε, να μην ψηφίσουν τροπολογίες οι οποίες προσπαθούν να επιφέρουν διακριτική μεταχείριση μεταξύ μισθωμένων οχημάτων και οχημάτων τα οποία λειτουργεί μια εταιρεία για λογαριασμό της. Δεν θα πρέπει να υπονομεύσουμε τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών. Επομένως, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, πείτε όχι ε, στις προσπάθειες ε, να μπλοκαριστεί ένας ενιαίος πράσινος χώρος οχημάτων. Ε, μην ψηφίσετε λοιπόν τροπολογίες που θα δυσκολεύσουν ε, τις εταιρείε να ε, ενοικιάζουν οχήματα γιατί τελικά η επιβάρυνση θα είναι επιβάρυνση εις βάρος των εργαζομένων. Εδώ έχουμε μια οδηγία η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών ζωής όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Βεβαίως τα οχήματα θα πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές όσον αφορά τις εκπομπές και δεν θέλουμε να έχουμε επικαλύψεις. Επομένως, παρακαλώ, μην ψηφίσετε τις τροπολογίες που θα προσπαθήσουν να τροποποιήσουν την νομοθεσία προς ε, λάθος κατεύθυνση. Παρακαλώ να ψηφίσετε αύριο υπέρ της έκθεσης αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία εισηγήτρια, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα δίνω το λόγο στην Επιτροπή, στην Επίτροπο κυρία Μπούλτς. Έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Τραν και ιδιαίτερα την κυρία Μοντέιρο και τους σκιώδει εισηγητές για την γενικά ισορροπημένη και καλογραμμένη αυτή έκθεση πάνω στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, επικαιροποίηση της πρόταση της Επιτροπής για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων. Και ε, τα μισθωμένα αυτά οχήματα χωρίς οδηγό αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των οικονομικών φορέων και αποτελούν εναλλακτική λύση σε σχέση με ακριβά οχήματα τα οποία πιθανότατα να μην χρησιμοποιούνται επαρκώς. Τα μισθωμένα οχήματα γενικά είναι ε, καινούρια, πιο καθαρά από τα ε, οχήματα που βρίσκονται στην ιδιοκτησία του οικονομικού φορέα. Συνήθως τα μισθωμένα οχήματα πληρούν τα τελευταία ε, περιβαλλοντικά πρότυπα και έτσι είναι καλά και για την ασφάλεια στους δρόμους και για το περιβάλλον. Η αναθεώρηση των κανόνων σχετικά με ε, την χρησιμοποίηση μισθωμένων ε, οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές θα οδηγήσουν σε εξυγχρονισμό του στόλου και πιο καθαρά οχήματα. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν οχήματα που έχουν μισθώσει εκτός ε, της ε, χώρας εγκατάστασής τους και θα πρέπει να ε, έχουν ασφάλεια δικαίου στην περίπτωση αυτή. Όταν μισθώνει κανείς ένα όχημα θα πρέπει να μπορεί να το χρησιμοποιήσει οπουδήποτε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην επιβάλλονται διάφοροι περιορισμοί ανάλογα με το που εργάζεται κανείς. Για να αποφύγουμε ανεπιθύμητες συνέπειες μπορεί να περιοριστεί η χρήση των μισθωμένων οχημάτων σε κάποιο βαθμό, αλλά θα πρέπει να επιτρέπεται καταρχάς στους οικονομικούς φορείς να μπορούν να καλύψουν εποχικές ανάγκες ή να ε, αντικαθιστούν ε, ε, οχήματα δικά τους που έχουν πάθει βλάβη. Αυτά είναι παραδείγματα όπου οι έρευνε μα έδειξαν ότι η δυνατότητα να χρησιμοποιεί κανεί οχήματα μισθωμένα στο εξωτερικό ε, είναι πιο αναγκαία. Η έκθεση τη κυρία Μοντέιρο ε, πολύ σωστά λέει ότι ε, μεταφέροντας ε, την ε, χρήση αυτών των οχημάτων από το άρθρο 2 στο άρθρο 3 της οδηγίας, αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη δεν θα μπορούν να περιορίσουν την χρήση μισθωμένου οχήματος στο έδαφος τους, εφόσον επιτρέπεται στο έδαφος του κράτους μέλους όπου έχει από το οποίο προέρχεται το όχημα. Δηλαδή, αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μισθωμένο όχημα στη χώρα σα, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ε, σε οποιαδήποτε χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι, τροπο... Οι τροπολογίε ε, που έχουν υποβληθεί ε, για την αυριανή ψηφοφορία γενικά μπορούν να γίνουν αποδεκτέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, θα ήθελα να αναφέρω ιδιαίτερα δύο τροπολογίε που μπορούν να καταστρέψουν την λεπτή ισορροπία που έχει πετύχει η κυρία Μοντέιρο. Μία τροπολογία επιτρέπει στα κράτη-μέλη να περιορίσουν τη χρήση μισθωμένων οχημάτων ξένου οικονομικού φορέα εφόσον δεν πληρεί τα τελευταία περιβαλλοντικά πρότυπα. Ένα επιχείρημα υπέρ τη χρήση των οχημάτων αυτών είναι ότι είναι νεότερα και πιο καθαρά από άλλα οχήματα. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι πρόβλημα. Μια τέτοια ε, ρήτρα όμως ε, θα καταστρέψει την ισορροπία της έκθεσης τη κυρία Μοντέιρο, διότι έτσι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να επιβάλλουν διαφορετικούς περιορισμούς ε, στα μισθωμένα οχήματα. Δηλαδή θα πρέπει πρώτα να ελέγξει κανείς αν μπορεί να χρησιμοποιήσει το όχημα το μισθωμένο στην ε, χώρα όπου προτίθεται να το χρησιμοποιήσει. Ενώ δεν θα επιβάλλεται καν, κανένα τέτοιο περιορισμό ε, στα ιδιόκτητα οχήματα. Άλλη τροπολογία που οδηγεί σε ανησυχίε ε, είναι ο περιορισμό μισθωμένων οχημάτων ε, για ιδιωτική χρήση. Κάποιοι σε χώρες όπου εφαρμόζονται τέτοιοι περιορισμοί έχουμε πιο πολλές διαδρομές χωρίς φορτίο. Και επίση δεν θα έχουμε ασφάλεια δικαίου για τι επιχειρήσει που χρησιμοποιούν μισθωμένα οχήματα. Τούτων λεχθέντων μπορούμε να δεχτούμε όλε τι υπόλοιπε τροπολογίε που αυξάνουν τι πληροφορίε που παρέχονται στου ε, οδηγού και ενισχύουν την συμμόρφωση με την οδηγία και την υποβολή τη οδηγία. Σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Φτάνουμε στι πολιτικέ ομάδε. SND, η κυρία ε, Γκρίφιν, έχετε δύο λεπτά, παρακαλώ. Τα ενοικιαζόμενα οχήματα είναι ένα βασικό ε, κομμάτι της ε, δραστηριότητας μεταφορών. Η Ολομέλεια αυτή έχει ήδη πάρει μία απόφαση για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα ενοικιαζόμενα. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα η αλλαγή αυτή νομοθετική στα πλαίσια της αμφισβητούμενης γενικότερα πολιτικής για τις μετακινήσεις. Η σοσιαλιστική ομάδα έχει καταθέσει ορισμένες σημαντικές τροπολογίες που υποστηρίζονται από πολλούς βουλευτές και από άλλες πολιτικές ομάδες παρά επανειλημμένες προσπάθειες έβρεσης συμβιβαστικών λύσεων σχετικά με την εκπαίδευση των οδηγών, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την απελευθέρωση της αγοράς και των συνθήκων εργασίας, ο εισηγητής ή η εισηγήτρια μάλλον δεν δέχτηκε τις προτάσεις αυτές και έτσι το κείμενο δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρό. Θα πρέπει να υποστηρίξετε λοιπόν αύριο τις τροπολογίες μας έτσι ώστε να ξεκινήσουμε σε σωστή βάση τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Τα ενοικιαζόμενα θα πρέπει να είναι συμβατά με τα επίπεδα εκπομπών τα οποία προβλέπουν οι κοινοτικοί κανόνες. Όταν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη, θα πρέπει το κράτος υποδοχής να αποφασίζει αν θα μπορεί να αποδεχθεί την λειτουργία στο έδαφος τους ενός ενοικιαζομένου επαγγελματικού οχήματος. Θα πρέπει να υπάρχουν επίσης οι απαιτούμενες πληροφορίες, θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις κατάλληλες σε περίπτωση παράβασης της οδηγίας και νομίζω ότι όταν παραβιάζεται η νομοθεσία θα πρέπει να θεωρείται σαν κάτι το σοβαρό και θα πρέπει να, λαμβάνεται, να αναλαμβάνεται δράση εις βάρος των παρανομούντων. Συνεπώς λοιπόν η σοσιαλιστική ομάδα ως έχει το κείμενο δεν μπορεί αν δεν το απολογηθεί να το στηρίξει. Ευχαριστούμε. Μάκες εκ μέρους του ECR. Ευχαριστώ. Εδώ προσπαθούμε να βρούμε μια λεπτή ισορροπία μεταξύ αφενός μεν του να ανοίξει η αγορά για τα μισθωμένα εμπορευματικά οχήματα που θα έχει και θετική επίδραση στην αγορά και από την άλλη πλευρά ε, το να αποφύγουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό ε, για λόγους ασφάλειας και για λόγους ε, δημοσιονομικής αυτονομίας. Και νομίζω ότι η συγγήτρια κατάφερε να επιτύχει την ισορροπία αυτή. Για τη ρύθμιση της εσωτερικής αγοράς υπάρχουν κάποιοι όροι και παράλληλα τα κράτη-μέλη μπορούν να ρυθμίζουν το τι θα ισχύει για τις επιχειρήσεις χωρίς ε, να στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά. Η πρόταση αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί σωστά όταν θα έχει επιτευχθεί συμφωνία με το Συμβούλιο. Και στη συνέχεια, μετά την συμφωνία από το Συμβούλιο, θα πρέπει η επιβολή της νομοθεσίας να γίνει σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Μίλτενμπουργκ, δύο λεπτά, εκ μέρους των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η χρήση μισθωμένων οχημάτων έχει πολλά πλεονεκτήματα στις οδικές εμπορευματικέ μεταφορές. Μπορεί έτσι να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ευελιξία των ε, επιχειρήσεων. Επιπλέον, με τη χρήση μισθωμένων οχημάτων, αποφεύγουμε την σπατάλη κεφαλαίου, διότι ε, χρησιμοποιούνται στο έπακρο τα οχήματα. Επίση, ε, τα μισθωμένα οχήματα γενικά είναι πιο καινούρια, πιο φιλικά προς το περιβάλλον, πιο καθαρά. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι σημαντικό βήμα στην απελευθέρωση της ευρωπαϊκής αγοράς για τα μισθωμένα οχήματα. Μπορούμε έτσι να έχουμε συνθήκες ίσου ανταγωνισμού ανάμεσα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Επίσης μπορούμε έτσι να εξαλείψουμε περιτά εμπόδια θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαραίτητη η σωστή καταχώρηση των μισθωμένων οχημάτων ε, για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τους ε, κανόνες για τις ενδομεταφορές. Επίσης, θα πρέπει να βελτιωθεί η επικοινωνία ανάμεσα στις αρχές ε, των κρατών μελών, ώστε να είναι πάντα σαφές ποια είναι η χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα. Στο κείμενο που θα ψηφίσουμε αύριο έχουμε πολύ καλές διατάξεις και το ίδιο ισχύει για τη χρήση οχημάτων από άλλα κράτη-μέλη καθώς και την ε, δυνατότητα κρατών μελών να περιορίζουν τη χρήση των οχημάτων. Έτσι θα αποφύγουμε την μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε χώρες με πιο ευνοϊκούς κανόνες. Πρόκειται για ένα ισορροπημένο κείμενο το οποίο θα μας οδηγήσει σε μια σωστή εσωτερική αγορά μισθωμένων οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στηρίζω λοιπόν το κείμενο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Στο όνομα των Πρασίνων, ο κύριος Νταλούντε, έχετε ένα λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το... Οι δέσμοι μέτρων για τις μεταφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι αξιέπαινοι. Λόγω όμως ε, υπερβολικού εστιασμού στις οδικές μεταφορές ε, χάνουμε την ευκαιρία να πετύχουμε τον απαραίτητο μετασχηματισμό στον τομέα των μεταφορών. Στη συζήτηση για τα μισθωμένα οχήματα θα θέλαμε να εστιάσουμε περισσότερο στον σωστό έλεγχο και στα τέλη για να έχουμε δίκαιο φορολογικό ανταγωνισμό. Θα έπρεπε να εστιάσουμε επίσης περισσότερο στον πράσινο προσανατολισμό, την, ε, ε, ε, να τονίσουμε περισσότερο τις σιδηροδρομικές μεταφορές σε σχέση με τις οδικές και καλύτερη εκπαίδευση για τους οδηγούς των φορτηγών. Θα θέλαμε πιο αυστηρούς ε, κανόνες, για παράδειγμα, για τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις ε, και πιο αυστηρούς φορολογικούς κανόνες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Στο όνομα της GUE NGL, η κυρία Βίο, έχετε ένα μισή λεπτό. Merci. Ευχαριστώ το ότι ανοίγει η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ενοικιάζουν οχήματα για μεταφορά εμπορευμάτων θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις ε, να αντιμετωπίσουν τις διαφορές που μπορεί να υπάρχουν εποχιακά στη δραστηριότητά τους. Αυτό όμως δείχνει ε, κάτι, ότι υπάρχει ένα κενό ρυθμιστικό το οποίο δημιουργεί πάρα πολλά περιθώρια για καταχρηστική ε, αντιμετώπιση. Εγώ σαν παράδειγμα μπορώ να προτείνω την μείωση του χρόνου διάρκειας της μίσθωσης όπως επίσης και στην συγκεκριμένη οριοθέτηση του ποσοστού του συνόλου των οχημάτων. Νομίζω όμως ότι δεν έχουμε τις εγγυήσεις οι οποίες απαιτούνται. Το να επιτρέψουμε την ενοικίαση χωρίς όρια και να επαναλαμβάνουν ανατετράμινο τις μισθώσεις, αυτό θα οδηγήσει σε καταχρήσεις. Καταχρήσεις και φορολογικές και ε, επανειλημμένες ε, δράσεις επιχειρηματικές που οδηγούν σε απώλεια φορολογικών εσόδων, εκμετάλλευση ε, των εργαζομένων και παραβίαση των όρων εργασία τους, όπως επίσης ενίσχυση του κοινωνικού dumping και παραβίαση των περιβαλλοντικών ρυθμίσεων. Εγώ φυσικά δεν μπορώ να κάνω δεκτή την πρόταση αυτή. Η κυρία Γιούτο για ένα λεπτό, FDD. Επίτροπε, συνάδελφοι, βλέπουμε ότι η χρήση ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς οδηγό είναι μια λύση που δίδει εγγυήσεις σε κάποιες μεταφορικές επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούνται πιο πρόσφατα οχήματα με μικρότερα επίπεδα ανασφάλειας, αλλά αυτό δημιουργεί και κάποια προβλήματα σε σχέση με τον σεβασμό του ανταγωνισμού ανάμεσα σε επιχειρήσεις διαφορετικών χωρών και προβλήματα επίσης σε σχέση με τον σεβασμό των συνθήκων εργασίας. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε την μαζική χρήση των οχημάτων ανεφοδηγού ιδιαίτερα σε σχέση με τα άνω των 6 τόνων οχήματα ιδία χρήση. Ευχαριστούμε. Εκ μέρους των πολιτικών ομάδων ακούσαμε τους ομιλητές και περνάμε στους υπόλοιπους ομιλητές. Κύριε Ντεμόντε, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Είμαι υπέρ του να γίνει ένα επιπλέον βήμα για την κατάργηση των εμποδίων της σωστής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της δημιουργίας ενός ενιαίου διακανονιστικού πλαισίου. Νομίζω ότι η μείωση των περιορισμών χρήσης ενοικιαζόμενων οχημάτων θα πρέπει να συνοδευτεί επίσης από τροποποίηση συγκεκριμένων κανονισμών έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το παράνομο καμποτάζ το οποίο δυστυχώς σοβεί σήμερα. Είναι η κατάσταση δύσκολη και αν δεν ληφθούν συγκεκριμένες ρήτρες προστασίας θα χειροτερεύσουν 4 μήνες και 25% του συνόλου του στόλου της επιχείρησης θα πρέπει να βοηθήσουμε φυσικά την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να υπάρχει ισότητα ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ένα λεπτό, κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Η ε, χρήση ενοικιαζόμενων οχημάτων ε, είναι κάτι το οποίο επιτρέπεται εδώ και 25 σχεδόν χρόνια. Θα πρέπει να προσαρμοστεί η ρύθμιση αυτή για να καλύψει τις νέες ανάγκες. Υπάρχουν ε, δυνατότητες έτσι ώστε να προστατεύσουμε τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις εταιρείες ενοικίασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να αποκλείεται η χρήση οχήματος εταιρεία από άλλη χώρα, σε συγκεκριμένη χώρα, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να πληρεί ε, συγκεκριμένους όρους ασφαλείας. Ε, απαιτείται λοιπόν αυξημένη προσοχή η ηλεκτρονική εθνική καταγραφής θα πρέπει να καταγράφουν τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, την ε, κοινοτική άδεια κυκλοφορίας, όπως επίσης και τον χρόνο που επιτρέπεται ε, το συγκεκριμένο όχημα να κυκλοφορεί στο έδαφος τους. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Ο κύριος Μαριάς έχει ζητήσει το λόγο. Ένα Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το άνοιγμα της αγοράς είναι δεδομένο ότι θα οδηγήσει σε προβλήματα. Θα οδηγήσει σε αθέμητο ανταγωνισμό, θα οδηγήσει σε κλείσιμο μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κυρίως των ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι αυτή τη στιγμή λειτουργούν ε, τις ε, επιχειρήσεις ε, μεταφορών, οδικών μεταφορών ιδίως στην Ελλάδα. Θα ενισχυθούν έτσι κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα αυτό πρέπει να γίνει θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πρότυπα ασφαλείας υπάρχει ζήτημα με τα τέλη θα πρέπει να έχουμε πολύ πιο πράσινο προσανατολισμό επομένως καλύτερα να ενισχυθούν οι σιδηροδρομικές ε, μεταφορές. Ε, χρειάζεται εκπαίδευση των οδηγών νομίζω ότι μέτρα συγκεκριμένα όπως το ποσοστό των αυτοκινήτων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή ο χρόνος μίσθωσης είναι καθοριστικά. να επισημάνω ότι στην ελλάδα αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε εκατοντάδες πλέον βουλγαρικά φορτηγά τα οποία εισέρχονται στην ελλάδα και κάνουν κυρίως μεταφορές εσωτερικές δηλαδή καταστρατηγούν τις αποφάσεις που απαγορεύεται να κάνουν εσωτερικές μεταφορές και αυτό είναι ένα καθοριστικό θέμα το οποίο η κυρία bulc κατά την άποψή μας θα πρέπει να το δει. ευχαριστώ. Äh, Και τώρα δίνουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επίτροπο κυρία Μπουλ, θα έχει την ευκαιρία να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, σας ευχαριστώ για αυτή την σύντομη αλλά πολύ εμπεριστατωμένη συζήτηση. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλους τους βουλευτέ που βοήθησαν στη συζήτηση αυτού του σημαντικού θέματος και βεβαίω να ευχαριστήσω την εισηγητρία. Η χρήση μισθωμένων οχημάτων στην εσωτερική αγορά θα πρέπει να διευκολυνθεί. Και δεν υπάρχει λόγος να γίνει πιο δύσκολη η χρήση μισθωμένων οχημάτων από ότι η χρήση οχημάτων που είναι στην ιδιοκτησία του μεταφορέα και νομίζω ότι από αυτού συμφωνούμε όλοι. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι η πρόταση αυτή είναι υπέρ της υψηλότερης ασφάλειας για τους οδηγούς και της υψηλότερης οδικής ασφάλειας γενικότερα. Παράλληλα, συνεισφέρει άμεσα στη μείωση των εκπομπών ανθράκα για τις μεταφορές και για άλλη μια φορά τονίζουμε ότι μας απασχολεί το θέμα των οδικών μεταφορών γιατί αντιπροσωπεύουν το 70% όλων των εκπομπών των μεταφορών στην Ευρώπη. Άρα εστιάζουμε την προσοχή μας στη μείωση των εκπομπών μέσω των οδικών μεταφορών. Να προσθέσω δύο σχόλια μετά τα δικά σας σχόλια. Καταρχήν, για τον αποτελεσματικό έλεγχο, θέλω να πω ότι οι πινακίδες όλων των οχημάτων θα καταγράφονται στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα των μεταφορέων που είναι τμήμα του κανονισμού 1071. Το δεύτερο σχόλιο έχει σχέση με ένα σχόλιο που έγινε ε, λέγοντας ότι θα ε, είναι ε, λιγότερο ε, σωστές οι συνθήκες ανταγωνισμού για τους ε, οδηγούς. Θέλω να τονίσω ότι ο κανονισμός αυτός δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα δικαιώματα των οδηγών κατά κανένα τρόπο. Μετά την πρώτη ανάγνωση, πιστεύω ότι θα είναι εφικτό να ολοκληρωθεί ο τριμερής διάλογος εύκολα και μετά τη συζήτηση με τη Ρουμανική Προεδρία πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ελπίζω να έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση για αυτό το θέμα. Άλλη μια φορά θέλω να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική δουλειά που έχετε κάνει. Και τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους επικοδομητικό και ευτυχισμένο το 2019. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Και εμείς σας ευχόμαστε καλή χρονιά και θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την Επίτροπο για τα λόγια της καθώς και φυσικά όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην απόψινή συζήτηση και που συνεχίζουν τις προσπάθειες τους ε, για διαμόρφωση, οριστική διαμόρφωση της έκθεσής μου. Νομίζω ότι τελικά αύριο θα έχουμε ευρεία υποστήριξη και έτσι θα έχουμε ένα κείμενο που θα παρέχει ασφάλεια δικαίου σε μια αγορά όπου πρέπει να απελευθερώσουμε το δυναμικό της. Και αυτό μπορεί να το κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η διασυνοριακή αγορά μεταφορών είναι απαραίτητη ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να ανταποκρίνονται στις εποχικές τους ανάγκες. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι έτσι θα διασφαλίσουμε και μεγαλύτερη ασφάλεια στους δρόμους. Έτσι, οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν περισσότερα σε άλλους τομείς των επιχειρήσεών τους και όχι στον, στο όλο. Είναι πολύ σαφή η νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν όρια εκπομπών που θεσπίζονται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τα οποία θα πρέπει να τηρούνται. Δεν αναφέρθηκα στα οχήματα άνω των 6 τόνων, διότι αποτελούν αντικείμενο άλλη πρότασης. Θα πρέπει να φροντίσουμε τα, οχι... τα κράτη-μέλη να τηρούν το όριο των τεσσάρων μηνών για τη χρήση μισθωμένων οχημάτων και θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τα υπόλοιπα θέματα όπως είναι η φορολόγηση. Με αυτήν την νομοθετική πρόταση δεν θέλουμε να τροποποιήσουμε άλλες προτάσεις, όπως είπα στην εισαγωγή μου. Θέλουμε να φροντίσουμε όλες οι πληροφορίες να υπάρχουν σε εθνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων για να εξασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Σας ευχαριστώ πολύ. Έληξε η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί αύριο. Φτάνουμε στο επόμενο θέμα της ε, ημερησίας διάταξης, ε, την έκθεση της κυρίας Αγγέλικα Μιλνάρ, ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρία Μιλινάρ, έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές, και όλους ε, τους ε, συνεργάτες για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε για την έκθεση αυτή. Η ενσωμάτωση του φίλου, όπως γνωρίζουμε όλοι, τουλάχιστον όλοι εμείς που είμαστε υπέρ αυτής της έννοιας, είναι μια παγκόσμια αποδεκτή στρατηγική για να προωθήσουμε την ισότητα των φύλων. Η ενσωμάτωση της διάστασης του φίλου δεν είναι αυτός σκοπός, είναι όμως μια στρατηγική, μια προσέγγιση, ένα μέσο για την επίτευξη του σκοπού που είναι η ισότητα των φύλων. Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου διασφαλίζει ε, ότι θα, είναι, ε, θα έχουν κεντρική σημασία τα θέματα της ε, διάστασης του φύλου σε όλους τους τομείς. Στην ανάπτυξη πολιτικής, στην έρευνα, στην ομοθεσία, στην προετοιμασία των δαπανών των προγραμμάτων χρηματοδότησης. Και πιστεύω ότι το 2019 είναι απαράδεκτο ότι παρότι ο πληθυσμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά το ίμιση γυναίκε, κατά το ίμιση άνδρε, η σύνθεση ακόμη και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν αντικατοπτρίζει αυτή την ισορροπία. Μόνο 36,1% όλων των Ευρωβουλευτών είναι γυναίκε. Ω μόνιμη εισηγήτρια ε, για την ε, έκθεση σχετικά με την ισότητα των φύλων, θέλω να ενθαρρύνω όλες τις πολιτικές ομάδες ε, να διασφαλίσουν ε, την ε, ίση εκπροσώπηση των γυναικών και των ανδρών στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω συγκεκριμένων μεθόδων για ίση εκπροσώπηση και για τον, ε, για τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ισχύει το ίδιο, παρότι οι γυναίκες αποτελούν το 59% των υπαλλήλων, υποεκπροσωπούνται σε θέσεις ε, διευθυντών και προϊσταμένων και από το 2017 μειώθηκε μάλιστα το ποσοστό ε, γυναικών σε διευθυντικές θέσεις, σε υψηλές θέσεις και στην, σε μεσαίες διοικητικές θέσεις αυξήθηκε πολύ λίγο. Παραμένει χαμηλό το ποσοστό των γυναικών σε διοικητικέ θέσει και ζητώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προχωρήσει σε ίση εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσει που λαμβάνουν αποφάσει. Υπάρχουν ε, ε, γυναίκες ικανές ε, να καλύπτουν τα κενά αυτά και υπάρχει μεγάλος αριθμός γυναικών από τις οποίες μπορεί να γίνει η επιλογή αυτών των στελεχών. Και πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για να κινηθούμε προς μια κουλτούρα ισότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει τη συμμετοχή όλων και η έκθεσή μου ζητεί την ε, ε, ίση μεταχείριση προς όλους και προς την κοινότητα των ΛΟΑΔΜ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει ε, να μεριμνά για ίσα δικαιώματα όλων των ταυτοτήτων φύλου. Όσον αφορά τη σεξουαλική παρενόχληση, τονίζουμε ότι είναι ε, ένα σημαντικό έγκλημα, μια ακραία μορφή ε, παραβίασης της ισότητας των φύλων. Πολύ μικρή πρόοδος γίνεται για την υλοποίηση των ψηφισμάτων, των συστάσεων των ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάρτιση που θα πρέπει να προσφέρεται και στους ευρωβουλευτές και στο προσωπικό σχετικά με την σεξουαλική παρενόχληση και για την χρήση εξωτερικών εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα εξετάζουν τη σεξουαλική παρενόχληση στην, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι η ισότητα των φύλων δεν είναι θέμα που αφορά μόνο τις γυναίκες ίσως οι άνδρες έχουν και μεγαλύτερη ευθύνη να κινηθούν προς την κατεύθυνση της ισότητας των φύλων. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Χρειάζεται συνεχής δέσμευση υπέρ της ισότητας των φύλων για να μπορέσουμε σε όλα τα επίπεδα να την εφαρμόσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω λοιπόν ότι θα έχω αύριο την υποστήριξή σας και μια θετική ψήφο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία εισηγήτρια. Δίνουμε το λόγο στην Επιτροπή. Κυρία Κιούροβα. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μλινάρ για την ε, δεύτερη της έκθεση για την ενσωμάτωση της διάστασης ε, του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για, το Ευρωπαϊκό, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και, τους, ε, και τα θεσμικά τη όργανα δεν είναι επιλογή η ενσωμάτωση τη διάσταση του φύλου, είναι υποχρέωση η οποία θεσπίζεται στη συνθήκη, στο κεκτημένο και στο χάρτη θεμελιωτών δικαιωμάτων. Η, ισότητα των δύο φύλων δεν αποτελεί ακόμα απτή πραγματικότητα για όλους. Οι δείκτε δείχνουν στασιμότητα και εάν ε, βλέπουμε εξελίξεις είναι μάλλον περιθωριακές. Και αυτό δυστυχώ αληθεύει και για τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ισορροπία των δύο φύλων μεταξύ των Ευρωβουλευτών ε, ε, σχεδόν δεν έχει αλλάξει από το 2009, από το 35% στο 36,4%. Και οι γυναίκες αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύουν το 32,1% των ε, Ευρωπαίων Επιτρόπων, δηλαδή 9 από τους 28 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι περιορισμένη η θέση των γυναικών ε, στις ε, ηγετικέ θέσεις. Στη, σε μια δημοκρατία έχει σημασία η ισότητα των δύο φύλων. Η καλύτερη ισορροπία των φύλων μπορεί να αυξήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να βελτιώσει τη λειτουργία των δημοκρατιών μας. Μάλιστα, όπως είπε η κυρία Μλινάρ, φέτος πολιτικά κόμματα και τα κράτη-μέλη μπορούν να δείξουν την προσήλωσή τους στην ισότητα των δύο φύλων και να διασφαλίσουν η ισορροπημένη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις κορυφαίες θέσεις των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ε, σας καλώ λοιπόν ε, να φροντίσετε οι υποψηφιότητες σας να είναι ισορροπημένες. Τα θεσμικά όργανα πρέπει να εξυπηρετούν τους ανθρώπους και ε, πρόεδρος Γιούγκερ ε, έχει θέσει στόχο ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 40% στις κορυφαίες θέσεις να κατέχεται από γυναίκες. Οι γυναίκες κατέχουν, κατέχουν το 37% των υψηλότερων θέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ στις θέσεις μεσαίων διευθυντών έχει επιτευχθεί ο στόχος του 40%. Πρέπει να εντοπίσουμε και να στηρίξουμε τις ε, ικανές ε, γυναίκες ε, με στοχευμένες δράσεις. Η έκθεση θέτει το σκηνικό και για την επόμενη θητεία και γι' αυτό επικροτώ αυτή την προορατική προσέγγιση. Όπως γνωρίζετε, η στρατηγική προσήλωση ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, εκφράζεται με την πολιτική της ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός αυτής. Το 2019 επίσης λοιπόν εξετάζουμε την πρόοδο και ε, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία για να θέσουμε προτεραιότητες για το μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε πολύ να ακούσουμε και τις θέσεις ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Φτάνουμε στους ομιλητές από τις πολιτικές ομάδες. Ε, κύριε Φαρία, δύο λεπτά έχετε εκ μέρους του ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ συνάδελφοι, ευχαριστώ Επίτροπε. Ευχαριστώ τους εισηγητές για την εξαιρετική τους προσπάθεια στον τομέα του gender mainstreaming στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι αλήθεια ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διασφαλίσει την ισότιμη μεταχείριση των γυναικών. Ε, ξέρουμε ότι τα πράγματα επιταχύνθηκαν μετά από την αποκάλυψη του λεγόμενου σκανδάλου Βάινστάιν και η αλήθεια είναι ότι ναι να αντιμετωπίζουμε αρκετά θέματα αλλά εξακολουθούμε να αποσιωπούμε αρκετές περιπτώσεις μέχρι τώρα. Καιρός είναι να αλλάξουν τα πράγματα. Θα πρέπει η Συμβουλευτική Επιτροπή ε, για τέτοιου είδους θέματα να προσπαθήσει να διαγράψει αυτό τον φόβο ο οποίος εξακολουθεί να σοβεί στο Κοινοβούλιο σήμερα. Οι συμπεριφορές αυτές είναι απάνθρωπες και αποδεικνύουν την ανισότητα που εξακολουθεί να υπάρχει ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Επίσης στις διαδικασίες εξέλιξης επαγγελματικής και καριέρας υπαλλήλων θα πρέπει οι επιλογές να γίνονται αποκλειστικά βέβαια με τις ικανότητες ε, και ε, τα ποιοτικά στοιχεία του κάθε υποψηφίου και όχι με το φύλλο. Νομίζω όμως ότι η προοπτική του φύλου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη συνολικότερα και γι' αυτό το έγγραφο που έχει προετοιμαστεί προς ψήφιση αύριο είναι σωστά προπαρασκευασμένο, είναι δίκαιο έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η σκοτεινή πραγματικότητα. Ζητώ από τους συναδέλφους να υπερψηφίσουν την αυριανή πρόταση. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Χέτ, δύο λεπτά εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Μλινάρ και όλου τους άλλους για μια εξαιρετική έκθεση η οποία λαμβάνει υπόψη τις περισσότερες πτυχές που είναι αποφασιστική σημασία ώστε το Κοινοβούλιο κάποια στιγμή στο μέλλον να πετύχει την απόλυτη ισότητα ανδρών και γυναικών. Αυτό θα πρέπει να συμβεί, διότι οι πολιτικές που υιοθετούμε θα πρέπει ε, να αφορούν εξίσου και τα δύο φύλλα τα έγγραφα του Κοινοβουλίου και οι συζητήσεις ε, θα πρέπει ε, να εκπονούνται σε απόλυτο πνεύμα ισότητας ε, των δύο φύλων. Είναι σημαντικό δηλαδή να ενσωματωθεί αυτή η διάσταση σε όλες τις εργασίες του Κοινοβουλίου. Επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης που αποτελεί μορφή διάκρισης λόγω φύλου. Εάν μάθαμε κάτι από την εκστρατεία MeToo είναι ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σοβαρά το, το θέμα και θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για όλους τους ευρωβουλευτές ε, να ε, λάβουν εκπαίδευση στο θέμα της ε, σεξουαλικής παρενόχλησης. Σε σχετική εκδήλωση ήμουνα, είμαι μόνη ευρωβουλευτής που ήταν παρούσα. Ε, αυτό ε, ε, αυτό είναι ντροπή. Θα πρέπει λοιπόν η σχετική εκπαίδευση να γίνει υποχρεωτική. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ομάδα εργασία που εξετάζει το θέμα τη σεξουαλική παρενόχλησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι όμω δουλειά που δεν μπορεί να κάνει μόνο του το Κοινοβούλιο. Χρειαζόμαστε βοήθεια και εμπειρογνωσία από εξωτερικού παράγοντε. Επίση, είναι πολύ σημαντικό όλα ε, όλες οι πολιτικές ομάδες και όλα τα πολιτικά κόμματα να έχουν ε, ε, ισόρροπα ψηφοδέλτια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκέρικε από το ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση για την ισότητα των φύλων ε, ε, έγινε από την Επιτροπή Γυναικών. Μόνο τρει βουλευτέ είναι άνδρες. Τρει από τους 22. Ε, φαίνεται ότι για τη δημοκρατία μας η ισότητα των φύλων δεν μπορεί να μπει στο επίκεντρο των μελημάτων μας χρειαζόμαστε γυναίκες ε, στην οικονομία, χρειαζόμαστε γυναίκες στην αγορά ε, να αναλάβουν θέσεις ε, τις οποίες πολύ συχνά δεν θέλουν. Υποχρεώνουμε τις γυναίκες να αφήνουν τα παιδιά τους σε παιδικούς σταθμούς για να αναλάβουν θέσεις εργασίας. Δεν είναι καλό ούτε για τις γυναίκες, ούτε για τα παιδιά αυτά, ούτε για τις μητέρες, ούτε για τα παιδιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση ενωμένη στην πολυμορφία. Πού είναι ε, η πολυμορφία όταν θέλουμε να εξομοιώσουμε τις γυναίκες με τους άνδρες. Θα πρέπει ε, να χαιρετίζουμε την πολυμορφία και τη διαφορετικότητα ανδρών και γυναικών και να αφήνουμε τις γυναίκες να επιλέξουν ε, το επάγγελμα που θέλουν. Αυτό θα οδηγήσει και σε περισσότερους άνδρες στην Επιτροπή Γυναικών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε και εγώ θα χαρώ αν είναι περισσότεροι άνδρες στην Επιτροπή Γυναικών. Και σίγουρα ε, θα ήταν ε, θετικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχουμε ίση εκπροσώπηση γενικότερα. Εκ μέρους των φιλελευθέρων, Μπιλμπάου Μπαραντίκα. Ευχαριστώ Επίτροπε. Θέλω να συγχαρώ την Αγγέλικα Μίλλερ γιατί πράγματι με ιδιαίτερα παιδαγωγικό τρόπο επιδεικνύει την κατάσταση ανισότητας η οποία υπάρχει σήμερα. Ε, εδώ δεν μένουμε στη θεωρία. Γίνονται συγκεκριμένες ε, προτάσεις ε, και θα πρέπει να δούμε όχι το τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανα, αλλά το τι κάνουν. Θα πρέπει να υπάρξει μια προσπάθεια και πολιτική και δημοσιονομική έτσι ώστε να περάσουμε στις πράξεις. Οι σκέψεις οι οποίες παρουσιάζονται και τα μέτρα τα οποία προτείνονται είναι απλά μία αναγκαιότητα, γιατί αλλιώς χωρίς τα μέτρα αυτά δεν θα υπάρξει ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών. Βλέπουμε τα ποσοστά Επίση ακούγονται διάφορα σεξιστικά συμβάντα, κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα σωστά μέτρα τα οποία έχουμε αναλάβει να παίρνουμε. Θα πρέπει να επικοινωνούμε καλύτερα εγώ η ίδια και το έχω πει προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπάρξει πραγματικά μια προσπάθεια διαφορετική από αυτήν που έγινε ε, μέχρι τώρα με οργανωτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Λουξεμβούργο και η οποία είχε σαν βάση θα έλεγα μια εκπροσώπηση κυρίαρχα αρένων και όχι γυναικών. Συνεπώς λοιπόν δεν θα πρέπει να μείνουμε σε τέτοιου είδους ρυθμίσεις. Ε, η σεξουαλικότητα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σωστό τρόπο και να μην αντιμετωπίζεται με επιθετικότητα ανάλογα με τον προσανατολισμό του καθενός. Θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες προτάσεις και θα πρέπει να κρίνουμε τα αποτελέσματα των προτάσεων αυτών. Τότε μόνο θα μπορέσουμε να διορθώσουμε την κατάσταση. Ο λαϊκισμός της άκρας δεξιάς μας στρέφει στο παρελθόν και προωθεί την έννοια της βίας της σεξουαλικής. Ευχαριστούμε κυρία Μπιλμπάου. Ο κύριος Όσνιας ε, έχει μια γαλάζια κάρτα. Τη δέχεστε? Ναι. Κύριε Όσνιας παρακαλώ. E, Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε 130 οδηγούς, 110 οδηγούς, εκ των οποίων δύο είναι γυναίκες. Νομίζετε ότι αυτό είναι διακριτική μεταχείριση κατά των γυναικών ή είναι κατανοητό ότι ενδεχομένως δεν ενδιαφέρονται οι γυναίκες για μια θέση οδηγού. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για θέσεις διευθυντικές. Αυτό δεν θα το λάβετε υπόψη σας. Κυρία Μπιλμπάου. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Εσείς αναπαράγετε τα στερεότυπα τα οποία ισχύουν για τις γυναίκες. Οι γυναίκες είναι ικανές να αναλάβουν η αδίποτε μορφή επαγγελματικής δραστηριότητας και ευθύνης. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν στη διάθεσή τους τις ίδιες ευκαιρίες. Όταν μάθαινα να οδηγώ, ο καθηγητής μου μου έλεγε, ο δάσκαλός μου, ε, μου έλεγε ότι οι μελέτες έδειχναν ότι οι γυναίκες οδηγούν καλύτερα, είναι πιο προσεκτικές, ε, οργίζονται λιγότερο και προκαλούν λιγότερα ατυχήματα. Αυτό πρέπει κάτι να σας πει. Και φυσικά αν υπάρξουν περισσότεροι οδηγοί γυναίκες στο Κοινοβούλιο η κατάσταση σίγουρα θα βελτιωθεί. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Έγκστρομ από τους Ένα λεπτό. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια, την κυρία Μπλινάρ, που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά με την έκθεση αυτή. Μπορούμε και πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μια ίση Ευρώπη. Σήμερα έχουμε ένα σχέδιο δράσης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για όλες τις εργασίες του Κοινοβουλίου. Η ισότητα δίνει σε όλους τους ανθρώπους τη δυνατότητα ε, να εκμεταλλευτούν τις ικανότητές τους ε, στο έπακρον η διακρίση η παρενόχληση και η βία στις ανθρώπινες σχέσεις ε, αποτελούν σημαντικό κόστος και για τα άτομα και για την κοινωνία. Χρειάζεται σωστή εκπαίδευση, αλληλεγγύη. Θα πρέπει όμως επίσης να μπορούμε να εντοπίσουμε τα προβλήματα και να αλλάξουμε την κατάσταση. Και ε, οι άντρες πλήττονται από διακρίσεις. Ε, θα πρέπει να να καταρρύψουμε το, και το ε, ανδρικό ιδανικό. Θα πρέπει να φροντίσουμε όλες οι εργασίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διεξάγονται η μισότητα των δύο φύλων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φορένσα από την ΚΟΕ, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι στη συγκήτρια τη ΚΟΕ Ευχαριστώ την Αντζέλικα για την προσπάθεια που έκανε. Επίσης ευχαριστώ και τους υπόλοιπους σκιώδεις και τους υπαλλήλους που πήραν μέρος για να αντιμετωπιστεί ένα τόσο δύσκολο πρόβλημα ε, σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη συμπερίληψη της πολιτικής και προβληματικής των φύλων σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα φεμινιστικά κινήματα τα οποία ιστορικά επιδιώκουν να υπάρξει μια ισότητα για όλα τα ανθρώπινα όντα, για όλους τους πολίτες που υφίστανται διακρίσεις, που υφίστανται βία στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών σχέσεων και γενικότερα των κοινωνικών διακρίσεων θα πρέπει να υπογραμμίσουμε κάτι το οποίο νομίζω περιλαμβάνεται στην έκθεση και με ικανοποιεί αυτό. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά το mainstreaming στους ευρωπαϊκούς κανόνες αν δεν υπάρξει δυνατότητα, αν θέλετε, ε, αυτονομίας των γυναικών οι γυναίκες σαν παράδειγμα παράγουν στην Ιταλία μέσω συγκεκριμένων οργανώσεων ιδέες, προγράμματα και σε τοπικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο και αυτό θα πρέπει να γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θα πρέπει με τη λογική της υπερχρέωσης και με το άλοθη το λογιστικό ε, να θίγονται οι γυναίκες και τα συμφέροντά τους. Οι γυναίκες είναι συν, οι γυναίκες δεν είναι μείον. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή φεμινιστική πολιτική, κάτι το οποίο εμπνέει καθημερινά την δράση μου εδώ. Παρακαλώ όλους τους ομιλητές να τηρούν το χρόνο ομιλία τους και δίνω το λόγο για Τροτζίνσκι. Κύριε Επίτροπε. Η έκθεση αυτή είναι πραγματικά θα έλεγα σαν να έχει έρθει από τη σελήνη. Στην ουσία προτείνεται μια ισοτιμία αυστηρότατη και ποσοστώσεις απόλυτες και ταυτόχρονα βλέπετε ότι αμφισβητείται η θέση των γυναικών εσείς στα πλαίσια αυτής της λογικής σας που εξισώνει τα πάντα δεν κατανοείτε την πραγματικότητα. Πώς μπορεί να έχει εμπιστοσύνη ε, σε κάποιον ο οποίος είναι μέλος μιας επιτροπής πρόσληψης όταν είναι υποχρεωμένος να σεβαστεί παράλογες ποσοστώσεις. Δεν μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι όταν λέμε ότι εξελέγει η συγκεκριμένη γυναίκα επειδή είναι γυναίκα. Υπάρχουν και άλλες βλακίες μέσα στην έκθεση αυτή χρησιμοποιείται μια ρητορική εις βάρος ε, των γυναικών και η κατάσταση δυστυχώς ε, θα ήταν κομική αν δεν ήταν τόσο σοβαρή. Εγώ σκέφτομαι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Γαλλία, τα κίτρινα γυλαίκα που δεν θέλουν να διαλέγουν οι άνθρωποι αυτοί μέσα στο να πάρουν παιχνίδια για τα παιδιά τους και να ζεστάνουν το διαμέρισμά τους και να βλέπουν το τι κάνουμε εμείς. Δυστυχώς ε, έχουμε αυτά τα σύνορα τα διάτρητα με χιλιάδες ε, μετανάστες να πηγαίνουν έρχονται και οι πολιτικές ε, του Γιούνκερ επιτρέπει στον κοινοτισμό και στον Ισλαμισμό να διαβρώνουν τις κοινωνίες μας και εσείς προωθείτε ε, πρότυπα όπως ο κύριος Μακρό, ο οποίος ε, θέλει στην ουσία να αποδείξει ότι δεν έχει, όπως και εσείς, καμία σχέση με την πραγματικότητα. Νομίζω ότι στην εκλογική αναμέτρηση θα σας δείξουν. Ευχαριστώ πολύ. Μία γαλάζια κάρτα από την κυρία Φορέντζα. Τη δέχεστε? per δευτερόλεπτα. Αν εσείς ακούσατε μια ε, αμφιβολία που ακούστηκε προηγουμένω ότι οι γυναίκες μπορεί και να μην είναι σε θέση να οδηγούν αυτοκίνητα. Προφανώς αυτό είναι προκατάληψη. Δεύτερον, υπάρχει μια τεράστια απόσταση στις αμοιβέ ανδρών και γυναικών. Τώρα για τις προσλήψεις. Εγώ δεν θέλω να είμαι ένα ποσοστό ε, για τον άνδρα ο οποίος επιλέγει ε, είτε άνδρες είτε γυναίκες για συγκεκριμένες θέσεις. Θέλω να υπάρχουν και γυναίκες που να είναι σε θέση να προσλαμβάνουν. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Εγώ δεν μίλησα για αυτοκίνητα και για οδηγούς γυναίκες. Θα συμφωνήσω μαζί σας για την ισότητα ανδρών γυναικών στο μισθολογικό. Είναι το ελάχιστο επιδιώξιμο. Πρέπει να αλλάξουν οι νοοτροπίες, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να προέλθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει εσείς να υποχρεώσετε τον κόσμο ε, να προσλαμβάνει γυναίκες επειδή είναι γυναίκες. Πρέπει να προσλαμβάνονται οι γυναίκες και να είναι υποψήφιες στις εκλογές σαν παράδειγμα οι γυναίκες επειδή είναι ικανές να το κάνουν. Μπρούνο Γκόλνης είναι ο επόμενος ομιλητής. Ένα λεπτό. Το 1453 όταν η Κωνσταντινούπολη πολιορκείται από τους ε, Τούρκους βυζαντινολογούσαμε. Τώρα μιλάμε για το φίλο των βουλευτών. Η έκθεση αυτή έχει όλα τα μειονεκτήματα τα οποία θα μπορούσαμε να βρούμε. Ε, είναι πάρα πολύ εκτεταμένη ξεκινάει από την ιδέα ότι ο ρόλος των ανδρών και των γυναικών που εκ είναι συμπληρωματικός θα πρέπει να είναι παντού και πάντοτε απόλυτα ταυτόσιμος. Το μόνο που μετράει για σας είναι να υπάρχουν απόλυτα ίσοι αριθμοί ανδρών και γυναικών παντού, ανεξάρτητα από τις ευαισθησίες και τις προτιμήσεις των μεν και των δε. Ισότητα παντού το τρίτο, τέταρτο, πέμπτο φίλο των ΛΟΑΔΜ που συνέχεια πιπηλάτε εδώ, πού θα το βάλετε λοιπόν αν έχετε ισότητα ανδρών και γυναικών. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κοσλόφσκα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ξεκινήσω με μία παρατήρηση. Με εκπλήση, που σε τούτη την αίθουσα ακούμε ανθρώπους να αμφισβητούν την ε, ανάγκη κατάρριψης των ε, στερεοτύπων. Εάν δεν είχαμε καταρρύψει τα στερεότυπα αυτά, δεν ε, θα είχαμε γυναίκε σε τόσο υψηλέ θέσει. Ε, θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ την κυρία Αγγέλικα Μίλνερ για την εξαιρετική τη έκθεση. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η ενσωμάτωση τη διάσταση του φύλου είναι υψή τη σημασία εάν θέλουμε να πετύχουμε την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών. Άλλωστε, αυτό είναι κάτι το οποίο στηρίζεται από τις συνθήκες και το κοινοτικό κεκτημένο. Εάν θέλουμε να πετύχουμε το στόχο αυτόν και να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να καταβάλουν προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή, είναι σαφές ότι τα θεσμικά όργανα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποτελέσουν υπόδειγμα, να δείξουν πώς πρέπει να λειτουργεί ένα τέτοιο θεσμικό όργανο με την εφαρμογή των αρχών της ίσης μεταχείρισης. Έχουμε πολλές αιτιολογημένες προτάσεις ε, έχουμε συμπεράσματα ε, Αναφερόμαστε στην ε, καταπολέμηση της ε, σεξουαλικής παρενόχλησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναφερόμαστε και στο θέμα της σύνθεσης του Κοινοβουλίου. Είναι πολύ σημαντικά τα θέματα αυτά. Επίσης, η έκθεση καλή. μεγαλύτερη συμμετοχή σε ενημερωτικές εκστρατείες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Δέχεστε μία γαλάζια κάρτα από τον κύριο Σόσνιετς. Δέχεστε γαλάζια κάρτα από τον συνάδελφο κύριο Σόσνιερτς. Όχι, δεν δέχομαι ερώτηση διότι θέλω να καταπολεμήσω τις ανισότητες. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα να συνεχίσουμε. Ροντρίγε από το S&D και μετά η κυρία Βυσνιεύσκα. Ροντρίγε, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, καλή χρονιά σε όλους. δεν έχουμε περισσότερους άντρες στην ε, Επιτροπή Γυναικών, ε, διότι ε, δεν θέλουν να συμμετέχουν. Όταν βλέπουμε το θέμα της ενσωμάτωσης τη διάσταση του φίλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να τα εξετάσουμε τα θέματα αυτά. Το συζητούσαμε πριν χρόνια, το συζητάμε ακόμα και σήμερα. Το 36% των μελών του Κοινοβουλίου είναι γυναίκε και αυτό αποτελεί δείγμα τη έλλειψης προοπτικής για τα δύο φύλλα. θα ήταν πολύ χρήσιμο εάν και άλλα κρατημέρια ακολουθήσουν το παράδειγμα της Πορτογαλίας να έχουν ε, ψηφοδέλτιο με εξίσου πολλούς άντρες και γυναίκες. βλέπουμε ότι στις ψηλέ θέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μόνο το 33% των είναι γυναίκες. Αυτό λοιπόν δεν είναι πολύ καλό δείγμα. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Βυσνιεύσκα, αλλά βλέπω ότι ο κύριος Σόσνιερτς ε, ζητάει γαλάζια κάρτα. Θα σας δώσω το λόγο σε λίγο όμως, ε, γι' αυτό δεν θα σας δώσω τη δυνατότητα να μιλήσετε τώρα. Κυρία Βυσνιεύσκα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η έκθεση για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, λίγα κοινά στοιχεία έχει με τον τίτλο της. Αν θέλουμε πραγματικά να εστιάσουμε στα προβλήματα που έχουν σχέση με τη διάσταση του φίλου, ένα από τα βασικά προβλήματα, αν όχι το πλέον βασικό πρόβλημα, είναι η συμφιλίωση της ε, προσωπικής με την επαγγελματική ζωή. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα των γυναικών και μου κάνει εντύπωση που η έκθεση αυτή δεν ε, εστιάζει σε αυτό το σημαντικό πρόβλημα γιατί οι γυναίκες θέλουν και να είναι μητέρες και να έχουν οικογένεια και να αναπτυχθούν επαγγελματικά. Πρέπει λοιπόν ε, να θεσπιστούν κανόνες που θα δίνουν τη δυνατότητα στις γυναίκες να συμφιλιώνουν την προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Οι γυναίκες έχουν τη ζωή τους είναι μορφωμένες και δεν χρειάζονται βοήθεια ε, στο να προωθηθούν. Οι βοηθοί μας δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το πιο σημαντικό ζήτημα για τις εργαζόμενες αυτές είναι να μπορέσουν να συμφιλιώσουν τη δουλειά τους στο κοινοβούλιο με τη δουλειά τους στην οικογένειά τους. Είπατε ότι είναι πολύ λίγοι οι άνδρες βουλευτές στην Επιτροπή Γυναικών και δεν μου κάνει εντύπωση γιατί σε αυτή την Επιτροπή ε, κυρίως επικρατεί λαϊκισμός της άκρας αριστεράς που καταλήγει στο ότι η πραγματική ισότητα γελιοποιείται από την αριστερά πτέρυγα του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Θέλετε να δεχτείτε μια καλά διακάτα από την κυρία Ρέγνερ. Ναι, βεβαίως. Κυρία Ρέγνερ, μία σύντομη ερώτηση. Ε, γνωρίζετε ότι ο τίτλος της έκθεσης «Ενσωμάτωση της διάστασης του φίλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» ε, είναι ακριβώς αυτό το θέμα το οποίο περιλαμβάνεται στην έκθεση. Η έκθεση δεν μιλά για τη συμφιλίωση ε, της επαγγελματικής με την προσωπική ζωή. Αυτό είναι ο τίτλος ε, και περιλαμβάνει αυτά τα σημαντικά θέματα που έχουν άμεση σχέση. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, και η Επίτροπος και η συγγήτριά μας είπαν ότι αναλογικά λίγες ε, γυναίκες ε, είναι σε διευθυντικές θέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι τόσο λίγες οι γυναίκες, κατά τη γνώμη μου, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα για τις γυναίκες αυτές να συμφιλιώσουν την προσωπική με την επαγγελματική ζωή. Και αυτός είναι και ο λόγος που προχωρούν πιο αργά οι γυναίκες στην επαγγελματική τους καριέρα. Στην έκθεση αυτή προβλέπεται κατάρτιση για τη σεξουαλική παρενόχληση. Η γνώμη σα για του βουλευτέ και του υπαλλήλου του Κοινοβουλίου είναι τόσο χαμηλή ότι πρέπει να του διδάξουμε πώ να αποφεύγουν τη σεξουαλική παρενόχληση. Σα κάνει εντύπωση που δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή δεν συμμετέχουν σε, τέτοιες, ε, σε τέτοιου είδους κατάρτιση γιατί είναι μορφωμένοι άνθρωποι που δεν θα ε, ενεπλέκονται σε τέτοιες ε, πράξεις. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό κύριε Σόσνιετς. Είχατε κάνει και ερωτήσεις νωρίτερα με γαλάζια κάρτα. Μπορείτε να τα πείτε όλα τώρα κύριε Σόσνιετς. Ο τίτλος της έκθεσης θα έπρεπε να είναι σεξισμός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να γνωρίζουν όλοι περί τίνο ε, πρόκειται. Τα αρνητικά στερεότυπα μάλλον προέρχονται από τέτοιες ανόητε εκθέσεις όπως είναι αυτή. Είναι ντροπή για γυναίκες και για τις φεμινίστριες να θέλουν να προσλαμβάνονται γυναίκες μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκες. Ο φεμινισμός είναι ντροπή για τις γυναίκες. Στο σημείο 40 λέει ότι ε, θέλει κυρώσεις για όσα λέγονται. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να πω ότι δεν φοβάμαι τις κυρώσεις σας. Δεν μπορείτε να επιβάλλετε κυρώσεις για όσους λένε την αλήθεια. Και δεν θα αποφασίσετε εσείς τι μου επιτρέπετε να λέω και τι όχι. Θα έπρεπε να αποσυρθείτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν δεν καταλαβαίνετε τι είναι η ελευθερία λόγου και το ίδιο ισχύει για τον κύριο Ταγιάννη. Παρακαλώ. Η κυρία Ζαμπόρσκα, μισή λεπτό από το ΕΛΚ. Κύριε Επίτροπε. Κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα Σύμφωνα με το κείμενο αυτό θα έπρεπε να σας απευθύνω το λόγο με όρο που δεν θα περιγράφει αρσενικό ή θηλυκό, αλλά στη μητρική μου γλώσσα δεν δίνεται η δυνατότητα να κάνω διάκριση μεταξύ του και της Προέδρου, του και της ε, Επιτρόπου. Αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε τη γλώσσα η οποία εξελίσσεται επί εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια. Ε, μερικές φορές αυτές οι εκκλήσεις ε, προς κάτι το παράλογο υπονομεύουν την αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πολλές φορές επισκιάζουν χρήσιμες πρωτοβουλίες, παραδείγματο χάρη για τη βελτίωση των γυναικών στο χώρο εργασίας ή την μηδενική ανοχή για σεξουαλική παρενόχληση ή την ε, ίση αμοιβή για ίση εργασία ανδρών και γυναικών. Μετά από 14 χρόνια ε, εμπειρίας στην ε, ευρωπαϊκή πολιτική, είμαι πεπισμένη ότι σε κάθε θητεία του Κοινοβουλίου συζητούνται αυτά τα θέματα και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο συζητούνται αυτά τα θέματα είναι εις βάρος των ίδιων των γυναικών. Μιλάμε για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, για την ίση θέση και ανδρών και γυναικών και αυτό θα προωθήσει την καλύτερη θέση των γυναικών στην κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Julie Ward από τους Σοσιαλδημοκράτες. Ένα λεπτό. Χαίρομαι γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίρνει σοβαρά το θέμα της ισότητας. Ζούμε μια εποχή όπου οι συντηρητικοί στρέφονται εναντίον των γυναικών, των νέων γυναικών όπως και των ΛΟΑΤ. Είναι σαφές ότι πρέπει να ρυθμίσουμε καλύτερα τα πράγματα και να προσθέσουμε την προοπτική του φύλου και στις ευρωπαϊκές πολιτικές και στην διοικητική λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το θέμα εδώ δεν αφορά μόνο στις γυναίκες. Είναι σημαντικό επίσης και για τους ΛΟΑΤΣΙΝ που πολλές φορές αγνοούνται πλήρως στο σχεδιασμό των πολιτικών. Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε σε επίπεδο προστασίας της διαφορετικότητας και ε, φοβάμαι ότι οι ανώτερες τάξεις κυρίως εκπροσωπούνται σε όργανα σαν το δικό μας. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε συνθήκες πραγματικής δημοκρατίας όπου όλοι να εκπροσωπούνται. Πρέπει επίσης να βοηθήσουμε τις γυναίκες με συμβούλους εργασίας, ε, όπως επίσης και τους ΛΟΑΤΣΙΝ. Κάποιοι από αυτούς θα είναι στη θέση μας και δεν θα πρέπει εμείς φεύγοντας να πάρουμε τη σκάλα εισόδου στο επίπεδό μας μαζί μας. Μία ερώτηση από την κυρία Βυσσεύσκα. Δέχεστε γαλάζια κάρτα? Madam Vishnevska, from ECR. Thank you. The floor is yours, Madam. E, e, e, Ευχαριστώ. Θα ήθελα ε, να διαμαρτυρηθώ διότι αναφέρετε τους συντηρητικού ως εχθρούς ε, των γυναικών και των ε, κοριτσιών. Δεν είναι σωστό αυτό και παρακαλώ να μην στιγματίζετε άλλους με αναλυθείς δηλώσεις. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Κατά τη γνώμη σας, πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε ε, γλώσσα ουδέτερη ως προς το φύλλο και κατά αυτόν τον τρόπο ε, να βελτιώσουμε τις ευκαιρίες για τις γυναίκες. Σας ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε και δίνω το λόγο στον κύριο Ούντο Βόιχτ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μου κάνει εντύπωση το σημείο 40 του σχεδίου κειμένου. όπου αναφέρεστε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά στηρίζεται μία μη θεμητή απόφαση του Προέδρου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να παρεμβαίνει στην ελευθερία του λόγου και η πολιτικά ορθή λογοκρισία από την αριστερή πτέρυγα της αίθουσας ε, ε, έχει λάβει τώρα έναν κόλαφο και βλέπουμε ότι το κείμενο αυτό αποτελεί προσπάθεια να αναμειχθεί στις εργασίες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παρέμβει στις εργασίες του. Ευτυχώς ακούγονται όλα και περισσότερες φωνές, όπως ε, και η δική μου. που τολμούν να μιλήσουν ειλικρινά. Ναι, για μένα η οικογένεια αποτελείται από γυναίκα, άντρα και παιδιά και η Ευρώπη θα έχει μέλλον μόνο όταν ξεφύγουμε από την ε, αφύσικη πολιτική και από την αναγνώριση περισσότερων φίλων από αυτά τα δύο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σόντροβα από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, θα ήθελα να θυμίσω σε όλους μας ότι η τελευταία έκθεση για την ενσωμάτωση του, της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητήθηκε το 2016. Τότε έγινε έκκληση για ίση συμμετοχή στην Επιτροπή Γυναικών. Τρία χρόνια έχουν περάσει σχεδόν και ελάχιστα έχουν αλλάξει. Η ίση εκπροσώπηση απέχουμε πολύ από την ίση ε, συμμετοχή και ιδιαίτερα στην Επιτροπή Ισότητας που θα έπρεπε να έχει αν μη τι άλλο συμβολική αξία για το Κοινοβούλιο. Ε, εάν δεν πετύχουμε τον στόχο αυτό, είναι υποκριτικό να υπαγορεύουμε σε άλλους ε, την ίση μεταχείριση εφόσον δεν μπορούμε εμείς να πετύχουμε τους στόχους μας, πόσο μάλλον στην Επιτροπή που στόχο έχει να ασχοληθεί ακριβώς με το θέμα αυτό. Εφτά άντρες από τα 33, 7 είναι άντρες από τα 33 τακτικά μέλη και από τους 22 αναπληρωτές ε, πάλι έχουμε 7 άντρες. Αυτό απέχει πολύ από την ίση εκπροσώπηση. Ό,τι και να λέμε εδώ πέρα αποτελούν δικαιολογίες. Έχουμε στρατηγικές, εκθέσεις, ψηφίσματα, αλλά τίποτα δεν αλλάζει επί της ουσίας. Πιστεύω ότι πραγματικός μας στόχος θα πρέπει να είναι η πραγματική ισότητα ανδρών και γυναικών. Αυτό σημαίνει για τις γυναίκες να κάνουν αυτό που μπορούν να κάνουν καλά, τη μητρότητα δηλαδή. Χρειάζονται μια αξιοπρεπή σταδιοδρομία αλλά και αξιοπρεπή συνθήκες για να μπορέσουν να φροντίσουν τις οικογένειές τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής η κυρία Ρέγνερ. Σας ευχαριστώ. Ο στόχος της ισότητας ε, θεσπίζεται στην ε, Ιδρυτική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Ανήκει δηλαδή στο DNA της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ίση μεταχείριση και αντιμετώπιση και σημαίνει επίσης και σωστή κατανομή της εξουσίας. Αυτό φαίνεται να δυσκολεύει κάποιους ε, εδώ στο Κοινοβούλιο. Σημαντικό για μένα στην έκθεση είναι τα πρακτικά ζητήματα. Τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον. Και για μένα είναι ιδιαίτερα σημαντικό από την ε, εκστρατεία ε, MeToo ε, να απομείνει όχι μόνο ένα hashtag, αλλά να έχουμε βοήθεια από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που να μπορούν να είναι τα προβλήματα με το όνομά τους ε, χωρίς ε, ντροπή και φόβο. Επίσης, ε, σημαντικό είναι και το οικονομικό θέμα. Θα πρέπει να έχουμε ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Προχωράμε στην διαδικασία Catch the Eye. Η κυρία Τόμασιτς είναι η πρώτη ομιλήτρια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν αναφέρεστε στο gender mainstreaming στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην σταθεί κανείς στις μαρτυρίες που έχουν υπάρξει για τη σεξουαλική καταπίεση παρενόχληση όλες ε, οι γυναίκες που έχουν πέσει θύματα θα πρέπει να ε, προστατευθούν. Δεν θα πρέπει να δώσουμε εμείς ε, στις γυναίκες την αντίληψη ότι για να προωθήσουν την καριέρα τους θα πρέπει να υφίστανται τέτοιου είδους συμβάντα. Προφανώς δεν θα πρέπει να προσλαμβάνουμε μια γυναίκα μόνο και μόνο αν είναι γυναίκα. Νομίζω ότι εγώ είχα εργαστεί παλαιότερα στις αστυνομικές δυνάμεις και είχα κερδίσει υψηλούς βαθμούς στην ιεραρχία λόγω της μεγάλης προσπάθειας την οποία είχα κάνει. Σημαίνει λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ανάγκη από βουλευτές και από προσωπικό το οποίο να είναι ειλικρινές τίμιο. Η κυρία Κούνεβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τι φαίνεται να κάνουμε σήμερα εδώ, επανάσταση. Δεν τα το λέγατε. Κι όμως, το πιο επαναστατικό πράγμα που μπορεί κανείς και καμία να κάνει είναι πάντα να διακηρυχθεί δυνατά αυτά που συμβαίνει. Το είχε πει η Ρόζα Λουξεμπούργκ Και η σημερινή έκθεση λέει δυνατά μια πραγματικότητα που η πλειοψηφία δεν φαντάζεται πώς ισχύει στο Ευρωκοινοβούλιο ανισότητα. σε πόσες θέσεις στο κοινοβούλιο είναι γυναίκες μόλις το 36% και να μην πω για φύλλα που δεν εκπροσωπούνται καν. Χρειαζόμαστε άμεσα ισόρροπη εκπροσώπηση των υποψηφίων σε εκλογές και υψηλά αξιώματα εκπαίδευση και ενημέρωση για αμερόληπτη και μη στερεοτυπική συμπεριφορά απέναντι στις γυναίκες και τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο λεπτό. Ο Θεός δημιούργησε τον άντρα και τη γυναίκα κατ' εικόνα και καθομοίωση. Δεν περιμέναμε ξένους να μας κηρύξουν την ισότητα που η αρχαία ελληνική γραμματεία και ο ελληνοορθόδοξος χριστιανισμός διδάσκει επί χιλιετίες. Είναι οξύμορο πως οι γραφειοκράτες των Βρυξελών που τόσο κόπτονται για τη διαφορετικότητα προσπαθούν να πείσουν για την απόλυτη εξίσωση και εξάλληψη κάθε φυσιολογικής διαφθοράς. Θεμελιώδη δικαιώματα και βασικοί κανόνε ειδική τάξη γίνονται όχημα πολιτική εκμετάλλευση για την προώθηση συγκεκριμένη ρητορική. Ναι στην ισότητα όχι εκμυδένιση ή κατάργηση των δύο φύλων ναι στις ίσες ευκαιρίες όχι στις θεσμικές διακρίσεις και την κωδικοποιημένη αποδοχή του ρατσισμού και του σεξισμού ναι στην αξιοκρατία όχι επιπλέον ευνοιοκρατία υπέρ ορισμένων εκλεκτών. η τυπική επίτευξη στόχων και η διαδικαστική εκπλήρωση κριτηρίων δεν αποτελεί πρόοδο. επιμένουμε για την επίτευξη πραγματικής προόδου και την εξάλληψη της εκμετάλλευσης της κακοποίησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης με λογικές και αποτελεσματικές δράσεις. ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι η ισότητα των δύο φύλων είναι ένα ζήτημα κοινωνικό και ως εκ τούτου πρέπει να υπάρξουν κοινωνικές πολιτικές προκειμένου να οδηγηθούμε στην ισότητα των δύο φύλων. φυσικά υπάρχουν και ιδεολογικές αντιλήψεις και στερεότυπα τα οποία πρέπει και αυτά να αντιμετωπιστούν. στη βάση αυτή λοιπόν πρέπει κανείς να αντιμετωπίσει το θέμα της ισότητας των δύο φύλων. θα μείνω στο ζήτημα των ψηφοδελτίων εν ώψη των ευρωεκλογών. Ε, στην ελλάδα υπάρχει η πρόβλεψη ότι τουλάχιστον το ένα τρίτο των υποψηφίων πρέπει να εκπροσωπεί ένα εκ των δύο φύλων που σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει και μεγαλύτερη εκπροσώπηση. Υπάρχει όμως στην έκθεση μια πρόταση σε περίπτωση λίστας που λέει ότι πρέπει να γίνεται εναλλαγή στη σειρά των δύο φύλων. Θα έλεγα ότι η λίστα είναι αντιδημοκρατική συμπεριφορά και αντιδημοκρατική ρύθμιση. Είναι σωστό να έχουμε την κατελάχιστον εν τρίτον εκπροσώπηση ή ουδήποτε φύλου ή και 50% αλλά από εκεί και πέρα να εκλέγεται με βάση το σύστημα του σταυρού προτίμησης όποιον προτιμούν οι ίδιοι ψηφοφόροι. επομένω να έχουμε την εκπροσώπηση την ισότιμη εκπροσώπηση των δύο φίλων στα ψηφοδέλτια και οι ίδιοι οι εκλογεί να αποφασίζουν ποιον θα εκλέξουν ω ευρωβουλευτή στι επόμενε ευρωεκλογέ. ευχαριστώ κυρία πρόεδρε για την ανοχή σα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήδη από τον προηγούμενο αιώνα η ισότητα των δύο φύλων έχει γίνει πραγματικότητα ε, και οι γυναίκες έχουν λάβει την θέση που τους αρμόζει όχι μόνο στον τομέα της εργασίας αλλά και στον τομέα της πολιτικής καθώς επίσης και στον ε, τομέα κάθε άλλης κοινωνικής δραστηριότητας. πολλές γυναίκες ακόμη και σήμερα έχουν ασκήσει και εξακολουθούν να ασκούν με μεγάλη επιτυχία υψηλού επίπεδου καθήκοντα σε επιχειρήσεις ε, διαφόρους οργανισμούς και άλλους φορείς υπενθυμίζω επίσης ότι πολλές γυναίκες υπήρξαν και εξακολουθούν να είναι ε, πρωθυπουργοί και πρόεδροι των χωρών τους. άρα λοιπόν η ισότητα υπάρχει. σε ό,τι αφορά το ευρωκοινοβούλιο και εδώ έχουμε ισότητα διότι το 55% του προσωπικού είναι γυναίκες και ό,τι αφορά το θέμα της εκπροσωπήσεως των γυναικών ε, στα ανώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας τόσο τα διοικητικά όσο και τα πολιτικά του ευρωκοινοβουλίου δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε το θέμα ως θέμα ποσοστώσεως και ως στατιστικό αλλά ως θέμα αξιοκρατίας. πρέπει να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες και τις θέσεις υψηλής ευθύνης να τις αναλαμβάνουν όσες και όσοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. εάν δεν δούμε το θέμα αυτό υπό το πρίσμα που σας ανέφερα τότε η όλη υπόθεση απλά θα καταλήξει σε έκφραση ενός ανικανοποιήτου πόθου. ευχαριστώ. Η κυρία Ward θα ήθελε να σας θέσει μια ερώτηση. Τη δέχεστε? Ερώτηση από την Julie Ward. Κυρία Πρόεδρε, όχι, απλά ήθελα ε, να αποσπάσω την προσοχή σας, διότι δεν μου δώσατε δυνατότητα να απαντήσω στη γαλάζια κάρτα από ε, τον συνάδελφο απέναντι. Ε, αυτό ήθελα και νομίζω ότι θα έπρεπε να απαντήσω, διότι ο αγώνας για τα δικαιώματα των γυναικών είναι αγώνας όλων μας και είμαι πολύ περήφανη που στην πολιτική μας ομάδα λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη το θέμα αυτό και ε, βρίσκεται στην κορυφή των εργασιών μας στην ομάδα σοσιαλιστών και δημοκρατών. Όλοι όμως όσοι ζουν στον 21ο αιώνα θα έχουν προσέξει ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι ο πιο συντηρητικός άνθρωπος που έχουμε δει εδώ και δεκαετίες και η επιρροή του στις δυνάμεις της δεξιάς σε όλον τον κόσμο ε, σημαίνει ότι ε, οι γυναίκες τελικά ε, δεν μπορούν να συνεχίσουν να προοδεύουν όσο και στο παρελθόν και έχει επαναφέρει τη, ε, τις διακρίσεις βάρος των γυναικών που είχαμε δει στο παρελθόν. Τέτοιες δυνάμεις πρέπει να καταπολεμήσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη, κυρία Πρόεδρε, που δεν σας έδωσα τα λόγια. Θα έπρεπε να σας είχα δώσει δυνατότητα να απαντήσετε νωρίτερα. Δίνω το λόγο στην Επίτροπο, την κυρία Γιούροβα. Ευχαριστώ. Ε, ξέρω ότι η Επιτροπή ε, κάνει ό,τι μπορεί, όπως κάνει και το Κοινοβούλιο. Ε, σας ευχαριστούμε λοιπόν κυρία Επίτροπε. Ευχαριστώ πρόεδρε κυρία Γιούροβα. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Η συζήτηση προχώρησε και πέρα από την έκθεση και θα υποφεληθώ και εγώ της ευκαιρίας για να μιλήσω για βασικές αρχές ε, τις οποίες ε, και η Επιτροπή επιδιώκει και εγώ προσωπικά για τα θέματα της ισότητας των φίλων. Οι ε, περισσότερε σημαντικές αρχές κατά τη γνώμη μου είναι οι ίσες ευκαιρίες. Κανείς δεν λέει ότι οι άνδρες και οι γυναίκες είναι ακριβώς ίδιοι. Μιλάμε για παροχή ίσων ευκαιριών. Μιλάμε για άρση των στερεοτύπων τα οποία εμποδίζουν τις γυναίκες να φτάσουν σε κάποιες θέσεις διευθυντικές ή διοικητικές. Και όλοι γνωρίζουμε ότι συνεχίζουν να υπάρχουν τέτοια εμπόδια. Ισότητα ευκαιριών λοιπόν ζητάμε και μηδενική ανοχή για διακριτική μεταχείριση και βία κατά των γυναικών. Υπάρχουν πολύ ανησυχητικά στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι και η διακριτική μεταχείριση και η βία είναι προβλήματα και αυτά πρέπει να επιληθούν. Και άλλη μια αρχή είναι ότι πρέπει να βοηθήσουμε τις γυναίκες να αναπτύξουν το δυναμικό τους σε όλους τους τομείς, γιατί αυτό θα είναι προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι είναι κοντόφθαλμη η στάση της κοινωνίας που δεν δίνει στις γυναίκες τη δυνατότητα να έχουν ανώτατες ε, διευθυντικές ε, θέσεις. 62% των αποφύτων πανεπιστημίου είναι γυναίκες που θέλουν να αναλάβουν ευθύνες για την ανάπτυξη της κοινωνίας μας και δεν τους δίνουμε την ευκαιρία. Όπως είπατε, ένα από τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετά καλές συνθήκες για τις εργαζόμενες μητέρες, ώστε να μπορούν να συνδυάσουν την προσωπική και επαγγελματική ζωή. Αυτές είναι λοιπόν οι βασικές αρχές ε, τις οποίες προωθεί η Επιτροπή και εγώ μέχρι το τέλος της θητείας μου και ελπίζω ότι στη συνεργασία μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ολοκληρώσουμε κάποιες από τις προσπάθειες. Καταρχήν, όσον αφορά την νομοθεσία, θέλουμε να υπάρχει σωστή ισορροπία, συνδυασμό νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλε συνθήκε, καλύτερε συνθήκε για τι εργαζόμενε γυναίκε, για του εργαζόμενου γονεί, για να έχουμε γλώσσα ουδέτερη ω προ το φύλλο, γιατί θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα και στου άνδρε να μοιράζονται τι εργασίες του σπιτιού με την ε, γυναίκα τους και να έχουν ε, ίση συμμετοχή στην ανατροφή των παιδιών και μπορούμε να συνεχίσουμε να καταπολεμούμε τις διακριτικές, τη διακριτική μεταχείριση προσπαθώντας να ενισχύσουμε τους φορείς και οργανισμούς που εκπροσωπούν τις γυναίκες ή υποστηρίζουν τις γυναίκες και μέσω της χρηματοδότησης ποικίλων προγραμμάτων προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα όπως η βία κατά των γυναικών. Βρισκόμαστε συνεχώς σε επαφή με τις διοκτικές αρχές στα κράτη-μέλη για θέματα βίας κατά των γυναικών, ενδοοικογενειακής βίας, που πρέπει να είναι προς όλους αντιληπτό ότι είναι ένα έγκλημα το οποίο πρέπει να τιμωρείται προωθούμε ε, τις αποφάσεις της ε, διάσκεψης ε, της Κωνσταντινούπολης. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε την διαφορετικότητα και είναι πολλά αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμη το έργο μας και στην επόμενη θητεία θα είναι πολύ σημαντικό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπάρχουν και άνδρες και γυναίκες που θα κατανοούν ότι δεν είναι θέμα επιλογής η ισότητα των φύλων, είναι υποχρέωση για όλους μας να προωθήσουμε τις ίσες ευκαιρίες, γιατί η έλλειψη ισότητας είναι ένα πρόβλημα όχι μόνο των γυναικών, αλλά της κοινωνίας μας γενικότερα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι οι εκλογές θα φέρουν πολλούς πεφωτισμένους βουλευτές στην ε, ε, ε, αίθουσα της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου, και από την πλευρά της Επιτροπής θα συνεχίσουμε το έργο μας και θα χαιρετίζουμε και νέες ιδέες που μπορούν να επιφέρουν εφικτά μέσα για την επίλυση του προβλήματος. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, ζητώ από την κυρία Μλινάρ να λάβει το λόγο για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ η Επιτροπή ΦΑΜΗ είναι μη νομοθετική επιτροπή. Αναφέρθηκε ότι δεν συμμετέχουν πολλοί άντρες και φαντάζομαι ότι γι' αυτό δεν συμμετέχουν πολλοί άντρες. Λυπάμαι γι' αυτό, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Η έκθεση για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου είναι επίσης ε, μη νομοθετική έκθεση. Η συζήτηση όμως ε, δείχνει πόσο έντονη είναι η σχετική συζήτηση εδώ στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους ε, και αυτούς που στηρίζουν την έκθεση και αυτούς που την ε, κατακρίνουν. Η ανοιχτή συζήτηση αποτελεί τη βάση για οποιαδήποτε δημοκρατία λειτουργεί καλά, όπως άλλωστε και η ψηφοφορία. Γι' αυτό θα ήθελα να σας καλέσω να στηρίξετε ευρέως την έκθεση αυτή για να έχουμε μια σαφή δημοκρατική απόφαση και ισχυρή δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου για ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και για ισότητα των δύο φύλων. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μλινάρ. Έτσι ολοκληρώνουμε τη συζήτηση αυτή και η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί αύριο. Εάν δεν έχετε αντίρρηση, θα προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης, έκθεση του κυρίου Μαρινέσκου. Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση για τον ΙΤΕΡ και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύνδεξης. Κύριε Μαρινέσκου, είστε εισηγήτης, έχετε τέσσερα λεπτά στη διάθεσή σας. Η ασφάλεια στην προμήθεια καυσίμων είναι κάτι το στρατηγικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις έτσι ώστε στο μέλλον να καλύψουμε με ασφάλεια τις ανάγκες μας. Και εδώ έρχεται το πρόγραμμα ITER, παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω της πυρηνικής ενέργειας, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επιδιωχθεί να υποστηριχθεί κατά τη διάρκεια του επομένου δημοσιονομικού πλαισίου σε συνεργασία και με ε, αυτούς οι οποίοι έχουν ε, πάρει μέρος μέχρι τώρα στις προσπάθειες και εκτός Ευρώπης. Έτσι θα μπορέσουμε λοιπόν να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ο οποίος θα ε, διασφαλίσει το ενεργειακό μέλλον της ε, Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Αυτά τα έξι δις για τα επόμενα χρόνια είναι μια σωστή επένδυση στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς εμείς δεν είμαστε συνομοθέτες αλλά θα στηρίξουμε και θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις για τα επόμενα χρόνια. Ε, θα πρέπει λοιπόν η αρμόδια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ατομική Ενέργεια σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους να αποτρέψει την δημιουργία καθυστερήσεων και να μην ξεπεραστεί και το προβλεπόμενο κόστος. Σας ευχαριστώ. Πρόκειται για μία πρώτη και σύντομη παρουσίαση. Παρ' όλα αυτά κάποιοι συνάδελφοι έχουν ζητήσει τον λόγο και ο κύριος Ζενονάτο και ε, μετά θα ακολουθήσουν άλλοι δύο και στο τέλος ο κύριος Μαριάς. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρινέσκου γιατί νομίζω ότι πολλά από αυτά τα οποία είπε με βρίσκουν σύμφωνο και μετά από την ψηφοφορία στην Ήτρε βλέπω ότι πολλές από τις τροπολογίες που είχα καταθέσει συμπεριλαμβάνονται. Η σωστή χρηματοδότηση του Ίτερ έχει μεγάλη σημασία, είναι ένα από τα πιο έγκυρα πειράματα για την χρήση αυτής της μορφής σύνδεξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει πρωτοπόρο ρόλο σε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ε, και συμβολικό ρόλο ε, στο Κανταράς ε, σημαντικές χώρες που εκπροσωπούν πάνω από το 50% του πληθυσμού συμμετέχουν στις εργασίες, τις πειραματικές. Αυτά όλα διευκρινίζονται λοιπόν στο κείμενο το οποίο θα ψηφίσουμε. Θα πρέπει η οργάνωση αυτή να εξορθολογιστεί ε, διαχειριστικά θα πρέπει να μην αποκλίνει από τους στόχους και θα πρέπει να αποφύγουμε τις αυξήσεις του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο. For the floor. course. Thank you very much. Ε, το πρόγραμμα ITER, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση για την Ανάπτυξη Πυρηνικής Σύνδεξης, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πούμε ότι αυτή τη στιγμή όπως αναφέρθηκε συνεργάζονται πολύ σημαντικά μη ευρωπαϊκά κράτη όπως είναι οι ηνωμένες πολιτείες η ρωσία η ιαπωνία η κίνα η νότια κορέα και η ινδία. βεβαίως η ευρωπαϊκή ένωση παίζει ένα σημαντικό ρόλο ε, που αυτό δείχνει ότι η επένδυση στην οικονομία της γνώσης είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό φυσικά θα πρέπει να προσέξουμε να μην ξεφύγει ο προπολογισμό. γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολες οι διαδικασίες και όλο το πείραμα ξέρουμε ότι πολλές φορές υπάρχουν αρκετά προβλήματα αλλά στη βάση του ότι μπορούμε πραγματικά να επιμείνουμε σε αυτό το πρόγραμμα και κυρίως με έναν τρόπο που να μην ξεφύγει οικονομικά αλλά να συμβάλλει ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της ίδιας της τεχνολογίας θα είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό και στο πλαίσιο αυτό θα έλεγα ότι ορισμένες πλευρές αυτού του προγράμματος χρηματοδότηση θα μπορούσε να δοθεί και σε ελληνικά ερευνητικά κέντρα σε πανεπιστήμια ούτως ώστε και αυτά να συμβάλλουν σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Ευχαριστώ. Ε, Κοιτάξτε, ε, σε σχέση με αυτά τα οποία ελέγχθησαν, εγώ κάπως διαφωνώ, διότι αυτό το σχέδιο, το ITER, δεν είναι το σωστό, διότι είναι καθυστερημένο, έχει καθυστερήσει πολύ. Διότι για να επιληθούν τα προβλήματα της υπερθέρμανσης του κλίματος, θα πρέπει να μπορούμε να παράγουμε ε, ηλεκτρισμό πριν από το 2050 χωρίς εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Το έργο ITER έχει καθυστερήσει πάρα πολύ και το πρώτο πρωτότυπο δεν θα φτάσει πριν από το 2050. Επομένως, δαπανούμε πάρα πολλά χρήματα για ένα έργο το οποίο θα καθυστερήσει πάρα πολύ. Εξαιρετικά πολλά χρήματα, διότι στην αρχή μας είπαν 5 δις για το ITER. Τώρα είμαστε στα 20 δις. Και όταν ε, είχα δει ε, το Αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας, αξιολογούσε το κόστος του ΙΤΕ στα 65 δις μαζί με τη λειτουργία του. Ε, υπερβολικά μεγάλο λοιπόν. Και δυσανάλογο αυτό το έργο. Είναι πολύ κεντρικοποιημένο με πάρα πολλά τεχνικά προβλήματα. Θα βάλουμε τον ήλιο μέσα σε ένα κουτί και το κουτί δεν μπορούμε να το κατασκευάσουμε. Και όπως έλεγε και ο συνάδελφος Μαρινέσκου, για αυτό το έργο θέλουμε να έχουμε δημοκρατικές εγγύησεις και εμείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει δυνατότητα συναπόφασης, συναποφασίζει η Ευρατόμ. Κατά τη γνώμη μου δεν επιφέρει και τη λύση που θέλουμε για τα προβλήματα του κλίματος. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πόλτσακ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι η πυρηνική ενέργεια αποτελεί εναλλακτική λύση χαμηλών εκπομπών υψηδίου του άνθρακα σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα και επίσης συμβάλλει σε ένα καλό ενεργειακό μείγμα. Αποτελεί την πηγή του 30% σχεδόν της ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΙΕ έχει δημοσιεύσει έκθεση υπέρ της πυρηνικής ενέργειας για την προστασία του περιβάλλοντος, προτού να είναι πολύ αργά. Η έκθεση λέει ότι η πυρηνική ενέργεια έχει να παίξει ρόλο κλειδί. Φυσικά μιλάμε για ένα σχέδιο που ε, παρουσιάζει κάποια προβλήματα. Θα πρέπει να καλυφθεί το κόστος Μπορεί όμως να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προόδου και να μας βοηθήσει να πετύχουμε και τους στόχους του Παρισιού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χάουερ έχει το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για μια πολύ καλή και λογική έκθεση. Ωστόσο, ο ελέφαντας στο δωμάτιο, το προφανές θέμα που δεν αναφέρεται είναι ο ρόλος του Ηνωμένου Βασιλείου. Βέβαια, όλα αυτά εξαρτώνται από το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο. Δυστυχώς, η Πρωθυπουργό η κυρία Μέη, τα έχει κάνει άνω κάτω. Ε, είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να αποχωρήσει από την συνθήκη Ευρατών. Η δική μου εκλογική περιφέρεια είναι ο μόνος τόπος που έχει πετύχει την πυρηνική σύνδεξη, είναι πηγή εμπειρογνωσίας και χωρίς τη στήριξη ε, της ε, Ευρώπης ε, θα δούμε περισσότερα προβλήματα. Μάλιστα, ε, πριν ε, το Brexit είχε ανακοινωθεί η επέκταση του σχεδίου αυτού με τη δημιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης. Ε, ελπίζω να έχουμε επιτυχία τελικά στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Όπως είπα πριν λίγο, ο κύριος Χάουερθ ήταν ο τελευταίος ομιλητής. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Γιούροβα στο όνομα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Εάν θέλετε να πάρετε το λόγο. Ναι, θέλω να πάρω το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, σα ευχαριστώ πολύ για την επικοδομητική συζήτηση σήμερα. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Μαρινέσκου, για την έκθεσή του και την έκκληση προ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να υπερψηφίσει την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συνεχιζόμενη χρηματοδότηση ε, του ΙΤΕΡ στο επόμενο χρηματοδοτικό διάστημα. Όπω πάντα, η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σημαντική για να πετύχουμε ε, ευρωπαϊκή στήριξη στο σημαντικό αυτό έργο. Ο ενεργειακό μετασχηματισμό και η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματο αποτελούν ε, τι βασικέ προκλήσει που αντιμετωπίζουμε σήμερα και γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε μια φιλική προ το περιβάλλον ε, πηγή ενέργεια με χαμηλέ εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα όπως είναι η πυρηνική σύνδεξη. Ε, είναι πολλά υποσχόμενη αυτή η πηγή ενέργειας. Το ΙΤΕΡ σε παγκόσμιο επίπεδο ε, συγκεντρώνει την καλύτερη εμπειρογνωσία από όλο τον κόσμο και στοχεύει σε σημαντικά βήματα προόδου ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια ανεξάρτητη πηγή ενέργειας που θα στηρίξει τις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Ένωση για καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Ε, τα ωφέλη θα είναι σημαντικά και για την οικονομία και για την κοινωνία. Θα επιτρέψει στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και τους ερευνητές να εισέλθουν σε νέε αγορέ. Υπόσχεται πολλά και για την εκπλήρωση των άλλων πτυχών της ενεργειακής μας ένωσης. Να έχουμε ασφαλή ενέργεια για τους πολίτες μας ε, και ε, δημιουργία θέσεων εργασίας. Θέλουμε να ε, θέλουμε να διασφαλίσουμε την ηγετική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα της, της πυρηνικής σύνδεξης. Χάρη στην κατασκευή του ίτερ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να απολαύσει τα, τους καρπούς και η έκθεση αυτή δημοσιεύεται σε πολύ σημαντική στιγμή για το ίτερ. Τα τελευταία χρόνια είδαμε σημαντικές βελτιώσεις στην διεύθυνση του ίτερ και η και το έργο που ε, χρειάστηκε να κατασκευαστεί για να γίνουν τα πειράματα έχει ολοκληρωθεί κατά 60%. Ε, πιστεύουμε ότι τα πρώτα πειράματα θα μπορούν να γίνουν το 2022. Και για να απαντήσω στην κυρία Ρίβαζη, είναι αλήθεια ότι η πυρηνική σύνδεξη δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί εμπορικά πριν το δεύτερο μισό του αιώνα και γι' αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στις στρατηγικές μας για μετριασμό ε, της αλλαγής του κλίματος ε, μέχρι το 2020. Ε, οι στόχοι μας όμως είναι μακροπρόθεσμοι και θα χρειαστούμε βιώσιμες λύσεις και για μετά το 2050. Και γι' αυτό η πυρηνική σύνδεξη παρέχει μια πολύ ελκυστική λύση για το δεύτερο μισό του αιώνα, τότε που η σύνδεξη θα μπορέσει να συμπληρώσει τις βιώσιμες πηγές ενέργειας. Θα έχουμε έτσι κάψιμα χαμηλού κόστους και ε, με ε, περιορισμένο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Όλοι οι διεθνείς παράγοντες που συμμετέχουν στον ΙΤΕΡ ε, εργάζονται σκληρά για να μπορούν να ακολουθήσουν το, το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα που εκπονήθηκε το 2016. Η συνεχιζόμενη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, καθώς και το ε, επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα αποτελέσουν σημαντικά στάδια στο έργο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Bonsoir, mes chers collègues. Le débat σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Τελειώνει αυτή η συζήτηση και η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί αύριο. Ε, ε, ε, Προχωράμε στην έκθεση του κυρίου Χέις, δεν τον βλέπω όμως. Θα περιμένουμε λοιπόν λίγο. Μικρό διάλειμμα. Κοιτάξτε, είναι κάπω ενοχλητικό. Πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό. Η συγγετή λείπει. Ε, έχουμε αυτό τα θέματα, τα σύντομε παρουσιάσεις. Θα ξεκινήσουμε με όσους ζήτησαν να συμμετέχουν στο Catch the Eye. Να ακούσουμε την κυρία Γιούρεβερ, λυπούμε για τον κύριο Χέις. Ίσως και να έρθει, αλλά εάν δεν έχετε πρόβλημα να δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο ε, Πόλτσακ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι μάλλον ασυνήθις αυτή η διαδικασία, αλλά εν πάση περιπτώσει να σας πω κι εγώ πως στην Τσεχία γίνονται μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα και αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προχωρήσουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Να σας πω πως οι ευρωπαϊκοί πολιτικές δεν θα πρέπει να υποκαταστήσουν την εθνική χρηματοδότηση, τουλάχιστον όχι στο 100%, θα πρέπει να είναι μια επιπρόσθετη πηγή χρηματοδότησης και αυτά τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά θα πρέπει βέβαια να προσανατολίζονται προς αυτά αποτελέσματα και να δούμε και ποια θα είναι οι θετικές επιπτώσεις ε, έτσι ώστε να γίνουν οι σωστές μεταρρυθμίσεις ε, στα εν λόγω κράτη-μέλη. Οπότε, να δούμε και την ποιότητα των μεταρρυθμίσεων και όχι μόνο το πώς θα χρηματοδοτούνται αυτές. Αυτά μπορώ να πω γιατί δεν έχω ακούσει βέβαια τι θα μας έλεγε η και δεν ήταν και άσχημα αυτά που είπατε, αρκετά καλά είπατε και ήταν ε, πραγματικά εντυπωσιακό. Πρώτη φορά μας συμβαίνει. Ε, να σας επαναλάβω ότι, γιατί δεν είχα προλάβει να πω το τύπο, ότι έχουμε να κάνουμε με την έκθεση που έχει να κάνει για την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, την έκθεση Hayes. Η ευχαριστώ τον συνάδελφο Ευχαριστώ συνάδελφο Χέιζη και τους ε, συναδέλφους Σκιώδης. Ε, όπως μας θυμίζει η Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι πολίτες έχουν δικαίωμα σε μια ε, <clears throat> σωστή ε, σε ένα σωστό διοικητικό μηχανισμό. Είναι σημαντικό λοιπόν να εγγυηθούμε τον καλύτερο δυνατό συντονισμό των πόρων που προβλέπει ο Ευρωπαϊκό προπολογισμό ε, για να στηρίξει τη ε, διοικητική διακυβέρνηση των κρατών μελών. Και αυτό σημαίνει υπηρεσίε και εγγύηση τη της εφαρμογή εφαρμογής των ευρωπαϊκών πολιτικών για την αλληλεγγύη και την ανάπτυξη. θεωρώ πω είναι πολύ σημαντική η πρόθεση τη ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη σχέση μεταξύ διοίκηση και πολίτη, η εφαρμογή της πληροφορικής και της τηλεματικής μπορεί να συμβάλλει όχι μόνο στη μείωση των σπαταλών, αλλά και να καταστήσει πιο εύκολη, άμεση και διαφανή την πρόσβαση των εταιρεών και των πολιτών στις υπηρεσίες και στις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να επισημάνω ότι οι μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση των κρατών μελών είναι αρμοδιότητα των ίδιων των κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Ένωση επ' αυτού δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Και το λέω αυτό διότι η Τρόικα όλα αυτά τα οκτώ χρόνια στην Ελλάδα επέβαλε βίαιες μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα, παρεμβαίνοντας σε περιοχές στις οποίες δεν είχε καμιά αρμοδιότητα. Και όλα αυτά εκβιάζοντας την ελληνική κυβέρνηση ότι δεν θα έδινε δάνεια σε σχέση βεβαίως με τα εννέα δισεκατομμύρια τα οποία δίνει η ευρωπαϊκή ένωση για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα νομίζω ότι πρέπει αυτά να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο να μην αποτελούν άλοθη για να παρεμβαίνει με επιλογές δικές της η ευρωπαϊκή ένωση και κυρίως οι βρυξέλλες να δοθεί μεγάλη έμφαση ιδίως σε θέματα αξιοποίησης νέων τεχνολογιών να περιλάβει όχι μόνο την κεντρική διοίκηση αλλά επίσης και την τοπική αυτοδιοίκηση να έχουμε σημαντικό ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων και να έχουμε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αξιοποιήσουν τις, ε, τα προσβάσιμα κονδύλια. Κάποια κράτη-μέλη είναι καλύτερα σε αυτό από ό,τι άλλα. Αλλά είμαστε ειλικρινεί, δεν υπάρχει κάποια συνωμοσία. Είναι σφάλμα και ευθύνη των κρατών μελών αν δεν είναι ικανά να απορροφήσουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δική μας δουλειά είναι να εντοπίσουμε τα σφάλματα, τις παραλήψεις και να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη που έχουν συλλέξει ε, και αποκομίσει αρνητικέ ε, εμπειρίε, προκειμένου οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσουν το πλήρε δυναμικό τη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Πρέπει να σα πω ότι η εμπειρία τη της Κροατία δείχνει ότι η απλούστευση των διαδικασιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Συνοχής και άλλων ταμείων μπορούν να ε, μπορεί να βελτιώσουν δραματικά την κατάσταση. Είναι σημαντικό τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να είναι πιο οργανωμένα και πιο επαγγελματικά στον, στον, στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η κυρία Γιούροβα να το λόγο παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρωτοβουλία σας, ε, για αυτό το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τον ε, τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται ε, τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τον δημόσιο τομέα. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαιρετίζω την πρωτοβουλία σας αυτή. Συμφωνώ με την ανάλυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η δημόσια διοίκηση στα κράτη-μέλη αποτελεί ε, ύψιστη σημασία στοιχείο για την εφαρμογή του και την εκτέλεση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και όταν είναι αποτελεσματική μπορεί να συμβάλλει στην ύπαρξη αποτελεσματικών συστημάτων που μπορούν να συνεισφέρουν στην ευημερία και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνούμε επίσης όσον αφορά τη σημασία για τον, την ανταλλαγή εμπειρίας, ε, εμπειριών και γνώσεων μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε ήδη αναγνωρίσει διάφορες προτάσεις που έχετε εντάξει στην ε, πρόταση ψηφίσματός σας και θα τις ε, παρακολουθήσουμε. Για παράδειγμα, μια υποστηρικτική υπηρεσία η οποία θα προσφέρει βοήθεια στις εθνικές διοικήσεις. Εμείς θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα των δικών μας εργασιών. Επίσης, η υπηρεσία αυτή θα συντάξει κάποιους συγκριτικούς δείκτες για την ανταλλαγή πληροφοριών, βέλτιση των πρακτικών και για την ενίσχυση ενός στενότερου διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται και θα συνεχίσει να χειρίζεται μια σειρά από τεχνικές δραστηριότητες και έργα μεταρρύθμισης στον τομέα της διοίκησης ε, και της διακυβέρνησης. Ιδιαίτερη ε, στήριξη παρέχεται και υπό την πολιτική συνοχή ε, για την καλύτερη απορρόφηση και αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Επενδυτικών Ταμείων και Ταμείων Συνοχής. Θεωρώ ότι έχουμε τις ίδιες, ε, τους ίδιους στόχους και με το Κοινοβούλιο και με τα κράτη-μέλη προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη ε, μιας σύγχρονης και ποιοτική δημόσιας διοίκησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει έρθει ο κύριος Χάρης, λυπάμαι πολύ. Εν περιπτώσει κλείνει εδώ η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Θα μπορέσουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την επόμενη ε, με το επόμενο σημείο που είναι οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντολή του ειδικού αποστελμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της θρησκευτική ελευθερίας και της ελευθερίας των πεπιθήσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Γκρίπς, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες και όλους τους σκιώδεις εισηγητές για την υποστήριξη που μου προσέφεραν στην πρωτοβουλία μου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ανάγκη να δραστηριοποιείται για την θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεπιθήσεων. Και θέλω να ασχοληθώ και να τοποθετηθώ για αυτό το θέμα. Πρέπει να πούμε ότι στον 21ο αιώνα η ελευθερία της, ε, ε, των θρησκευτικών πεπιθήσεων και εν γέννη των πεπιθήσεων αντιμετωπίζει μια δραματική κατάσταση σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουμε να κάνουμε με μια δραματική επιδείνωση ε, της κατάστασης στον κόσμο. Εδώ και πέντε χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει τις συστάσεις της για τα θέματα αυτά. Το 2013 εγκρίθηκαν οι σχετικές ε, συστάσεις. Ο κ. Αντριουκένε ε, είχε μάλιστα προετοιμάσει τις συστάσεις αυτές για να εγκριθούν από το Συμβούλιο. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι το εξής ένας ειδικό απεσταλμένο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης για την προώθηση της θρησκευτική ελευθερίας και της ελευθερίας των πεπιθήσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πρωτοβουλία του ίδιου του κυρίου Γιούγκερ έπειτα από ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2017 από την, την, ε, καθώς ε, εορτάζουμε την 70η ε, επέτειο της διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει τον ορισμό του άρθρου 18 της διακήρυξης αυτής που αφορά την θρησκευτική ελευθερία. Και εδώ πρέπει ως συνομοθέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τοποθετηθούμε. Έχει 10 χρόνια από τότε που εγκρίθηκε η Συνθήκη της Λισαβόνας. Και στην ε, Συνθήκη της Λισαβόνας κατοχυρώνεται η υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνει δράση σε ολόκληρο τον κόσμο για την προώθηση των αρχών της, μεταξύ των οποίων είναι και η θρησκευτική ελευθερία. Θεωρώ λοιπόν ότι οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να λάβουν έναν πιο, πιο συστηματικό χαρακτήρα και συγκεκριμένα εδώ ε, θέλω να αναφερθώ σε δύο ε, περιπτώσεις. Έχουμε την περίπτωση της Πακιστανής χριστιανή, χριστιανής, την Αζέρα Μπίμπη, η οποία ε, καταδικάστηκε σε θάνατο ε, για βλασφημία. Ευτυχώ η απόφαση αυτή έχει ανακληθεί, αλλά πρέπει να εξασφαλιστεί η προστασία της ζωής της και της οικογένειάς της. Επίσης έχουμε τον κύριο Χαντάφη, ο οποίος πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος, διότι κρατείται ακόμα στη φυλακή για ε, παρόμοια αδικήματα. Πρέπει όλοι λοιπόν να καταβάλουμε προσπάθειες για την προώθηση της θρησκευτική ελευθερίας και της ελευθερίας των πεπιθήσεων, ώστε οι αρχές αυτές να εξασφαλιστούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Θέλω να ξανατονίσω τη θρησκευτική ελευθερία και η ελευθερία των πεπιθήσεων. Είναι ζητήματα που πρέπει να εξασφαλίζονται με όλους τους εταίρους μας. Αν δείτε τα στατιστικά δεδομένα, οι πληθυσμιακές ομάδες, ε, η, ε, η κατηγορία του πληθυσμού που αντιμετωπίζει τις περισσότερες διώξεις είναι οι χριστιανοί. Μιλάμε για μαζικές σφαγές κατά χριστιανών σε ολόκληρο τον κόσμο. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχουμε ε, εγκρίνει τις συστάσεις οποίες αναφέρθηκα στην αρχή της τοποθέτησής μου. Γνωρίζουμε τη σημασία που έχει η υπόθεση αυτή του ειδικού απασταλμένου. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε έκκληση προς το Συμβουλίο και την Κομισιόν να ξαναδώσουν πνοή σε αυτή την πρωτοβουλία και να ενισχύσουν την κατάρτιση, της επενδύσεις στους θεσμούς, στα κράτη-μέλη. Θέλουμε για το σκοπό αυτό να εξασφαλίζεται και χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι και πέραν των ευρωπαϊκών κονδυλίων μπορούν αντίστοιχα έργα, αντίστοιχες πρωτοβουλίες να χρηματοδοτούνται και ε, από άλλες πηγές. Θέλουμε να υπάρχει συγκεκριμένη γραμμή χρηματοδότησης και στο πολιτές δημοσιονομικό ε, πλαίσιο. Σε λίγες μέρες γιορτάζουμε και την Παγκόσμια ημέρα ε, των θυμάτων των, ε, ε, της βίας κατά της θρησκευτικής ελευθερίας. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει σε αυτήν την πρωτοβουλία, σε αυτούς τους εορτασμούς. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάτσε the λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτή τη διαδικασία. Ο κύριος Φαρία, ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η αρχή διαχωρισμού μεταξύ κράτους και εκκλησία είναι μια αρχή οργάνωσης οποιοδήποτε δημοκρατικού κράτους που σημαίνει ότι δεν μπορεί να παρεμβαίνει η θρησκευτική αρχή στη λειτουργία των δημόσιων ε, ε, αρχών και τούμπαλιν. Είναι αξίες αυτές βασικές, καθολικές, δεν μπορούμε να τις εγκαταλείψουμε. Είναι η ουσία των όσων εμείς εκπροσωπούμε, ελεύθερη, δίκαιη, ε, δημοκρατική Ευρώπη. Προβλέπετε δε το βραβείο Ζαχάροφ για τα θύματα της ε, έλλειψης ανεξιθρησκείας. Είδαμε την άνοδο το θρησκευτικό εξεμισμό τα τελευταία χρόνια και σε αυτό προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντισταθεί με τα διάφορα αυτά σχέδια. Η δημιουργία της θέσης του ειδικού απεσταλμένου για την προώθηση της ανεξισυρισκίας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούμε πως είναι ένα πολύ μια πολύ σωστή πρόταση από πλευρά της Κομισιόν αναγνωρίζεται η ανεξιθρησκεία σε αντίθεση με τον φονταμεταλισμό. Κύριος Μαριάς. Κύριε Πρόεδρε, η θρησκευτική ελευθερία και η ελευθερία των πεπιθήσεων πρέπει να προστατεύονται τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, ο Μηχανισμός Αναπτυξιακής Συνεργασίας, ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας πρέπει να δίδονται υπό τον όρο ότι τα κράτη που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και παίρνουν αυτές τις χρηματοδοτήσεις θα τηρούν την αρχή της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεπιθήσεων. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει με την περίπτωση της Αλβανίας, όπου καταπιέζονται τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας της Βορείου Υπήρου, όπου δεν τους επιτρέπουν να ασκήσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, όπου γκρεμίζονται οι εκκλησίες, όπως ήταν η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου σημαίνει λοιπόν ότι η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να σταματήσει κάθε χρηματοδότηση προς την αλβανία μέχρι ότου να τηρήσει και να σεβαστεί τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας της βορείου ηπείρου. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κάθε άτομο έχει δικαίωμα να διαλέγει τι θα πιστεύει ή αν θα πιστεύει. Και αυτό το δικαίωμα πρέπει να προστατεύεται μέσω των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφενός χαιρόμαστε που όλες οι διαστάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεπιθήσεων αντικατοπτρίζονται στην τελική έκθεση, όχι μόνο η θρησκευτική ελευθερία αλλά και η ελευθερία της συνείδησης και των πεπιθήσεων. Επίσης χαιρόμαστε για τις αναφορές για, τις, ε, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άθεοι καθώς και τα προβλήματα που αντιμετώπιζουν πολλοί άνθρωποι ε, σε σχέση με την αποστασία τους, με την αποχώρησή τους από κάποιο συγκεκριμένο δόγμα. Αφετέρου, θέλουμε ε, να εξασφαλιστεί και το η δυνατότητα των ατόμων να, εκφράζουν, να εκφράζονται σατυρικά ή καλλιτεχνικά εναντίον ε, συγκεκριμένων θρησκειών. Κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται στην έκθεση. Και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να, του οποίου πρέπει να επιληφθεί ο ειδικό απεσταλμένο για να εξασφαλιστεί ότι η θρησκευτική ελευθερία θα ενταχθεί οργανικά στην πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Thank you. It was yesterday that... Ευχαριστώ, κύριε Σούγκο. Χθε ήταν 451η επέτειος της ε, διακήρυξης θρησκευτική ελευθερίας στην Τρασιλβανία. Ήταν η πρώτη τέτοια πράξη και αποτέλεσε το πρώτο εναρκτήριο έναυσμα μιας ε, μακραίωνης διαδικασίας. Δυστυχώς η κατάσταση δεν είναι καλύτερη σήμερα. Πάνω από 70% του παγκόσμιου πληθυσμού ε, πλήττεται από κυρώσει τι οποίε υφίσταται λόγω παραβιάσεων θρησκευτική ελευθερία. Και βλέπουμε και πολλέ ε, εκδηλώσει θρησκευτικού φονταμενταλισμού. Και αυτό, αυτό αιτιολογεί την ε, θέσπιση αυτή τη θέση του ειδικού επισταλμένου με σκοπό την προώθηση τη θρησκευτική ελευθερία στον κόσμο. Θα είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική η οποία θα βοηθήσει και την καλύτερη δικτύωση με άλλους είναι σημαντικό να καθοδηγήσουμε αυτή τη διαδικασία θρησκευτική ελευθερία και ελευθερία των πεπιθήσεων ώστε να προωθηθούν αυτέ οι αρχέ σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω των εξωτερικών πολιτικών μα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει για άλλη μια φορά να αποτελέσει πρωτοπόρο σε αυτόν τον τομέα όπω το έκανε και πριν από 500 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να χαιρετήσω αυτή την πρωτοβουλία του κύριου Ξύπ. Τον γνωρίζω και ξέρω ότι ψυχείται και σώματι έχει δοθεί σε αυτήν την υπόθεση για την προώθηση θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεπιθήσεων. Όμως, να μιλήσουμε για τη συγκεκριμένη έκθεση. Αυτή η έκθεση δυστυχώς ε, περιλαμβάνει όλα τα, ε, τα ίχνη που έχουν εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να συντάξουν εκθέσεις χωρίς να έρχονται σε αντίθεση με την, ε, με την επίσημη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε, καμία, ε, σε κανένα σημείο της ε, έκθεσης αυτής δεν μπορεί κανείς να βρει ούτε καν τον όρο χριστιανοσύνη. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι, είναι μια Ήπειρος χριστιανική. Ευχαριστώ. Πριν να δώσω το λόγο να σας πω ότι δεν σας ακούω πολύ καλά τα γαλλικά. Ο κύριος Πόλτσεκ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να επενέσω την έκθεση του κυρίου Γκζίμπ είναι εξαιρετική ποιότητα. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μιλάμε για την αρχή της ε, ισότητας μεταξύ πιστών και απίστων. Ε, επίσης είναι πολύ ατυχές ε, να βλέπουμε την ευρωπαϊκή πολιτική η οποία συχνά δεν κάνει διακρίσεις γιατί δίνουμε ευρωπαϊκή βοήθεια ακόμα και σε χώρες οι οποίες διώκουν τους χριστιανούς και αυτό είναι ε, λάθος. Από την άλλη πλευρά, η ιδέα θέσπισης ενός ειδικού απεσταλμένου υπέρ της ανεξιθρησκείας είναι ε, σωστή, τη στηρίζω. Η θρησκεία κάποιες φορές οδηγεί στα άκρα, σε ολόκληρο τον κόσμο, είτε μέσω της δίωξης των πιστών, είτε μέσω της χρήσης της θρησκείας ως πολιτικού ε, όπλου. Θα πρέπει να προβλέψουμε εγγυήσεις για την ανεξιθρησκεία. Ευχαριστώ. Κυρία Σέντροβα, ξέρετε πώς Το να έχουμε αυτό τον ειδικό αποσταλμένο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα πολύ θετικό βήμα και μια εξαιρετική απόφαση. Και είναι πολύ ε, σημαντικό πως ο πρώτος που ανέλαβε αυτή τη θέση από το 2016 είναι χριστιανοδημοκράτης από τη Σλοβακία. Και ήταν ο άνθρωπος αυτός ο οποίος μαζί με τους Τσέχους διπλωμάτες διαπραγματεύτηκε την απελευθέρωση του Πίτερ Γιάσεκ που είχε καταδικαστεί σε 20 ετή φυλάκιση ε, γιατί τεκμηρίωσε την δίωξη χριστιανών στο Σουδάν. Ο άνθρωπος αυτός απελευθερώθηκε ακριβώς μετά από πρωτοβουλία που ανέλαβαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και οι τσεχικές διπλωματικές αρχές. Υπάρχουν εκατομμύρια τέτοιοι άνθρωποι και θα πρέπει να προστατευτούν. Ευχαριστώ πολύ. Η, ιστορία παραλαμβάνεται, θα πρέπει να αισθάνονται δικαιωμένοι. Μετά 18 αιώνες, αφού το έληξαν οι διωγμοί εναντίον των χριστιανών, αυτοί δυστυχώς επαναλαμβάνονται στη σημερινή εποχή από διάφορα κράτη της μέσης ανατολής της ασίας της αφρικής. χριστιανοί διώκονται για την πίστη τους και περισσότερο από 215 εκατομμύρια έχουν υποστεί κάθε είδους ταπεινώσεις και διωγμούς. Ακόμη και σήμερα δυστυχώς υπάρχουν γυναίκες και κορίτσια που υποφέρουν σεξουαλικά για την πίστη τους στον Ιησού Χριστό στην ελλάδα η οποία έχει το 95% του πληθυσμού ορθοδόξους χριστιανούς έχουν σημειωθεί περισσότερα από 556 ε, περιστατικά επιθέσεων εναντίον των θρησκευτικών τόπων, των τόπων δηλαδή ε, προσευχής. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το φαινόμενο να το πατάξει και να μην χρηματοδοτεί χώρες οι οποίες καταπιέζουν τις θρησκευτικές ναι, ελευθερίες και να μην δέχεται στην, ε, στην ε, ε, ένταξη, προς ένταξη χώρες όπως η Αλβανία που παραβιάζει τα θρησκευτικά δικαιώματα. E, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η θέσπιση θέσης ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θρησκευτική ελευθερία ήταν πρωτοβουλία του Ζαν κλοντ Juncker. Η πρωτοβουλία αυτή χαιρετίστηκε όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού. Ο Γιάνν Φιγγέλ έχει επιτελέσει πολύ σημαντικό έργο και έχει αποδείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο πλευρό εκείνων των οποίων η θρησκευτική ελευθερία δεν εξασφαλίζεται και δεν προστατεύεται. Το έργο του Γιάνν Φιγγέλ είχε και μια θετική επίδραση στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η συνείδηση που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες γύρω από τα ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας. Και ελπίζω και η εξωτερική πολιτική μας να επηρεαστεί εξίσου. Έχω μια ερώτηση για την κυρία Γιούροβα. Πώς σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει τον ρόλο αυτού του ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεπιθήσεων. Κυρία Γιούροβα, έχετε το λόγο για να απαντήσετε στον κύριο Πέτρελε. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γκζιπ, τον εισηγητή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στον τομέα αυτής της έκθεσης. Συμμεριζόμαστε και προσυπογράφουμε το, το περιεχόμενό της και τονίζουμε και εμείς τη σημασία που έχουν η θρησκευτική, η θρησκευτική ελευθερία και η ελευθερία των πεπιθήσεων. Όπως τονίζει η έκθεση, είναι αρχές οι οποίες ε, δέχονται πλήγματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Άνθρωποι όλων των ε, θρησκευτικών πεπιθήσεων διώκονται εξαιτία ακριβώς αυτών των πεπιθήσεών τους. Οι διακρίσεις λοιπόν στη βάση των θρησκευτικών πεπιθήσεων ε, είναι ένα ε, εξαιρετικά διευρυμένο ε, φαινόμενο καθώς και η νομοθεσία για την αποστασία που ποινικοποιεί την θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεπιθήσεων. Όπως είπατε και εσείς, πρόκειται στην ουσία για παραβιάσεις των, ανθρωπι... των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στην Γενική Διακήρυξη που εγκρίθηκε πριν από πάνω από 70 χρόνια. Δεν μπορεί η θρησκευτική συνείδηση ούτε να επιβληθεί ούτε και να απογορευτεί. Η έκθεση επίσης τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η αντοχή, η ανθεκτικότητα των κοινωνιών. Για τους λόγους αυτούς, ε, στο παρελθόν έχουμε εκφράσει τις ανησυχίες μας σχετικά με τις παραβιάσεις των θρησκευτικών ελευθεριών σε πάνω από 20 σχετικούς διαλόγους με χώρες από τη Μεσσηνή Ατολή, τη Βόρεια Αφρική, αλλά και με διάφορες ασιατικές χώρες. Τόσο ε, ο ειδικός απεστηλμένος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για, τη, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο ειδικός απεσταλμένος για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεπιθήσεων ε, προωθούν τα δικαιώματα αυτά σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουν πραγματοποιήσει πολλές αποστολές και έχουν έρθει σε επαφές με θρησκευτικούς ηγέτες και κυβερνήσεις. Θέλω να τονίσω την πολυδιάστατη διάσταση, την πολυδιάσταση, τον πολυδιάστατο χαρακτήρα των εργασιών μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να, τις προσπάθειές μας στο πλαίσιο του ΟΗΕ και να ενισχύσουμε την ε, δραστηριοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το 2019 θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, σε όλους τους διαλόγους μας. Τονίζουμε ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αλληλένδετα και η θρησκευτική ελευθερία και η ελευθερία των πεπιθήσεων πρέπει να συμβαδίζουν με την με την ελευθερία του συνέρχεσαι, τους, του, της ε, ελευθερίας έκφρασης αλλά και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ. Η έκθεση ε, καλεί να υπάρξει ισχυρότερη θεσμική συνεργασία και από το 2013 και την έγκριση των συστάσεων αυτός είναι γενικός και μόνιμο στόχο μας. Και ο καλύτερος τρόπος για να ενισχυθεί ο συντονισμός και ο διάλογος είναι να υπάρξει καλύτερη επαγρύπνηση γύρω από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Όπως λέει και η έκθεση, προκειμένου να ε, επιτύχουμε τους στόχους μας, έχουμε πολλαπλασιάσει την κατάρτιση για το προσωπικό, για το προσωπικό μας τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στις αποστολές. Και σύμφωνα και με τις συστάσεις της έκθεσης, θα συνεχίσουμε να δραστηριοποιούμαστε και να ερχόμαστε σε επαφές με ε, οργανώσεις, θρησκευτικού ηγέτες, οργανώσεις των αθέων και ε, ε, ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δυστυχώς η κατάσταση δεν είναι ρόδινη. Ωστόσο, βλέπουμε ε, ότι υπάρχουν σημάδια ελπίδας. Για παράδειγμα, το 2018 είδαμε κάποιους υπερασπιστές τις ε, των, της να απελευθερώνονται από, την, από τις φυλακές. Στην Αφρική έχουν ξεκινήσει διάλογοι συμφιλίωσης και καθώς ε, προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τις παραβιάσεις αυτών των ελευθεριών θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε και να στηρίζουμε τέτοιες κινήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Η συζήτηση έκλεισε και θα ψηφίσουμε αύριο. Περνάμε λοιπόν στην, στο επόμενο θέμα στην επόμενη ε, έκθεση είναι η έκθεση Ματίας και Ουρτασούν. Κυρία Ματίας, θα σας δώσω αμέσως το λόγο για την ισότητα των φύλων και τις φορολογικές πολιτικές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, θέλω να ευχαριστήσω τον Ερνέστο Ουρτασούν, καταρχά και ολόκληρη την ομάδα που εργάστηκε ώστε να ε, συνταχθεί αυτή η έκθεση. Ε, Επίση, θέλω να ευχαριστήσω τους κοιόδης ηγητέ από τις διάφορες πολιτικέ ομάδες για τη συμβολή τους και για τη διαθεσιμότητά τους να διαπραγματευτούν. Οι δυσκολίε ε, και ανισότητε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια θλιβερή πραγματικότητα. Πολλές φορές έχουν γίνει ψηφίσματα τα οποία έχουν υπερψηφιστεί που καλούν ε, για την ισότητα των φύλων. Όμως θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Θα πρέπει η ισότητα των φύλων να μπει μέσα σε όλες τις πολιτικές και να μην είναι μόνο δηλώσεις ε, και ε, ένας από τους διάφορους αγώνες είναι οι φορολογικές πολιτικές. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύονται στην αγορά εργασίας και εργάζονται μόνο ε, το 1 τρίτο εξ αυτών σε μερική απασχόληση. Η ισότητα ανάμεσα στους μισθούς είναι το 16% και στις συντάξεις φτάνει και το 40% είναι η ισότητα αυτή. Ε, πολλά χρόνια που έχουν συσσωρευτεί όλες αυτές οι ανισότητες. Μάλιστα, οι γυναίκες είναι αυτές που περισσότερο διακόπτουν τη σταδιοδρομία τους για ε, οικογενειακούς λόγους και που φροντίζουν ε, τους ανθρώπους με αναπηρίες με δυσκολίες. στις ε, φορολογικές πολιτικές έμεσες ή άμεσες πάλι οι γυναίκες βρίσκονται σε μενεχτική θέση. Οι περιοριστικές πολιτικές όσον αφορά την κατανομή της απασχόλησης, ε, του κατανάλωσης ή του πλούτου σημαίνει ε, μετάφραση σε μεγαλύτερη ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και ανισότητα όσον αφορά το φορολογικό φόρτο για τους μισθούς ε, που είναι χαμηλότεροι και αυτό πάλι επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες. Εδώ εμείς υποβάλλουμε διάφορες προτάσεις για να καταπολεμηθεί αυτή η ανισότητα των φύλων στον τομέα της φορολογίας. Και το πρώτον, αφορά, πρώτη πρόταση αφορά την άμεση φορολόγηση φορολόγηση των ατόμων, των εταιριών αλλά και του κεφαλαίου ε, και έμεση φορολόγηση έπειτα ειδικά όταν πρόκειται για το ΦΠΑ όπου ε, και πάλι οι γυναίκες φορολογούνται ε, όσον αφορά προϊόντα υγιεινής τα οποία φορολογούνται σαν να είναι προϊόντα πολυτελείας. Ε, επίσης, ε, όσον αφορά την ισότητα των φύλων ε, στις φορολογικές πολιτικές μέσω των, της τακτικής αναθεώρησης του αντικτύπου των φορολογικών πολιτικών σε θέματα φύλου. Εδώ Όλα αυτά που προτείνουμε μπορούν να υλοποιηθούν αν υπάρχει μια πραγματική πολιτική βούληση ώστε να υπάρχει ισότητα αντιμετώπιση και μεταχείριση των ανδρών και των γυναικών. Και αυτή την πρόταση θα πρέπει να τη σκεφτείτε αύριο όταν θα ψηφίσουμε για αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ, ο κύριο Σορτασούν. Σας ευχαριστώ. Ήθελα να ξεκινήσω ετοιμώντα την Πάμελα Νταμόβετ που μόλι δολοφονήθηκε στη Γκτάνσκ ήταν η δήμαρχος του Γκτάνσκ ε, δολοφονήθηκε, πράγμα που αποτελεί μια ευρωπαϊκή τραγωδία. Θέλω λοιπόν να αποτίσω φόρο τιμής και ο αγώνας της θα πρέπει να συνεχίσει να είναι αγώνας όλων μας. Επίσης θα ήθελα να ξεκινήσω ε, ευχαριστώντα τη Μαρίζα Ματία για τη συνεργασία στην εκπόνηση αυτή τη έκθεση, καθώ και ολόκληρη την ομάδα που μα βοήθησε, γιατί για πρώτη φορά θέσαμε ένα τέτοιο σημαντικό θέμα όπω είναι η φορολογία στο επίκεντρο των πολιτικών για την ισότητα των φύλων. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε ένα τέτοιο τόσο σημαντικό θέμα που ορίζει τον τρόπο ζωή μα ε, για το πώ δηλαδή δαπανούμε το, του πόρου μα να επηρεάζει και την προοπτική του ε, φύλου. Πρέπει λοιπόν ε, η ατζέντα μας για την ισότητα των φίλων να είναι πολύ φιλόδεξη. Τα τέσσερα χρόνια που είμαι εγώ εδώ είχαμε μια αρκετά ήπια ε, ατζέντα για την ισότητα των φίλων Είχαμε όλη εκείνη τη διαδικασία για την, ε, ακύρωση, για, την οδηγία για την άδεια μητρότητας, ε, τη σύμβαση της ε, Κωνσταντινούπολης, πολύ, πολύ δειλά βήματα σε θέματα ισότητας και πρέπει να δούμε ότι αυτή τη στιγμή αναδύονται δυνάμεις Πολλοί οι βίε σε ολόκληρη την Ευρώπη που αφισβητούν βασικές αρχές, όπως για παράδειγμα αφισβητούν ότι την ύπαρξη την ίδια της βίας που οφείλεται στο φύλλο. Για, από πολλές πλευρές βλέπουμε να ε, γίνονται επιθέσεις ε, όπως ας πούμε στην Ανδαλουσία ε, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αύριο στην Ισπανία κατεβαίνουμε στους δρόμους ε, σε, σε ένδειξη με τις γυναίκες ε, τη Ανδαλουσία. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο χτύπημα. Αλλά όπως είπα, δεν μπορούμε αυτές τις φάσεις να λέμε και να αμφισβητούμε ότι υπάρχει βία που οφείλεται στο φύλλο. Ε, θα πρέπει να έχουμε μια φιλόδοξη πολιτική, να καταπολεμήσουμε τη βία, να καταπολεμήσουμε την ανισότητα στους μισθούς και άλλες μορφές διακρίσεων που ποτέ δεν έχουμε εξετάσει, όπως ας πούμε τη φορολογία που το εξετάζουμε σε αυτήν εδώ την έκθεση. Να αρχίσουμε να έχουμε δημόσιες πολιτικές που αναλύουν πώς τα φορολογικά μας συστήματα άμεσης και έμεσης φορολόγησης είναι πολύ σημαντικά στα θέματα, για τα θέματα ισότητας. Ας πούμε, αν δούμε την άμεση φορολογία, Βλέπουμε ότι σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η υποχρέωση να κάνει κανείς ε, κοινή δήλωση, ε, φορολογική δήλωση, σημαίνει πως ε, ο δεύτερος φορολογούμενος δεν μπορεί εύκολα να μπει στην αγορά εργασίας. Αυτό επηρεάζει κυρίως τις γυναίκες. Και αν δούμε και την έμεση φορολογία σε πολλές χώρες και στην Γαλλία τονίστηκε πώς γίνεται προϊόντα τα οποία είναι πρώτες ανάγκες για τις γυναίκες να ε, ε, φορολογούνται με ΦΠΑ πολυτελείας. Αυτό είναι πραγματικά παράδεκτο. Και έπειτα θα πρέπει να δούμε και ποιο είδο, ποια συμπεριφορά διαφορετική έχουν οι άνδρες και οι γυναίκες όσον αφορά την κατανάλωση βλέπουμε πως κατά μέσο όρο οι γυναίκες πληρώνουν περισσότερο ΦΠΑ από ότι οι άνδρες. Ούτε το εξάμενο το ευρωπαϊκό, ούτε όλες οι συζητήσεις που έχουμε κάνει για τα φορολογικά θέματα που μας απασχόλησαν αυτή τη θητεία θα μπορούν να γίνονται ε, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το θέμα της ισότητας των φύλων. Γι' αυτό λοιπόν... Θα πρέπει από εδώ και στο εξή και κυρίως η επόμενη θητεία θα ασχοληθεί με αυτό το φαινόμενο πιο φιλόδοξα και να ε, κάνουμε μια τέτοια πολιτική ε, φιλόδοξη όπως αυτή που αξίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και ξεκινούμε το Κατσδιαή με την κυρία Σόιτροβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κατανοώ τις προθέσεις πίσω από αυτή την έκθεση και την ανάγκη να υπάρχει ισότητα των φύλων και να ε, καλυφθεί το χάσμα στις αμοιβέ μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ωστόσο, δεν θεωρώ ότι έχουμε επιλέξει τα καλύτερα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός δεν μπορεί να παραβιαστεί η αρχή της επικουρικότητας, ούτε μπορούν να περιγράφουμε εμεί από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το ποια μορφή θα έχουν τα φορολογικά συστήματα. Διότι αυτά εναπόκεινται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και τα κράτη-μέλη πάντοτε θα χρησιμοποιούν διαφορετικέ φορολογικέ πολιτικέ, βοηθήματα ε, για τις οικογένειε, γιατί αυτός ε, είναι ένα τρόπος που έχουν για την ε, προώθηση των οικογενειών, της οικογενειακής ζωής. Η έκθεση λοιπόν έρχεται σε αντίθεση με αυτήν την αρχή. Ε, λυπάμαι γι' αυτό. Αν και συμπαθώ πολύ τον κύριο Ούρτασον γιατί είμαστε μαζί και στην Επιτροπή αλλά δυστυχώς η έκθεση αυτή δεν είναι καλή. Um, Είναι πραγματικά αποτρόπαιο το γεγονός ότι έχουμε τέτοιου διακρίσεις για το φύλλο στα συστήματα, τα φορολογικά που έχουμε και πρέπει να δείτε τι συμβαίνει με τις γυναίκες και τα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί η φτώχεια δεν τους επιτρέπει ε, να έχουν πρόσβαση και στα πιο απλά ε, προϊόντα υγιεινής ε, για παράδειγμα, ε, στο Blackpool έχουμε το δωρεάν κόκκινο κουτί ε, που μοιράζει τέτοιου είδους προϊόντα στα ε, σχολεία. Γιατί υπάρχουν κορίτσια που δεν πάνε σχολείο κατά τη διάρκεια της εμεινουρίσης γιατί δεν έχουν παρά μόνο χαρτί τουαλέτας στη διάθεσή τους. Δεν μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους ε, έχοντας πρόσβαση σε τέτοια ε, προϊόντα υγιεινής. Ε, νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να δούμε τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ και επίσης ίσως και δωρεάν διάθεση αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μαριάς οι φορολογικές πολιτικές επηρεάζουν το εισόδημα των πολιτών και φυσικά επηρεάζουν και την ισότητα των δύο φύλων καθώς οι γυναίκες είναι πολύ πιο ευάλωτες στον τομέα της ε, οικονομίας. Το πρώτο που θα πρέπει να δούμε είναι ότι πρέπει να σταματήσει ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός γιατί με αυτόν τον τρόπο οι διάφορες πολυεθνικές δεν πληρώνουν φόρους εκεί όπου αποκομίζουν τα κέρδη αλλά σε φορολογικούς παραδείσους το δεύτερο θέμα είναι η υπερφορολόγηση. αυτό ισχύει ιδίως για την ελλάδα τεράστιοι φορολογικοί συντελεστές φορολογική λαιλασία από την πλευρά της τρόικας προκειμένου η ελλάδα να πετύχει τα περίφημα πλεονάσματα δηλαδή να δίδει 3% του ελληνικού αεπ στους δανειστές κάθε χρόνο μέχρι το 2022. Επιπλέον αυξημένος φόρος προστιθέμενης αξίας στα βασικά είδη διατροφής πολύ δε περισσότερο στα νησιά του Αιγαίου τα οποία βρίσκονται απομακρυσμένα από την κυρίως ελλάδα. αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πραγματικά να ενισχύεται η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός και πολύ περισσότερο ο κοινωνικός αποκλεισμός των γυναικών. επομένως πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα στο επίπεδο της φορολογίας. ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να σας πω το εξής. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που ε, θέσατε αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η έκθεση που συζητούμε σχετικά με την ισότητα των φύλων και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εγώ απορρίπτω κάθε μορφή διακρίσεων εις βάρος των γυναικών και ε, ωστόσο, νομίζω ότι οι κοινέ φορολογικέ δηλώσει δεν στρέφονται κατά των γυναικών. Το αντίθετο, με αυτόν τον τρόπο προωθούνται οι, οικογένειε, δηλαδή ζευγάρια τα οποία έχουν δεσμευτεί να φροντίζουν ένα τον άλλον και να μεγαλώσουν παιδιά. Ε, την έκκληση που υπάρχει στην έκθεση να υπάρξει ψηφοφορία στο Συμβούλιο νομίζω ότι είναι ατυχής διότι αυτό θα δημιουργούσε χώρο σε εθνικιστές και λαϊκιστές να ε, μας κατηγορήσουν ότι προσπαθούμε να παραβιάσουμε τις αρχές της εθνικής κυριαρχίας και νομίζω ότι δεν πρέπει να δώσουμε χώρο σε τέτοιες φωνές. Ο κύριος Πόλτσακ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, κύριε συνάδελφοι. Δεν θέλω να μειώσω τη σημασία του θέματος ε, της έκθεσης, η οποία περιέχει πολλά σημαντικά στοιχεία. Θέλω απλώς να τονίσω ότι ανισότητες υπάρχουν σε όλες τις κοινωνίες, σε όλες τις εταιρείες. Υπάρχουν, ε, υπάρχουν δυσκολίες πρόσβασης των γυναικών σε, είδη, σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας και υγιεινής και ε, πρέπει να σας πω ότι ήδη στην Τσεχία έχουν ξεκινήσει σχετικές πρωτοβουλίες και κινήσεις για την άρση αυτών των ανισοτήτων. Όπως για παράδειγμα οι ανισότητες στον τομέα των αμοιβών. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ε, το αναφέρει η έκθεση. Νομίζω λοιπόν ότι Πρέπει εδώ να τονίσουμε τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζουν τα κράτη-μέλη για την ε, ανάπτυξη φορολογικών συστημάτων τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τους στην αρχή της ισότητας των φύλων. Εγώ δεν έχω αντίρρηση με το περιεχόμενο της έκθεσης, αλλά θέλω να τονίσω ότι η επικουρικότητα είναι μια αρχή που πρέπει πάντοτε να γίνεται σεβαστή. Κυρία Γιούροβα έχει το λόγο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ε, για το γεγονό ότι θέσατε το ζήτημα της ισότητας των φύλων και των φορολογικών πολιτικών στην ημέρηση διάταξη εδώ της Ολομέλειας. Όπως είπατε και εσείς, η φορολογία είναι σημαντικό στοιχείο της ε, δημόσιας πολιτικής και αποτελεί εργαλείο για την εξασφάλιση αποτελεσματικής, ε, λειτουργικής και συμπεριληπτικής κοινωνίας. Ε, και αυτό, αυτές είναι και αρχές που μας καθοδηγούν εμάς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ισότητα των φύλων αποτελεί βασικό και πρωταρχικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η σχετική στρατηγική για την ισότητα των φύλων ακριβώς αποσκοπεί στο να λαμβάνεται υπόψη αυτή η διάσταση σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της φορολογίας χωρίς να παραβιάζεται βεβαίως η αρχή της επικουρικότητας και της εθνικής κυριαρχίας. Οι συστάσεις σας σχετικά με το πώς μπορεί να λαμβάνετε υπόψη αυτή η διάσταση της ότα των φίλων στην φορολογία θα συμβάλλουν στην διαμόρφωση σύγχρονων φορολογικών συστημάτων που θα αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις μιας ολοένα και πιο ε, ολοκληρωμένης ε, οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η σημασία των σχετικών κινήτρων έχει κοιτονιστεί στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής το 2018. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Κομισιόν έχει εντάξει το θέμα αυτό στην ετήσια ε, έρευνα που εκπονεί για την ανάλυση των φορολογικών εργασιακών πολιτικών και την, και την συνεισφορά του στην ανάπτυξη. Η ισότητα των φύλων αποτελεί επίσης σημαντική διάσταση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που συζητείται ε, σε βάθος σε πολλές εκθέσεις ε, αναχώρα πολλά κράτη-μέλη έχουν λάβει σχετικές συστάσεις για να άρουν τις ανισότητες και να ξεπεράσουν τα εμπόδια που υπάρχουν ε, στον τομέα της ισότητας των φύλων. Και η έκθεση αυτή ε, καλύπτει και το ζήτημα των εκείνων που ε, συνεισφέρουν σε δεύτερο βαθμό στο οικογενειακό εισόδημα και την ελάφρυνσή τους μέσω των φορολογικών πολιτικών. Αυτό είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε στο ευρωπαϊκό εξάμεινο, ιδίω για τη Γερμανία και το Βέλγιο. Η φορολογία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση τη ισότητα των φύλων, για παράδειγμα, ω ε, πηγή χρηματοδότηση δημόσιων πολιτικών και υπηρεσιών. Και από αυτή την άποψη εκτιμούμε την συνεισφορά της, ε, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν μπορούμε να, βασιζόμαστε στο ότι τα νοικοκυριά πάντοτε διαχειρίζονται με ισότητα το εισόδημά τους. Η κατανάλωση ε, ε, δεν μπορεί να ε, χαρακτηρίζεται από πολιτικές οι οποίες θα θέτουν σε δεύτερη μοίρα ή θα πλήττουν συγκεκριμένες κατηγορίες του πληθυσμού όπως είναι οι γυναίκες για παράδειγμα. Βεβαίως τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας αφορούν και απευθύνονται μόνο σε γυναίκες. Γι' αυτό και πράγματι τα κράτη-μέλη πρέπει να ε, μειώσουν τον ΦΠΑ όπως κάνουν και στα τρόφιμα. Ε, γιατί η ανισότητα στο εισόδημα ε, πολλές φορές οφείλεται ακριβώς στην έλλειψη σχετικών υπηρεσιών και σχετικών πολιτικών που δεν επιτρέπουν σε εκείνους που προσφέρουν φροντίδα στα μέλη της οικογένειας, ε, ένα ε, αξιοπρεπές εισόδημα, μια ισορροπία σε αυτό το τομέα. Γι' αυτό και χρειάζεται να γίνουν περισσότερα πέραν από τις φορολογικές πολιτικές για να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες μεταξύ των φύλων. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση λοιπόν χρειαζόμαστε που θα συμπεριλαμβάνει νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα. Και αυτή είναι η προσέγγιση που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παράδειγμα, στο πακέτο μας για την ε, ε, συμφιλίωση επαγγελματική και προσωπική ζωή και στι σχετικέ στρατηγικές που έχουμε εκπονήσει. Θέλω επίσης να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις δράσεις της παραμένει πάντοτε προσελωμένη στην ε, εξασφάλιση της οικονομικής ανεξαρτησίας ανδρών και γυναικών, το ξεπέρασμα του χάσματος στις αμοιβέ μεταξύ των δύο φύλων, που σε κάποια κράτη-μέλη είναι πολύ υψηλό στην καταπολέμηση της ε, βίας κατά των γυναικών και την πρόθεση της ε, ισότητας των δύο φύλων. Όπως είπα, η φορολογική πολιτική είναι ένας πολύ σημαντικός ε, τομέας για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Έκθεση Βιν Βαντεκάμπ, αυτόνομη οδήγηση σε ευρωπαϊκές μεταφορές. Κύριε εισηγητή, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να ευχηθώ σε όλους όσους δεν το έκανα ήδη. Καλή χρονιά. Υγεία. Φέτος μας περιμένουν ευρωεκλογές. Καλή επιτυχία. Θέλω να ευχαριστήσω τους σκιώδεις ηγητές, αλλά και τους ε, σκιώδεις της Επιτροπής ε, ΙΜΚΟ και της ε, Επιτροπής της Νομικής γιατί με βοήθησαν να συντάξουμε μια εξαιρετική, ε, μάλλον με τις εξαιρετικές τους γνωμοδοτήσεις συνέβαλαν στην σύνταξη της δικής μου έκθεσης. Αυτή η έκθεση λοιπόν δεν αφορά μόνο τα αυτόματα οχήματα αλλά και διάφορα μέσα μεταφορών όπως ας πούμε το μετρό, το τρένο αλλά και σκάφη αυτόνομα. Πρόκειται για βιομηχανικές εξελίξεις που θα πρέπει να δούμε με θετική ματιά. Γίνεται λόγος για νέες λοιπόν τεχνολογίες βλέπουμε για εξελίξεις και στον τομέα της, ε, του διαστήματος. Είναι εξαιρετικά σημαντική η ανάπτυξη αυτόνομων ε, οχημάτων. Αν λάβουμε υπόψη και τα project καινοτομίας ε, μέχρι το 2030. Εν τω μεταξύ, ο ανταγωνισμό και η θέση μα απέναντι στο ΗΠΑ, την Κίνα και το Ισραήλ είναι εξαιρετικά σημαντική. Όλε αυτέ οι χώρε αναπτύσσουν αυτόνομα οχήματα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ένα άλλο όμως πολύ σημαντικό θέμα παράλληλα είναι η ασφάλεια στους δρόμους. 90% των οδικών ατυχημάτων οφείλονται στο ανθρώπινο λάθος. Και όταν μιλάμε για οδικά ατυχήματα, μιλάμε και για ευθύνη. Ποιος φέρει την ευθύνη όταν ε, γίνει ατύχημα με αυτόνομο όχημα πολύ ενδιαφέροντα και πολύτιμα τα όσα μας είπε η νομική υπηρεσία περί όλων αυτών. Κάτι άλλο σημαντικό είναι η ψυχολογία του αυτόνομου αυτοκινήτου ή οχήματο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο πολίτης είναι σε θέση να παραδώσει τον αυτό του σε ένα τελείως αυτόνομο όχημα. Αυτό ε, θα... Ε, ε, είναι μεγάλη αλλαγή. Επίσης θέλω να ζητήσω την προσοχή σας για τους εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονται στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μεταφορών που ανησυχούν για τις θέσεις απασχόλησής τους εφόσον έχουμε μία μετακίνηση προς τα πλήρως αυτόνομα οχήματα. Να ρωτήσω λοιπόν την Κομισιόν, είναι δυνατόν να έχουμε μόνο ένα σύνολο νομοθεσία στην Ευρώπη. όσον αφορά τα αυτόνομα οχήματα, είτε είναι αυτοκίνητα, είτε είναι ε, ε, σκάφη για την εσωτερική ε, ναυσιπλοεία, είτε είναι λεωφορεία, είτε οτιδήποτε. Θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή νομοθεσία η οποία θα συζητηθεί στην Γενέβη και έπειτα προστασία προσωπικών δεδομένων. Προστασία δηλαδή και ε, των ε, δεδομένων ε, σε αυτά τα οχήματα. Θα πρέπει η Κομισιόν να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει ισότιμο πεδίο. Να καλέσω λοιπόν την Κομισιόν αυτό να το φροντίσει και να καλέσω και την επόμενη νέα Επιτροπή να μελετήσει και το κεφάλαιο της ανάπτυξης των αυτόνομων οχημάτων εντός της Ένωσης μέχρι το 2024. Ευχαριστώ. Πολτσακ. Eh, ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Να σας πω πως καταγράφω το μεγάλο δυναμικό που έχει αυτού του είδους η αυτόνομη οδήγηση, νέες εμπορικές ε, προπτικές, επίσης και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτό να το κρατήσουμε, μεγάλες δυνατότητες που ανοίγονται στον κλάδο, και νομίζω πως θα πρέπει να καλωσορίσουμε και τη δυνατότητα νέων υπηρεσιών, νέων θέσεων εργασίας. Βεβαίως μπορεί να χαθούν για κάποιες θέσεις εργασίας ε, μέσω αυτών των εξελίξεων, αλλά πρέπει να δούμε και τη διάσταση της ασφάλειας, ε, πώς θα ασφαλίζονται αυτά τα αυτόνομα οχήματα, τι θα γίνει με τις υποδομές και αν θα αντέξουν όλα αυτά δεν πρόκειται να λυθούν ε, ως διαμαγές από το γεγονός πως θα έχουμε αυτόνομα αυτονομή οδήγηση, θα πρέπει να προκρίνουμε ακόμα πιο πολύ τις δημόσιες συγκοινωνίες της πόλης μας. Νομίζω ότι νομοθετικά πολλά καθήκοντα ακόμα έχουμε μπροστά μας. Κύριε Μαριά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η αυτόνομη οδήγηση στις μεταφορές είναι πραγματικά μια σημαντική εξέλιξη η οποία εκ των πραγμάτων θα επιβληθεί πλέον τα επόμενα χρόνια. Και είναι δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ανταγωνισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, την Ιαπωνία, που προχωρούν με ταχύτερους ρυθμούς στην αυτόνομη οδήγηση. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες, πολύ σημαντικές, κυρίως κοινωνικές, κυρίως στον τομέα της απασχόλησης. Αυτά όλα πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να υπάρχει μια κοινωνική στήριξη σε όσους καθώς η τεχνολογία θα αναπτύσσεται στον τομέα της αυτόνομης οδήγησης αυτοί οι άνθρωποι ενδεχόμενα θα χάνουν τις δουλειές τους. από εκεί και πέρα υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με την ασφάλεια ασφάλεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των μεταφορών το οποίο επίσης θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. επομένως ναι στην εξέλιξη της τεχνολογίας ναι στην πρόοδο αλλά με τρόπο ο οποίος να είναι ασφαλής και κοινωνικά δίκαιος. ευχαριστώ κύριος η αλματώδης εξέλιξη στους τομείς ε, της ρομποτικής και της τεχνικής ε, νοημοσύνης μας δίνει την ικανότητα αλλά και τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε και να υλοποιήσουμε ε, ένα όραμα που υπήρχε από το παρελθόν σχετικά με την αυτοματοποίηση της κινήσεως βεβαίως αυτή η εξέλιξη θα έχει αρκετά θετικά στοιχεία όπως παραδείγματος χάρη θα αυξήσει την ασφάλεια θα μειώσει το κόστος της ε, μεταφοράς θα αυξήσει την προστασία του περιβάλλοντος και γενικώ θα ε, επηρεάσει κατά τρόπο θετικό την καθημερινή μας ζωή. πέραν αυτών όμως υπάρχουν και κάποια προβλήματα κάποιες δυσχέρειες κάποιοι κίνδυνοι οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως είναι παραδείγματος χάρη η ασφάλεια στην οδήγηση η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο η ασφάλεια και η προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς επίσης και η δυνατότητα να ελέγχεται η προσωπική ζωή των ε, ανθρώπων. πέραν αυτών υπάρχουν και νομικής φύσεως θέματα αλλά και κοινωνικής όπως παραδείγματος χάρη οι επιπτώσεις που θα υπάρξουν στις ε, θέσεις εργασίας. άρα λοιπόν η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να ε, υλοποιήσει και να εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αυτοματοποίησεως. ευχαριστώ voertuigen, collega's, zullen. Ευχαριστώ. Η αυτόνομη οδήγηση αργά ή γρήγορα θα έχει σημαντικότατε επιπτώσει στον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε, οδηγούμε και μεταφέρουμε τα εμπορεύματά μας. Ο εισηγητή δικαίω. Ε, παραπέμπει και σε άλλα είδη μεταφορών, εσωτερικές πλωτές οδοί, μετρό, drones. Η αυτόνομη οδήγηση θα προσφέρει νέες δυνατότητες και στις διατροπικές μεταφορές. Θέλω να υπησέλθω και στα, στους, στις ροές δεδομένων που θα δημιουργούνται μέσω αυτών των νέων μορφών οδήγησης. Το εύρος των δυνατοτήτων που θα δημιουργηθούν από ε, οχήματα τα οποία θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και με το περιβάλλον είναι απρόβλεπτο ακόμα. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να προστατευτούν τα προσωπικά δεδομένα για να μπορούν να εφηλθούν όλοι από τις νέες αυτές τεχνολογίες θα χρειάζεται να υπάρχει πρόσβαση και για τρίτους στα δεδομένα που θα δημιουργούν τα οχήματα, κάτι που θα ενισχύσει συνολικά και, το, και την καινοτομία. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Γιούροβα έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, ο κλάδος των μεταφορών αλλάζει ραγδαία και πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτές τις αλλαγές και να καταστήσουμε την ευρωπαϊκή κινητικότητα πιο βιώσιμη, πιο ασφαλή και πιο προσβάσιμη. Χρειάζονται δράσεις. Αν θέλουμε ο ευρωπαϊκός κλάδος ε, να γίνει πιο ανταγωνιστικός και να εξασφαλίσουμε τις θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Αυτές οι πραγματικότητες αντικατοπτρίζονται ε, εξαιρετικά στην έκθεση του κυρίου Βίντεκάμπ ε, που υποστηρίζει την, περισσότερη, την μεγαλύτερη συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πω δύο λόγια για το πώς θα επιτευχθεί η βιωσιμότητα. Οι μεταφορές συμβάλλουν σημαντικά στις εκπομπές ε, ε, αερίων του θερμοκηπίου και στην ρήπανση του αέρα. Γι' αυτό και οι δράσεις μας θα πρέπει να κατευθύνονται στην απαλλαγή από τον άνθρακα. Η αυτόνομη και αυτόματη οδήγηση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εργαλείο γιατί βοηθά στην ομαλότητα ευκολότερη διαχείριση των κυκλοφοριακών ροών και γι' αυτό σας ευχαριστώ για την ασφάλεια, για την οδική ασφάλεια. Πριν από ε, λίγο καιρό, το να λέμε ότι έως το 2050 θα επιτύχουμε το στόχο μηδέν νεκροί στους δρόμους φαίνονταν πολύ φιλόδοξος. Όμως, με τη στρατηγική που έχουμε εκπονήσει, έχουμε κατακτήσει ένα σημαντικό ορόσημο μέσω του πακέτου για την αυτόνομη κινητικότητα με μια νέα ε, δομή για την ασφάλεια προτείνοντας μια νέα δομή η οποία θα καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ηγέτη στον κόσμο στον, ε, στην αυτόνομη οδήγηση. Σε τρεις πυλώνες βασινόμαστε. Πρώτον, ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα δημιουργήσει ένα μια ενιαία αγορά για την ε, αυτόματη ε, κινητικότητα. Δεύτερον, χρηματοδοτική στήριξη που θα καλύπτει όλο τον ε, κλάδο της οικονομίας και τρίτον μια σε βάθος αξιολόγηση των κοινωνικο-οικονομικών και διοντολογικών πτυχών της αυτοματοποιημένης οδήγησης. Τα οχήματα Όλο ένα και πιο πολύ γίνονται καθαρά συνδεδεμένα και αυτοματοποιημένα και στο τέλος αυτού της διαδρομής ε, θα καταλήξουμε να έχουμε οχήματα χωρίς οδηγούς πράσινα, χωρίς εκπομπές. Χρειάζεται όμως και ε, ταυτόχρονα όμως οι καταναλωτές αλλάζουν και στάση απέναντι στις, ε, στις διάφορες μορφές μεταφορών. Χρειάζονται ε, καλύτερες πληροφορίες, καλύτερη πρόσβαση. Τα οχήματα μπορούν λοιπόν να αποτελέσουν συστατικό στοιχείο της ε, πολυτροπικής μεταφοράς, των πολυτροπικών μεταφορών, δίνοντας ε, και προσφέροντας ε, ολοκληρωμένες λύσεις σε όλους τους πολίτες συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων των αναπήρων. Προτού όμω φτάσουμε στο στόχο αυτό, πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια σειρά από εμπόδια, τα οποία αναφέρατε κι εσεί και που σχετίζονται με την ασφάλεια, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την προσβασιμότητα στα δεδομένα, την ευθύνη και τι δεοντολογικέ πτυχέ, την ε, ένταξη των αυτοματοποιημένων οχημάτων στα υπάρχοντα συστήματα ε, κυκλοφορίας στις πόλεις και στην Ήπεθρο. Γι' αυτό και θέλω να τονίσω τρεις διαστάσεις των ε, δράσεων που έχουμε ε, θεσπίσει. Δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας για τη συνεργατική και αυτοματοποιημένη κινητικότητα στην οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να συνεργάζονται για να προωθήσουμε αυτήν τη φιλόδοξη ατζέντα μας. Δεύτερος πυλώνας, κοινή επιχείρηση για αυτήν την συνεργατική αυτοματοποιημένη κινητικότητα η οποία θα βοηθήσει στην, ε, στο συνδυασμό δημόσιων και ιδιωτικών πρωτοβουλειών που θα κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Έχω σημειώσει και σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας και σε αυτή τη διάσταση της δράσης μας. Τρίτον, αναθεώρηση των ευρωπαϊκών κανόνων και θέσπιση νέου νομοθετικού πλησίου για τα συνδεδεμένα και αυτοματοποιημένα οχήματα. Και σε αυτόν τον τομέα θέλω να σας ευχαριστήσω για τη στήριξη, αλλά θέλω πραγματικά να σας καλέσω έως το τέλος της θητείας να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για αυτό το νομοθετικό κείμενο. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Όπως βλέπετε, το μέλλον της κινητικότητας και ε, ο, ο ρόλος του τελικού χρήστη βρίσκονται στο επίκεντρο των δικών μας δράσεων και των δικών μας σκέψεων βλέπουμε ότι η κινητικότητα είναι θεμέλιος λίθος των ελευθεριών των πολίτων και αποτελεί συστατικό στοιχείο και απαραίτητο όρο για την ομαλή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έκλεισε η συζήτηση. Θα ψηφίσουμε αύριο. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στις παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού, άρθρο 163 του κανονισμού. Ο κύριος Βίγκλε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Από τότε που προσχώρησε τη Ρουμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για πρώτη φορά βρέθηκε στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τεράστιες προκλήσεις και δεν ξέρουμε αν θα είναι πετυχημένη αυτή η Προεδρία και δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει να μπει στην αίρια, στο χώρο Σέγγεν η Ρουμανία. Ο κύριος Γιούνκερ στο Βουκουρέστι δήλωσε πως θα ήταν πολύ σημαντικό το βήμα αυτό. Ο κύριος Γιάννη είπε πως τα κράτη-μέλη που είναι κατά αυτής της προχώρησης της Σέγγεν θα έπρεπε να αλλάξουν ε, άποψη. Εδώ και 8 τουλάχιστον χρόνια η πρόσβαση, η προσχώρηση της Σέγγεν ε, έχει εμποδιστεί και ελπίζουμε πως στους επόμενους έξι μήνες αυτό θα γίνει υπέρ της χώρας μας, υπέρ των πολιτών μας και υπέρ ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι ώστε να μην θεωρούνται οι πολίτες μας δεύτερης κατηγορίας. Η κυρία Μικρόφωνο παρακαλούμε. Ευχαριστώ πολύ. Πήρα το λόγο γιατί θέλω να μιλήσω για ένα κλάδο που είναι τα εσπεριδοειδή στη Βαλένσια, που είναι πολύ σημαντικά για την κοινότητα την οποία εκπροσωπώ, την Ισπανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Βαλένθια είναι η πρώτη εξαγωγική περιοχή ε, περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω από 2 δις ε, ευρώ και τεράστιοι κίνδυνοι ε, λόγω ε, κακών συνθήκων στην αγορά με πολύ χαμηλές ε, τιμές παραγωγού. Ε, χρειαζόμαστε λύσεις για τον κλάδο. Είναι γύρω στο 130.000 ευρώ το μήνα οι απώλειες σε αυτή την περιοχή. Οπότε χρειάζεται επιδοτήσεις για να μπορούν να ανταγωνιστούν την Αίγυπτο και την Τουρκία. Εναρμόνιση των ε, τελωνιακών διαδικασιών για να μην έχουμε ε, προβλήματα ανταγωνισμού και οποιοδήποτε, μεγαλύτερη παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίπτωση που έχουμε ε, καρτέλ στις τιμές. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριος Τζαμπάτσκι. Ευχαριστώ. Τρεις προτάσεις για το πακέτο της κινητικότητας θέλω να κάνω. Εδώ στον τομέα αυτό Δυστυχώ ε, απορρίφθηκαν προτάσεις που συζητούνταν επί μακρόν. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί θα χάσουν τις δουλειέ τους ε, και φαίνεται ε, έχουμε να κάνουμε μια, με περίπτωση παραβίασης των αρχών της ενιαίας αγοράς υπάρχουν στρεβλώσεις εναντίον των ανατολικών χωρών είναι πραγματικά μια σοβαρή αποτυχία αυτή που έχουμε στα χέρια μας εδώ με, το, με την κινητικότητα ε, και τις μεταφορές. Ε, δυστυχώς το Κοινοβούλιο δεν έχει πλέον εντολή, αλλά ε, για να ε, ξεκινήσουμε νέες διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή, αλλά πραγματικά δεν πρέπει να επιτρέψουμε να ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ. Ευρωεκλογέ. Δυστυχώς δεν θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μόνο τον ε, φόβο αφενός και την εφορία βεβαίως που, που νιώθουν τα εθνικιστικά και λαϊκιστικά κόμματα. Έχουμε να κάνουμε με την ίδια την αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε και την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον πρόεδρο της Ισπανίας λίγες μέρες πρωτού ξεκινήσει η δίκη ε, κατά των ε, ε, ακτιβιστών ε, της Καταλωνίας. Θα μιλήσουμε και για τα όσα επικρατούν στην Δυτική Σαχάρα, για παράδειγμα, όπου επίσης ε, παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης έχουμε υποσχεθεί ευρωπαϊκό μέλλον στην Μακεδονία και εδώ πραγματικά ε, θα κριθεί η αξιοπιστία μας και όχι στην ρητορική των λαϊκιστών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με πλειοψηφία 92% ε, ε, ενέκρινε την πολιτική ε, διπλής, ε, για τις ουσίες διπλής χρήσης για να παρεμποδιστούν αυτή η προμήθεια ε, δικτατόρων, δικτατορικών καθεστώτων με ουσίες που μπορούν να, να στρέψουν, να χρησιμοποιήσουν εναντίον των ε, πληθυσμών τους. Να ε, υπενθυμίσω μόνο τις περιπτώσεις Σόκη και την Αραβική Άνοιξη. Αυτή η, αυτός ο κανονισμός για τη διπλή χρήση πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο. Αλλά εκεί τα πράγματα παρακολύονται. Αρχικώς από Σουηδία ε, και Φιλανδία και τώρα από τη Γαλλία. Είναι πραγματικά ακατανόητο πώς η Γαλλία αρνείται να αναλάβει δράση για την καταπολέμηση των παραβιάσεων, των καθημερινών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται με την αξιοποίηση γαλλικής τεχνολογίας και αυτό παρά τις προσπάθειες που έχει αναλάβει η Ρουμανική Προεδρία. Είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος, η γαλλική κυβέρνηση δεσμεύεται και εκείνη από την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κύριος Μακάρθη. Το περασμένο μήνα εγκρίναμε εδώ αυτό το ταμείο που θα δώσει 30 δις ε, στο Ταμείο Άμυνας και θα καλύπτει όλο τον κύκλο ζωής ε, όπλων, φωνικών όπλων, ε, στηρίζοντας την αμυντική βιομηχανία που στηρίζει δολοφονικούς πολέμους στην Ιωμένη, στη Συρία ε, και με τεχνολογία που χρησιμοποιούν οι πιο βίαιες κυβερνήσεις στον κόσμο. Και αυτό είναι κατά της ουδετερότητας που ε, επικαλείται η Ιρλανδία και που υποσκάπτουν οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια. Θα έπρεπε να παίζουμε ένα πιο επικοδομητικό ρόλο στις διεθνείς σχέσεις και να κάνουμε μόνο ειρηνευτικές αποστολές έτσι ώστε να μην ε, βοηθάμε σε οτιδήποτε άλλο παρά την επίλυση σειράξεων και όχι στην δημιουργία ε, πολέμων. Γιατί με την πολιτική αυτή γινόμαστε λιγότερο ασφαλείς και συνδυόμαστε με τις χειρότερες δράσεις των δυνάμεων που συμμετέχουν στις ε, ε, αποστολές αυτές. Πρέπει για μια φορά ακόμα να υποστηρίξουμε την Ιρλανδική ουδετερότητα. Ο κύριος παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γαλλία είναι η αρχή του τέλους αυτής της Ευρώπης που επιχειρείται εδώ ουτοπικά να ε, πραγματοποιηθεί. Και αυτό είναι πραγματικά απόδειξη για το πόση απόσταση χωρίζει τους ευρωγραφειοκράτες από τους ε, λαούς. Ε, ξεκίνησε η υπόθεση από την κλιματική αλλαγή, τις σχετικές πολιτικές και την αύξηση της τιμής των καυσίμων. Μέσω της ε, δίθερα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής έχουν ακουστεί οι πιο αδιανόητες υποσχέσεις και οι πολίτες ε, πλέον βλέπουν μπροστά τους αυτήν τη χρεοκοπία του κρατικού σοσιαλισμού. Έτσι λοιπόν ε, αυτή την τροπή πήρε η δημόσια συζήτηση ε, την ίδια άκουσα θα ακολουθήσουν και συζητήσεις όπως αυτή για την κατάρριξη θανατικής ποινής κτλ. κτλ. Κύριος Φαρή. Ευχαριστώ. Το 2019 ξεκίνησε με πολύ έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στην ε, Κίνα και την Ταϊβάν. Ο πρόεδρος της Κίνας, Σινπίνγκ, ε, ε, επανέλαβε τις απειλές του εναντίον της Ταϊβάν. Αυτές οι απειλές είναι ακόμα πιο επικίνδυνες γιατί η Ταϊβάν μπορεί να μάλλον η αντιπαράθεση αυτή με την Ταϊβάν μπορεί να οδηγήσει σε εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στην Κίνα και στις ε, ΗΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να διακόψει τους ε, εμπορικούς και διπλωματικούς της ε, δεσμούς με την Ταϊβάν γιατί με την χώρα αυτή συμμεριζόμαστε κοινέ αξίες και γι' αυτό και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε μη ειρηνικό τρόπο αποφα... Ε, λήψης απόφασης για το μέλλον της Ταϊβάν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φεραντίνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η διαδικασία παγκοσμιοποίηση έδωσε όθεση στι τεχνολογικέ καινοτομίε σε δύο τομεί κλειδί: επικοινωνίε και μεταφορέ. Σε σύγκριση με το παρελθόν, οι επιλογέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο εύκολο να μετακινηθεί κανεί ε, μέσα στο ίδιο το κράτο, αλλά και ανάμεσα σε αυτά. Όμω υπάρχουν και διάφορε ε, ε, περιοχές όπου υπάρχουν μεγάλε δυσκολίε, ε, μια από τι πιο γνωστέ προβληματικέ περιοχέ είναι η Καλαβρία. Δεν υπάρχουν τόσο εύκολες είσοδοι έξοδοι είναι απομονωμένη η Καλαβρία, κυρίως αφού η Ryanair ακύρωσε τις επιτήσεις της. Η Αλιτέλεια ε, κυριαρχεί με τιμές ε, στην οικόνομη που, στη θέση οικόνομη που φτάνουν τα 160 ευρώ για, την, ε, για να πάει κανείς μέχρι τη Ρώμη. Ψηλές είναι τιμές και για το τρένο. Ε, το να φτάσει δε κανείς στην πρωτεύουσα με το τρένο ψηλής ταχύτητας χρειάζεται 80% 80 ευρώ. Πολύ ψηλό αντίτιμο δηλαδή, ενώ για να φτάσει κανείς από τη Ρώμη στο Μιλάνο κοστίζει μόνο 44 ευρώ. Η Καλαβρία μένει έξω ε, λοιπόν από τις ε, ευκαιρίες πρόοδου. Ο κύριος Κρύπεκ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από τη Συρία θα έχει πολύ σοβαρέ συνέπειε. Η τουρκική επιθετική εξωτερική πολιτική δεν εκπλήσει κανέναν. Οι πολιτικοί προφορικά απειλούν τους γείτονες ε, τους καθημερινά. Έχουμε δε ε, διαπιστώσει 100.000 χριστιανούς που βρίσκονται ε, στα σύνορα με την Τουρκία και περιμένουν ε, ε, φοβούνται μάλλον ότι θα πέσουν στα χέρια των τζιχαντιστών μόλι φύγουν οι αμερικανικέ δυνάμει από την περιοχή. Εμεί καλούμε την Αμερικανική κυβέρνηση να ε, επιβραδύνει την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων μέχρι ότου να είναι σε ασφάλεια οι χριστιανοί τη ε, Συρία. Καλό τα κράτη-μέλη να ενθαρρύνουν τον Τούρκο εταίρο να μην επιδεινώσει τις εντάσει εκεί και να θεσπίσει θεσπιστεί μία ε, ζώνη μη πτήσης ώστε να μπορέσουν οι Σύροι να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους ενάντια στον Τουρκο, στην στις τουρκικές επιθέσεις. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σελίμωβιτς. Ευχαριστώ πολύ. Τρία, τρία χρόνια δεν έχει καταλάβει η καταφερή Βοσνία και η Ερζεγοβίνη να εγκρίνει τους κανόνες για ε, τις σχέσεις μας. Και για αυτά τα τρία χρόνια ακούμε ιστορίες για το πώς θα έπρεπε εμείς να εγκρίνουμε ε, τους ε, διαδικαστικούς κανόνες και το πρόβλημα είναι πως το κράτος δεν λειτουργεί έτσι και δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς για αυτούς τους κανόνες γιατί έτσι δεν θα ε, λειτουργούμε ούτε εμείς. Αν θέλει να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εγκρίνουν τους κανόνες οι οποίοι ακολουθούνται εδώ. Τρία χρόνια χάσαμε και ελπίζω με, τις ε, ε, με τη νέα πολιτική ηγεσία θα βρεθεί μια λύση και η χώρα αυτή θα ξεκινήσει γιατί υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να γίνουν πριν προσχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σολέ. Ευχαριστώ πολύ. Η Ισπανική κυβέρνηση αρνήθηκε στην Open Arms την άδεια για να συνεχίσει να ζώσει ζωές στην ε, Μεσόγειο. Δεν έχουν δικαίωμα απόπλο από την Βαρκελόνη με το εξής διαστροφικό επιχείρημα αφού η Ιταλία, η Μάλτα και η Λιβύη δεν προσφέρουν ασφαλή λιμάνι για ε, όσους πνίγονται δεν είναι ασφαλές ε, να σώζονται αυτοί οι άνθρωποι και έτσι δεν γίνεται διάσωση μέσα στο διεθνές δίκαιο. Επίσης δεν μπορεί ε, να, να πλέει ε, το πλοίο αυτό γιατί είναι υπερβολικός ο αριθμός ανθρώπων που μεταφέρει. Λες και πρόκειτο για σκάψα να ή κρουαζιερόπλοιο γιατί ε, αυτοί οι καημένοι άνθρωποι δεν είναι ούτε πλήρωμα ούτε επιβάτες. 2.000 265 άτομα πνίγηκαν πέρσι στη Μεσόγειο. Πιστεύετε πως έχουμε ακόμα το δυνατότητα να μπλοκάρουμε ε, πλοία τα οποία ως μοναδικό στόχο έχουν να μειώσουν ε, τον αριθμό των ανθρώπων που υποφέρουν. Με κάθε πλοίο που δεν φεύγει από το λιμάνι, με κάθε άνθρωπο που πνίγεται, πνίγονται και οι ευρωπαϊκές αξίες. Ο κύριος Λιαρίκ. Στην αρχή της χρονιάς Μία Ολλανδική εφημερίδα ε, είπε πως η Google έστειλε 20 δις ευρώ στις Βερμούδες. Αυτή η απάτη είναι τραγική όταν έχουμε πολίτες εμείς που δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς και χάνουμε όλα αυτά τα εκατομμύρια δισεκατομμύρια ευρώ που θα έπρεπε να πληρώνονται φόρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε ε, για σχολεία, για νοσοκομεία, ε, για συγκοινωνίες και να μην ε, πηγαίνουν στη Βερμούδα στους λογαριασμούς των πλουσίων δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε κοινωνική πολιτική φιλοδοξία αν γίνεται. Τα χρήματα υπάρχουν στις μαύρες τρύπες της χρηματοδότησης. Είναι λοιπόν επίγον ε, το Συμβούλιο ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τις διεθνείς προτάσεις του ΩΣΑ να απαγορέσουν αυτή την πρακτική και να υποχρεώνουν τις τράπεζες και τις πολυεθνικές να επιστρέψουν τα χρήματα που έκλεψαν και να πληρώσουν αυτό που τους αντιστοιχεί σε φόρους. Ευχαριστώ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 ε, διαμαρτυρηθεί εναντίον της ε, Σοβιετικής εισβολής στην Τσεχοσλοβακία το 1968 για να ενισχύσει ε, τον, την ευαισθητοποίηση των πολιτών, των συμπολιτών του γύρω από τα ιδανικά της άνοιξης της Πράγας το 1968 ήθελε να αποδείξει την ανάγκη αλλά και την αξία της αντίστασης. Τη μνήμη του λοιπόν ε, τιμήσαμε το 1989 όταν πολλοί άνθρωποι εξεργέρθηκαν εναντίον της αστυνομικής καταστολής. Ο άνθρωπος αυτός πέθανε όμως ο θάνατός του δεν ήταν μάταιος διότι τώρα πια ζούμε ε, σε καθεστώς ελευθερίας. Ευχαριστώ. Κυρία Μάιερ. Ευχαριστώ. Οι άνθρωποι από εκεί μας είπαν ότι το Brexit θα ήταν εύκολο. Θα έφερνε εύκολες εμπορικές συμφωνίες, εύκολα λεφτά για το εθνικό σύστημα υγείας. Τι ήταν αυτά. Διότι τώρα πλέον έχουμε αυτό ακριβώς που θέλαν. Από την κυβέρνηση που έδωσε μάλιστα συμβόλαιο σε εταιρεία Ferry Bot που δεν έχει Ferry Bot και που δεν μπορεί να διαχειριστεί ούτε μια απλή κυκλοφοριακή συμφόρηση και που καλείται πλέον να πληρώσει δισεκατομμύρια σε μια συμφωνία διαζυγίου. Αυτή η συμφωνία είναι κακή για τους εργαζόμενους ε, στο Λούτον, στο Στάνστετ, για τους ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Αντικαταστήσαμε την πραγματική δύναμη με την, ε, με την κυριαρχία έναντι ε, μιας έννοιας, ε όχι στο όνομα Θέλω λοιπόν να καλέσω όλους, ιδίως στη Βουλή των ε, Εκπροσώπων, να καταψηφίσουν τη συμφωνία αυτή και να δώσουν ένα τέρμα σε αυτήν την εθνική ταπείνωση. Ο κύριος Μαριάς. Η Μέρκελ με την επίσκεψή της στην Αθήνα προκάλεσε τον ελληνικό λαό τόσο με την άρνησή της να καταβάλει τις γερμανικές αποζημιώσεις όσο και με τις πιέσεις της για εφαρμογή της κατάπτυστης συμφωνίας των πρεσπών μια συμφωνία που ξεπουλά το όνομα της μακεδονίας μας και της ιστορίας μας και ενισχύει την αδιαλαξία και τον σκοπιανό αλυτρωτισμό. ο ελληνικός λαός δεν ανέχεται την ταπείνωση και αντιδρά μαζικά καθώς βλέπει τον τσίπρα να μεθοδεύει τη διαμόρφωση μιας ετερόκλητης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας κουρελού προκειμένου να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης και να ακυρώσει τη συμφωνία των πρεσπών και όλα αυτά καθώς δεν τολμά να κάνει δημοψήφισμα για το σκοπιανό όπως απαιτούν οι έλληνες. μεθοδεύει κύρωση της συμφωνίας των πρεσπών με διάφορα πολιτικά ρετάλια και με 151 βουλευτές ενώ σύμφωνα με το σύνταγμα για την κύρωση απαιτούνται 180 ψήφοι μια και η συμφωνία αυτή εκχωρεί κυριαρχικά δικαιώματα στους σκοπιανούς. όμως ο τσίπρας σχεδιάζει χωρίς τον ελληνικό λαό που ενωμένος θα στείλει αποφασιστικό μήνυμα μαζικά ειρηνικά και δημοκρατικά στο συλλαλητήριο του συντάγματος την Κυριακή 20 Ιανουαρίου. Δεν βλέπω την κυρία Βιέ, οπότε θα ε, περάσουμε στην κυρία Πένιας. Πένιας πολυεθνικές εγκαθίστανται σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο λόγω των μεγάλων πλεονεκτημάτων που μπορεί εκεί να κερδίσουν και μόλις εγκατασταθούν θέλουν να μειώσουν το εργασιακό κόστος αλλά και τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Αυτό συμβαίνει με τη μεγάλη αμερικανική εταιρεία GOS που αποφάσισε να παράγει τώρα το αλουμίνιο στη Σαουδική Αραβία και όχι πια στην Ισπανία. Γιατί δεν θέλει να έχει καμία έναν ανταγωνισμό. 700 ε, ε, άμεσες θέσεις απασχόλησης κινδυνεύουν ε, πρέπει να δούμε και το σύνολο τη κοινότητα όπου εγκαθίστανται τέτοιου είδου εργοστάσια. Και γι' αυτό και ζητάμε, το ίδιο το ζητά και η πολιτική μα ομάδα στην κυβέρνηση τη Πενέζα, να χρησιμοποιήσει τι συνταγματικέ δυνατότητε που έχει για να σταματήσει το κλείσιμο των εργοστασίων τη Κορούνια και του, και του για να εγγυηθεί πως θα συνεχιστεί η απασχόληση, ότι αυτές, αυτά τα εργοστάσια θα συνεχίσουν να λειτουργούν και για να αποφευχθεί το δράμα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο κύριος Τόκες. Ευχαριστώ. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Γιούγκερ είχε εκφράσει σοβαρές αμφιβολίες για το αν η Ρουμανία έχει τη δυνατότητα να αναλάβει τα καθήκοντα της Προεδρίας. Και μάλιστα η χώρα μου καταδικάστηκε και από ψήφισμα του Κοινοβουλίου, του, η χώρα αυτή καταδικάστηκε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρ' όλα αυτά οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της η Ρουμανία ως Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε, την περιέγραψαν με τα πιο ζεστά χρώματα. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες θα επισκεφθούν το Βουκουρέστι και αυτό σημαίνει ότι είτε τους αρέσει είτε τους, ε, δεν τους αρέσει στην ουσία νομιμοποιούν το διεφθαρμένο μετακομμουνιστικό καθεστώς της Ρουμανίας που μάλιστα παραβιάζει τα δικαιώματα εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων. Θέλω να υπενθυμίσω το ψήφισμα της Άλμπα Ιούλια του 2017 όπου αναφερόταν ότι βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και θρησκευτικές ελευθερίες ε, παραβιάζονται στην ε, Ρουμανία. Δυστυχώς έκλεισε το μικρόφωνο του ομιλητή. Η κυρία Ζωάνα. Σας ευχαριστώ πολύ Ανησυχούμε πάρα πολύ για την απόφαση του Αυστριακού Κοινοβουλίου που επηρεάζει πάρα πολλού ε, ε, πολίτες της Ρουμανίας που ζουν στη χώρα αυτή και θεωρούμε ότι παραβιάζει τις αρχές των μη διακρίσεων. Κυρία Επίτροπε, πάνω από 130.000 ε, παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζονται από αυτή την απόφαση. Η Αυστρία παραβιάζει τις, τους, ε, την χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ε, καθιστά τα παιδιά των Ρουμάνων ως παιδιά δεύτερης κατηγορίας. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν μπορούν να λαμβάνονται οι ε, μέτρα εναντίον ε, Ευρωπαίων εργαζομένων Ρουμάνων που εργάζονται στην Αυστρία και να τους δίνονται λιγότερες παροχές από αυτές που δίνονται στους αντίστοιχους Αυστριακούς συναδέλφους τους. Αυτό σημαίνει ότι ε, θα παραβιαστούν, θα δοθούν 100 εκατομμύρια λιγότερα από ό,τι δίνονται για επιδόματα παιδιού από ό,τι δίνονται στους ε, αυστριακούς ε, εργαζόμενους. Πρέπει να αναλάβουμε άμεσες δράσεις για να επιβληθούν κυρώσεις εναντίον αυτής της παραβίασης των ευρωπαϊκών αρχών. Η κυρία Λόπες Μπερμέχου. Ευχαριστώ πολύ. Για μια φορά ακόμα έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες επιδοτούνται και παρόλα αυτά κρίνουν ε, τα εργοστάσια τους όταν αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία. Όπως η Αλκόα για παράδειγμα, πάνω από 700 εργαζόμενοι, η Βονταφών, 1200 θέσεις ε, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό απόλυση. Εντέσα, κλείσιμο του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς καμία πρόληψη για το προσωπικό. Τα επιχειρηματικά του σχέδια τους αφορούν πολύ περισσότερο από το προσωπικό τους. Η κυβέρνηση της Ισπανίας θα πρέπει να βρει κάποιες λύσεις με ένα παραγωγικό μοντέλο όπου το ΑΕΠ θα αυξηθεί και θα έχουμε περισσότερο προϋπολογισμό για τους εργαζομένους με δημόσιες επιχειρήσεις σε στρατηγικούς κλάδους οικονομίας και με μεταρρυθμίσεις ε, στην αγορά εργασίας. Από την αρχή της κρίσης οι εργαζόμενοι έχουν υποφέρει από τις λανθασμένες πολιτικές. Δεν είναι αυτός ο σωστός δρόμος. Ξεκινήστε με καλύτερα οικονομικά και κοινωνικά μέτρα όπου θα λάβετε υπόψη σοβαρά τα θέματα που αφορούν τους εργαζομένους.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 ε, ε, του έτους θα πρέπει να αποφασίσει αν ε, η Ρουμανία και η Βουλγαρία μπορούν να προσχωρήσουν στο χώρο Σέγγεν και ήδη κάποιες χώρες 12 χρόνια μετά από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα έχουν ε, λέει αμφιβολίε. Αυτό είναι εξοργιστικό. Θα πρέπει, εμείς έχουμε κάνει τα απαραίτητα βήματα, είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα ε, του, του χώρου Σέγγεν σε αντίθεση με χώρες που είναι ήδη μέλη του Σέγγεν. Ε, εμποδίζοντας τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία να προσχωρήσουν στο χώρο Σέγγεν, ε, ε, οι υπόλοιπες χώρες δίνουν ένα αρνητικό μήνυμα. Θεωρούν τους Ρουμάνους και τους Βούλγαρους δεύτερης κατηγορίας πολίτες που δεν αξίζουν ε, η συμμεταχείριση. Θα ήταν δίκαιο οι χώρες αυτές και οι κυβερνήσεις τους να αναλάβουν την ευθύνη για τις αποφάσεις αυτές και να τις αιτιολογήσουν. Ο κύριος Παπά. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε λοιπόν πως πολύ πρόσφατα εγκρίναμε την νομοθεσία ε, ε, για τα επιδόματα παιδιών ε, για μη κατοίκους. Μέχρι τώρα για όσους εργάζονται εκτός Ρουμανίας και έχουν τα, την οικογένειά τους στη Ρουμανία, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Γιατί, για παράδειγμα, ε, ε, οι Ρουμάνοι που εργάζονται στην Αυστρία πληρώνουν αυστριακούς φόρους, αλλά λαμβάνουν επιδοτήσεις, ε, επιδόματα τέκνου σε επίπεδα ρουμανικά. Αυτό καταστρατηγεί μια βασική πολιτική και κοινωνική αρχή που είναι τα ίδια επιδόματα όταν καταβάλει κανείς τους ίδιους φόρους. Η Αυστρία δεν έχει αυτό το δικαίωμα με αποτέλεσμα να έχει λιγότερη συνοχή το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τα μέτρα το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε οι, Ευρω... Ρουμάνοι πολίτες που εργάζονται στην Αυστρία να μην αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους ε, διακρίσει. Κυρία Πρόεδρε, τις προηγούμενες εβδομάδες βλέπουμε να υπάρχουν προσπάθειες να εκφοβιστούν μέλη του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Η, Μετρο... η Μητροπολιτική Αστυνομία μάλιστα συνέλαβε έναν ε, διαφωνούντα με το Brexit. Και αυτό συνδέεται με ακροδεξιές οργανώσεις οι οποίες ε, πολλές φορές ε, έχουν στους κόλπους τους και εγκληματίες. Ο Τζέραλτ Μπάτλερ, ηγέτης του UKIP, μάλιστα είχε τέτοιους ανθρώπους και ο συμβούλους του. Πρόκειται για ανησυχητικέ εξελίξεις σε πολύ επικίνδυνες περιοχές. Να μην ε, ξεχάσουμε ότι την ε, βουλευτή των εργατικών, Τζο Κόξ, που ε, δολοφονήθηκε τον ε, Ιούνιο του 2016 από έναν ακροδεξιό που ούρλιαζε πρώτα η Βρετανία. Πρέπει λοιπόν να καλέσω ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην κάνει, ανεκτές, ε, να μην κάνει ανεκτά τέτοια φαινόμενα και να κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να προστατευτεί η δημοκρατία. Η κυρία Απεργία πείνα. Αυτό είναι μια απόφαση που δεν παίρνει κανεί εύκολα. Παρ' όλα αυτά, χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο αυτό το απελπισμένο μέλος, ε, μέτρο ω ηθική ε, επιλογή. Πήγα στο Διαρμπακύρ όπου η Λέλα Γκούβεν, η πολιτικός του DHP, είναι σε κρίσιμη κατάσταση γιατί έχει 67 μέρες που είναι σε απεργία πείνα κατά τη απάνθρωπη πολιτική που επιβάλλουν στον ε, ο Τσαλάν στο Ιμραλί η Τούρκοι. Είναι ήδη ένα χρόνο φυλακισμένη, περιμένει να δικαστεί. Γιατί, γιατί ε, καταδίκασε, μάλλον άσκησε κριτική ε, στην επίθεση